Αγαπητοί συνάδελφοι, χτες ε, ορτάσαμε την ε, Διεθνή ημέρα νοσοκόμων ε, και ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας έχει κηρύξει το έτος 2020 έτος νοσοκόμων και με ευθύρων. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω με ευχαριστίες ε, προς τους άνδρες ε, και γυναίκες με τις άσπρες ε, ποδιές που παρέχουν τις απαραίτητες υγειονομικές υπηρεσίες με ανθρωπισμό και αυταπάρνηση. Και θα πρέπει βεβαίως να προσπαθήσουμε και εμείς να λειτουργήσουμε με αποτελεσματικότητα και ασφάλεια. Βεβαίως θα ήθελα να ευχαριστήσω και του εργαζόμενους στα νοσοκομεία και την πολιτική άμυνα, πολιτική προστασία. Και βεβαίως όλη αυτή η αλληλεγγύη αποτελεί έναν πλούτο για τις ε, χώρες μας. Φαίνεται λοιπόν ότι τώρα είναι ανάγκη να αυξηθούν οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της υγείας. Είναι κάτι το οποίο οφείλουμε στους πολίτες μας. ακριβώς για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε με έναν τρόπο κοινό σε οποιαδήποτε υγειονομική κρίση. Η πανδημία του COVID-19 κατέδειξε την αναγκαιότητα μιας πολιτικής δημόσιας υγείας η οποία θα έχει μεγαλύτερο ρόλο για την πρόληψη και την καλύτερη συνεργασία για να φτιάξουμε στήματα βοήθειας ε, και παροχής υγειονομικών υπηρεσιών με αντοχή που θα επιδεικνύουν και μεγαλύτερη αλληλεγγύη στην Ευρώπη. Πριν από 70 χρόνια η αλληλεγγύη μεταξύ έξι ευρωπαϊκών χωρών προσπάθησε να δημιουργήσει μια Ευρώπη ειρήνης και ασφάλειας. Αυτό το οποίο δηλαδή είχε οραματιστεί ο Ρόμπερτ Σουμάν. Και έχουμε πλέον επιτεύγματα συγκεκριμένα που αποδεικνύουν μια αλληλεγγύη στην πράξη η οποία βελτιώνει και τη ζωή των ανθρώπων. Ήταν ένα όραμα φιλόδοξο αλλά και πάρα πολύ ρεαλιστικό το οποίο βασιζόταν στην φρίκη του πολέμου και στις θυσίες που έγιναν για να τελειώσει αυτή 75 χρόνια σε ένα κοινό οικοδόμημα με τόσες πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η δουλειά αυτή. Ειδικά στην αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Όπως όμως απέδειξαν άντρες, γυναίκες και νέοι, είμαστε σε θέση να επιδείξουμε αλληλεγγύη. Και έτσι θα γίνει και η δουλειά αυτή πιο εύκολη. Έχουμε λοιπόν μια μεγάλη ευθύνη μπροστά μας, πρέπει να αρθούμε στο ύψος των προσδοκιών των Ευρωπαίων πολιτών και να προσπαθήσουμε ακριβώς να αναστοχαστούμε το μέλλον της Ευρώπης για να δούμε ποιες θα είναι οι απαντήσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Η κρίση αυτή μας διδάσκει πάρα πολλά πράγματα αλλά κυρίως ότι μόνο μαζί μπορούμε να επανεκκινήσουμε. Σας ευχαριστώ. Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση η οποία είχε διακοπεί στις 17 ε, Απριλίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας υπενθυμίσω ότι έχουν ληφθεί μια σειρά προληπτικών μέτρων για να σεβαστούμε... Με συγχωρείτε, μία στιγμή. Allora Ας περιμένουμε μια στιγμή λοιπόν. Λειτουργεί τώρα. Ωραία. Πρώτα απ' όλα λοιπόν θα ήθελα να σας πενθυμίσω μια σειρά προληπτικών μέτρων τα οποία έχουν ληφθεί για να σεβαστούμε την τήρηση των αποστάσεων. Οι βουλευτέ που βρίσκονται στον κατάλογο των ομιλητών παρακαλούνται να καταλάβουν τι θέσει του στο ημικύκλιο, στο καρτελάκι που αναγράφει το όνομά σας. Οι βουλευτέ που δεν βρίσκονται στον κατάλογο των ομιλητών παρακαλούνται να ακολουθήσουν ε, τους ε, κλητήρε προ τι θέσει που θα του υποδείξουν. Όσοι δεν μπορέσουν να χωρέσουν στο ημικύκλιο, παρακαλούνται να χρησιμοποιήσουν την αίθουσα στο κτίριο SPAC 3 σε 50 η οποία έχει συνδεθεί αποτελεσματικά για αυτόν τον σκοπό. Σας ενημερώνω πως ε, το βιβλίο των παρουσιών βρίσκεται μπροστά και στις δύο αυτές αίθουσες. Οπότε, για να λειτουργήσουμε αποτελεσματικά, είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε όλους τους χώρους του κτηρίου, άρα και στην αίθουσα της Ολομέλειας και στην αίθουσα 3 50 οι ομιλητές που θέλουν να παρέμβουν στην συζήτηση χωρίς την μάσκα θα μπορούν να το κάνουν μόνο για την διάρκεια της παρέμβασής τους. Τα πρακτικά της συνεδρίας 16 και 17 Απριλίου σας έχουν μοιραστεί. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, οπότε τα πρακτικά εγκρίνονται. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα διαδικαστικό βάσει το άρθρο 22. Ε, θα πρέπει να εξασφαλίσετε ότι ε, ακολουθούνται οι κανονισμοί του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και βάσει το άρθρο 167 όλοι οι ευρωβουλευτέ έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τη μητρική του γλώσσα, μια και είναι επίσημη γλώσσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχουν όμω κάποιοι ευρωβουλευτέ που ε, ξερούνται από το δικαίωμα συμμετοχή συμμετοχή στη συζήτηση, γιατί δεν μπορούν να ε, ακούσουν, να καταλάβουν αυτά που συμβαίνουν ε, και αυτά που ακούν, γιατί δεν έχουν τη μητρική του γλώσσα στη διερμηνία. Έχουν πέρασει δύο μήνες από την έναρξη της κρίσης. Θα σας παρακαλούσα λοιπόν να με ρημνήσετε ώστε όλοι οι εκλεγμένοι ευρωβουλευτές να μπορούν να συμμετέχουν στη συζήτηση και να έχουν διερμηνία. Κοιτάξτε αγαπητέ, ε, υπάρχει διερμηνία. Τι είστε ζήτημα. Κύριε Βάιτς. Υπάρχει διασφάλιση της ερμηνείας, δεν αντιλαμβάνομαι τι θέλετε να πείτε, σε όλες τις επίσημες συνεδριάσεις του Κοινοβουλίου. Ο κύριος Μπόνις Ρόπε, συνάδελφος Ευρωβουλευτής, που μόνο λιθωνικά γνωρίζει και δεν αντιλαμβάνεται άλλη γλώσσα, δεν μιλάει άλλη γλώσσα, δεν μπορεί να μιλήσει σε άλλη γλώσσα από αυτές που προβλέπονται. Αυτό είναι ένα από τα πολλά παραδείγματα. Κοιτάξτε, θα ενημερωθώ, αλλά νομίζω ότι υπάρχει διασφάλιση διερμηνία σε όλες τις γλώσσες. Θα επιληφθώ πάντως του θέματος που αναφέρατε. Διαδικαστικό από τον ε, κύριο Μόιτεν. Έχετε τον λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αναγνωρίζοντας ε, την ιδιαίτερη κατάσταση, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να παραμερίσουμε την δημοκρατία. Αυτό ακριβώς συμβαίνει όμως εδώ πέρα. Έχετε απορρίψει απλά τις τροπολογίες μας χωρίς κάποια δικαιολογία, αλλά δεν είναι δυνατόν να μειώνεται ο χρόνος ομιλίας ε, και οι τροπολογίες στις περισσότερες επιτροπές να υποβάλλονται μόνο στα αγγλικά και να μην επιτρέπονται σε μονομένους βουλευτές αλλά μόνο σε κοινοβουλευτικές ομάδες. Και μάλιστα θα πρέπει να είναι παρόντες οι βουλευτές μία ώρα πριν ε, από την ε, έναρξη της συνεδρίας, κάτι το οποίο υπονομεύει την ελευθερία της εντολής. Δεν ανταποκρινόμαστε πλέον σε κάποιες δημοκρατικές προδιαγραφές. Θα πρέπει να επανέλθουμε κατεπηγόντως στην κοινοβουλευτική και δημοκρατική κανονικότητα από την οποία πόρο απέχουμε αυτή τη στιγμή. Αλλιώς δεν μπορούμε να πούμε ότι πρόωθουμε δημοκρατία. Αντιθέτως φαίνεται ότι χρησιμοποιείται αυτή η κρίση για να υπάρξει ένας περιορισμός δημοκρατίας. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε σύνεπείς. Σας ευχαριστώ για τις ε, παρατηρήσεις σας κύριε Μόιτεν. Υπενθυμίζω ότι είμαστε ένα από τα λίγα κοινοβούλια τα οποία ε, διατήρησαν ε, την ε, κανονικότητα και συνέχισαν να λειτουργούν. Οπότε η κριτική η οποία ασκείται δεν είναι αποδεκτή. Γι' αυτό το οποίο είπατε τώρα συγκεκριμένα για τις τροπολογίες. Οι τροπολογίες έγιναν δεκτές σύμφωνα με τον κανονισμό. Βεβαίως, είναι μια στιγμή ιδιαιτέρως δύσκολη και όλοι πρέπει να επιδείξουν κατανόηση, γιατί ακόμα δεν έχει τελειώσει η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης εξακολουθεί να υφίσταται και πρέπει βεβαίως να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την υγεία. Και θεωρώ ότι αυτό το κοινοβούλιο κινήθηκε ταχαίως ε, για να τα διασφαλίσει αυτά. Σας ευχαριστώ για τις ε, παρατηρήσεις σας. Λοιπόν, επευκαιρία της ε, τελευταίας συνεδρίας της διάσκεψης των Προέδρων στις 7 Μαΐου αποφασίσαμε με τους επικεφαλεί των πολιτικών ομάδων να παρατείνουμε την Ολομέλεια μέχρι την Παρασκευή 15 Μαΐου. Παρά την πανδημία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεχίζει να εκτελεί τις θεμελιώδεις λειτουργίες του. Με την παράταση αυτή, μα ποιο μιλάει μεγαλόφωνα μέσα στην αίθουσα. Παρά την πανδημία λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεχίζει να ασκεί τις εμελιώδεις λειτουργίες του. Με την παράταση αυτή έχουμε βρει ένα σύστημα το οποίο επαρκεί για την εξαποστάσεως ψηφοφορία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεχίζει να ασκεί πλήρως τον ρόλο του και να εκτελεί τα καθήκοντά του, συγκεκριμένα δηλαδή ψηφοφορίες για συγκεκριμένα θέματα, κατεπήγοντα όπως αυτά που αφορούν την πανδημία του COVID-19 και θα είμαστε έτοιμοι επίσης ε, για να προχωρήσουμε τη ψηφοφορία και του νέου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ έστειλε ένα διορθωτικό κείμενο σύμφωνα με το άρθρο 241 παράγραφος ε, Τέσσερα του κανονισμού η διορθωσία αυτή εγκρίνεται εκτός εάν εντός 24 ωρών αριθμός βουλευτών ή ε, μια πολιτική ομάδα εκδηλώσει την διαφωνία της. Η διορθωσία υπάρχει στο site του Κοινοβουλίου και θα δημοσιευτεί προσεχώς. Οι επιτροπές Άγκρη και ΠΕΣ αποφάσισαν να ξεκινήσουν διοργανικές διαπραγματεύσει σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 1 του κανονισμού. Οι εντολέ για τι διαπραγματεύσει αυτές είναι διαθέσιμε στην ιστοσελίδα της Ολομέλειας και οι τίτλοι τους θα δημοσιευτούν με τα πρακτικά αυτή τη συνεδρίασης. Σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 2, ε, ένα αριθμό βουλευτών ε, ή περισσότερες ε, πολιτικές ομάδες μπορούν να ζητήσουν μέχρι τις 14 ε, ε, Μαΐου να τεθεί σε ψηφοφορία η απόφαση αυτή. Αν δεν γίνει αυτό, θα μπορέσουν να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Θα ήθελα να ενημερώσω την αίθουσα Πώς μετά την διακοπή στις 17 Απριλίου και σύμφωνα με το άρθρο 79 του κανονισμού υπέγραψα μαζί με τον πρόεδρο του Συμβουλίου τέσσερις νομοθετικές ε, πράξεις που έγιναν σύμφωνα με την τακτική νομοθετική διαδικασία. Οι τίτλοι τους θα δημοσιευτούν στα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης. Περνάμε τώρα στην διάταξη των εργασιών. όπως αυτή εγκρίθηκε στις 5 ε, Μαΐου σύμφωνα με το άρθρο 175 σας έχει διανεμηθεί. Θα δούμε τώρα κάποιες ε, τροποποιήσεις. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ενημερώσω πως έχω λάβει κάποια αιτήματα τα οποία αφορούν την προσθήκη των εξή νομοθετικών εγγράφων που σχετίζονται με την ε, επιδημία του COVID-19 στην Ολομέλεια αυτή της 13ης μέχρι 16ης Μαρτίου. Πρώτα απ' όλα, μακροοικονομική βοήθεια στις ε, χώρες της γειτονίας οι οποίες πλήττονται από τον COVID-19. Δεύτερον, προσωρινά μέτρα όσον αφορά την ε, Γενική Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Εταιριών και Ευρωπαϊκών Συνεταιριστικών Εταιριών. Τρίτον, μέτρα για τις λιμενικές υποδομές. Τέταρτον, μέτρα τα οποία αφορούν την ισχύ συγκεκριμένων αδειών και διπλωμάτων, όμνιμπους, ε, πέμπτο, παροχή αεροπορικών υπηρεσιών, έκτο, τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο, παράταση της ε, περίοδου ισχύω. Θα ήθελα λοιπόν ε, να υποβάλλω στην αίθουσα προς έγκριση τις αλλαγές αυτές της ημερήσιας διάταξη; Όσον αφορά λοιπόν την Τετάρτη, πρώτα απ' όλα η ψηφοφορία για τα ανώτατα επίπεδα σύγκλωση DIM. Το σημείο αυτό έχει αποσυρθεί και θα το παρουσιάσει η νέου Κομισιόν τον Ιούλιο. Όσον αφορά την ψηφοφορία, τον πρώτο γύρο ψηφοφορίας, αυτός θα ξεκινήσει 15 και 30 μέχρι τις 16 και 45 και θα ψηφίσουμε πρώτα απ' όλα τέσσερα έγγραφα τραν ίντα με τη διαδικασία κοντεπήγοντος τραν, τραν ίντα και γιούρι δεύτερον 8 ψηφοφορίες όπως προβλέπει αυτή τη στιγμή το σχέδιο ημερήσιας διάταξης τρίτον δύο εκθέσεις ε, του κυρίου Φέρμπερ μια έκθεση των κύριων Όλμπραϊτ και Μαρκές και μια έκθεση του κύριου Λόπες Αγγιλάρ. Τέταρτον, ψηφοφορία σε τμήματα για την γενετικά τροποιημένη σόγια. Και τελευταίο, όλες οι αποφάσεις της απαλλαγής. Ο πρώτος γύρος ε, λοιπόν θα γίνει 15 και 30, ο δεύτερος 8 με 9 και τέταρτο και η τελική ψηφοφορία για τις αντιρρήσεις για την γενετικά τροποποιημένη σόγια. Όσον αφορά τις ε, συζητήσεις. Είχαμε μία η οποία αφορά το έκτακτο συμβούλιο της 23ης Απριλίου και μία για το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο ήδη υπό όρη. Αυτά θα γίνουν μία κοινή συζήτηση. Η συζήτηση θα διεξαχθεί σήμερα από τις 4 μέχρι τις 7 το απόγευμα η ανακοίνωση της Κομισιόν ε, για την ε, νομοθεσία στην Ουγγαρία αναβάλλεται για την 5η από τις 9 μέχρι τις 10. Όσον αφορά την αυριανή ημέρα, 5η, η συνεδρία θα επαναληφθεί 9 η ώρα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας Τετάρτης. Ο πρώτος γύρος ψηφοφορίας θα ξεκινήσει 9.30 η ώρα και θα ψηφίσουμε το δεύτερο μπλοκ τροπολογιών το οποίο θα αφορά τα ψηφίσματα της απαλλαγής. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου γύρου της ψηφοφορίας θα λάβει η χώρα στις 13 και 15. Δεύτερος γύρος ψηφοφορίας θα γίνει 13 και 30 με τελική ψηφοφορία επί όλων των ψηφισμάτων περί απαλλαγής, επί των τροπολογιών του έκθεση του κυρίου Σαστέλ, ψηφοφορία για το έγγραφο Γιούρι με τη διαδικασία του κατεπήγοντο για τα προσωρινά μέτρα για τι γενικέ συνελεύσει των ευρωπαϊκών εταιριών. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στον δεύτερο γύρο θα λάβει χώρα 17 και 15. Τρίτος γύρος φοφορίας θα ξεκινήσει 17 και 30 μέχρι τις 18.45 με ψηφοφορία στο πρώτο μπλοκ τροπολογιών για το κοινό ψήφισμα για το νέο πι δελτα πι ήδη πόρη και τελική έκθεση του κυρίου Σαστέρ. Όσον αφορά την Παρασκευή, η διαδικασία θα επαναληφθεί στις 9 και 4 με ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της φοφορίας προηγούμενης μέρας. Πρώτος γύρος φοφορίας 9.30 μέχρι 10 και 45 και θα ψηφιστούν τα ε, οι εκθέσεις ε, των Επιτροπών είναι τα με τη δικασία του κατεπίγοντο και πιθανώ το δεύτερο μπλοκ τροπολογιών με την πρόταση ψηφίσματο για το νέο πι δελτα και ίδιους πόρους και το σχέδιο ανάκαμψης. Ε, θα έχουμε λοιπόν δεύτερο γύρο 15 η ώρα και με ψηφοφορίες οι οποίες θα αφορούν τα τελικά την τελική έκθεση για το ΠΔΠ ίδιους πόρου και το σχέδιο ανάκαμψη ε, και τα έγγραφα με τη διαδικασία του κατεπήγοντο Ίντα και Τράνη. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του δεύτερου γύρου ψηφοφορίας θα γίνει στις 17 και 30. Τρίτο γύρο ψηφοφορία επί των ε, θεμάτων αυτών του ψηφίσματος για το νέο ΠΔΠ θα μπορούσε πιθανώς ε, να λάβει χώρα 16.45 με 19 η ώρα. Όσον αφορά το Σάββατο, δεν προβλέπεται κάποια συνεδρίαση, εκτός αν υπάρξουν κάποιες αντιρρήσεις, οπότε αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις εγκρίνονται οι αλλαγές αυτές. Παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ. Είμαι κατά της διαδικασίας του κατεπήγοντος ε, για τις ε, αεροπορικές υπηρεσίες εκ μέρους της ΓΚΟΕ. Φυσικά θα θέλαμε να συμφωνήσουμε στη... Ε, συμφωνήσαμε στη διαδικασία αυτή την περασμένη φορά για τις ε, πτήσεις φαντάσματα που είχαν άμεσο αντίκτυπο, αλλά να και πάλι πρόταση για χαλάρωση πολύ σημαντικών κανονισμών ε, για τις αερομεταφορές χωρίς κανένα απολύτως κοινοβουλευτικό προηγούμενο έλεγχο. Θεωρούμε ότι αυτή η διαδικασία είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, γιατί στην ουσία επιτρέπουμε σημαντική χαλάρωση στην εφαρμογή των κανονισμών ε, μέχρι το 2023 για τις υπηρεσίες εδάφους χωρίς καμία συζήτηση ή συνεισφορά της Επιτροπής Μεταφορών ή συζήτηση στην Ολομέλεια. Δεν είναι κάτι τόσο κατεπίγον ώστε να μπορεί να περιμένει ένα μήνα ακόμη. Στο μεταξύ όμως ο κλάδος που υποφελείται από τα μέτρα αυτά έχει ήδη αναγγείλει χιλιάδες απολύσεις εργαζομένων και κατάφορα παραβιάζει τα δικαιώματα των επιβατών ε, για επιστροφή των χρημάτων για τις που έχουν ακυρωθεί. Θα πρέπει λοιπόν ε, να επανέλθουμε στην προστασία των καταναλωτών και των δικαιωμάτων των επιβατών. Είμαστε κατά τη διαδικασία του κατεπήγοντο. Δεν, δεν μπορούμε να χύνουμε κροκοδίλια δάκρυα, για, ε, να δεχόμαστε να χύνουμε κροκοδίλια δάκρυα για αυτέ τι ανησυχίε και αντί να χρησιμοποιούμε την πίεση που έχουμε να ε, επιβάλλουμε κάποια μέτρα. αυτό Ναι, βεβαίω όλα αυτά θα ψηφιστούν. Υπάρχουν άλλοι που θέλουν να παρέμβουν. Βάσκες. Όχι. Πού είναι. Ε, no Συγγνώμη, δεν είχα ακούσει το όνομά μου. Πριν ξεκινήσω την παρέμβασή μου, θα ήθελα εκ μέρου τη Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων ε, ε, τι ευχαριστίε μου και την έκφραση αλληλεγγύη για όσου του τομεί καταπώνητα εργάστηκαν για να υπερβούμε αυτή την υγειονομική κρίση και τι δυνάμει ασφαλεία του κράτου που συνέβαλαν ε, στην μέρημνα για να είμαστε όλοι ασφαλεί και υγιεί. Η πανδημία COVID-19 σήμανε ένα πριν και ένα μετά και η απομόνωση στα σπίτια μας, ε, μακριά πολλές φορές από τους αγαπημένους μας, ε, η παράλυση σημαντικών οικονομικών δραστηριοτήτων και η απώλεια σημαντικών ε, θέσεων εργασίας ήταν αδιανόητα πριν την πανδημία αυτή. Και Φαίνεται τι τεράστιε προσπάθειες απαιτήσαμε από του ευρωπαίου πολίτε. Θα πρέπει λοιπόν να σταθούμε και εμεί στο ύψο των περιστάσεων και να ανταποκριθούμε στι ε, προσδοκίε των πολιτών. Οι ελεύθεροι επαγγελματίε και επιχειρήσει ε, δίνουν τον καλύτερό του σε αυτό για να ξεπεράσουν την κρίση και να μπορέσουν να συνεχίσουν τι εργασίε του μετά την κρίση. Για να είμαστε λοιπόν στο ύψο των περιστάσεων θα πρέπει να προστατεύσουμε τα, τα συμφέροντα των επιχειρήσεων και ε, έχουμε μια εξαιρετική ευκαιρία να το κάνουμε. Ε, γιατί οι ανώνυμες ευρωπαϊκές εταιρείες δεν μπορούν στους ε, πρώτους έξι μήνες να οργανώσουν τις ε, γενικές του συνελεύσεις λόγω των όρων της πανδημίας. Γι' αυτό και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπαγορεύεται από την κοινή λογική και τροποποιεί την νομοθεσία ώστε στη διάρκεια του 2020 να προβλεφθεί μία εξαίρεση για τον κανόνα αυτό για τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων και η προθεσμία για, την για τη διοργάνωσή τους παρατείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους. Επίσης χρησιμοποιούνται τα διάφορα ψηφιακά μέσα για να γίνουν τέτοιες γενικές συνελεύσεις. Είναι αναπόδραστη και απαραίτητη αυτή η μεταρρύθμιση και συνάδει με τη διαδικασία του κατεπήγοντος και θέλω, θα ήθελα να εγκριθούν. Δεν μπορούν να μην γνωρίζουν οι επιχειρήσει θα είναι υποχρεωμένε να οργανώσουν τον επόμενο μήνα τι γενικέ συνελεύσει με όλου του κινδύνου που συνεπιφέρει κάτι τέτοιο ή να μπορούν να τι αναβάλουν για το επόμενο εξάμεινο. Θα πρέπει να στείλουμε ένα απερίφραστο μήνυμα ότι είμαστε υπέρ τη προστασία των επιχειρήσεων αυτών. Γιατί παίζουμε την αξιοπιστία μα και το μέλλον μα σε κάθε κρίση. Ε, εξαρτηθεί από τη φροντίδα και τη μέρημνα που θα δείξουμε για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Και για αυτούς όλους τους λόγους σας ζητώ να υπερψηφίσετε αυτή τη διαδικασία του καταπέκοντος. Μάλιστα, ακούσαμε. Τι και κατά περνάμε λοιπόν στην ψηφοφορία 6 αιτήματα αλλαγή ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με το άρθρο 163 του κανονισμού στα έγγραφα τα οποία ήδη αναφέραμε όσον αφορά τις ε, δύο θέσεις ε, του Συμβουλίου όσον αφορά την ε, σήμανση των ελαστικών για την κατανάλωση καυσίμου και την θέση για την χρήση των υδάτων. Να σας μεθυμίσω εδώ πέρα το άρθρο 67 και 68 του κανονισμού. Οι υπόλοιπες προτάσεις θεωρούνται εγκεκριμένες. Πριν περάσουμε στην ψηφοφορία να σας πω πώς θα διεξαχθεί αυτή. Θα ήθελα λοιπόν εδώ πέρα να ευχαριστήσω την ε, διεργασία που έχει κάνει η Γενική Διεύθυνση της Προεδρίας η οποία έχει βελτιώσει το σύστημα ψηφοφορίας μια δουλειά η οποία είναι συνεχής και αποτελεσματική τις εβδομάδες αυτές Τα αποτελέσματα λοιπόν έχουν αποσταλεί σε όλους τους βουλευτές, έγιναν δύο δοκιμαστικές ψηφοφορίες έτσι ώστε όλοι να μπορέσουν να εξοικειωθούν με την διαδικασία. Ξεκινάει τώρα η ψηφοφορία 15 και 30 μέχρι 16 και 45 όλες οι σημερινές ψηφοφορίες θα είναι ονομαστικές οι βουλευτές μπορούν να επαληθεύσουν το τι ψήφισαν και τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών στο site ε, της ε, Ολομέλειας. Κάτ' εξαίρεση θα γίνουν ε, δεκτές δηλώσεις επεξήγησης ψήφου μέχρι 400 λέξεις maximum. Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών θα ανακοινωθούν στις 19 και 45. Οπότε Τώρα, ωραιότατα. Διακόπτεται η συνεδρίαση και επαναλαμβάνεται στις 16 και 00 με τα συμπεράσματα τη έκτακτη συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, νέο πιδελταπή, ήδη υπόρρη και σχέδιο ανάκαμψη. Σα ευχαριστώ. Ah,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 είναι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 Συνάδελφοι, η μερίσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση για τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για, τις, για τους ιδίους πόρους και το ε, πρόγραμμα ανάκαμψης. Θα ακούσουμε τις, δισο, τις δηλώσεις του Ευρωπαϊκού του Συμβουλίου και της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να θυμίσω στους συναδέλφους ότι η αυτή, η συζήτηση αυτή δεν περιλαμβάνει τη διαδικασία Κατστιάη ούτε τις γαλάζιες κάρτες. Να δώσω το λόγο ευθύ αμέσω στον πρόεδρο Σαρλ Μισελ και να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Έχετε το λόγο, πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, Αγαπητοί Ευρωβουλευτές, πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε και πάλι αυτή την ευκαιρία να λάβω εδώ το λόγο. Η κρίση αυτή είναι άνευ προηγουμένου. Σημαίνει ότι πρέπει και εμείς να λάβουμε αποφάσεις που θα είναι πρωτόγνωρες. Γι' αυτό είμαι πεπισμένος ότι η στενή συνεργασία μεταξύ των δημοκρατικών και νομιμοποιημένων ε, ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων θα είναι ύψη τη σημασία στου ερχόμενου μήνες. Είναι μια καλή ευκαιρία σήμερα εδώ να παρουσιάσω μερικά ε, στοιχεία μετά την τελευταία τηλεδιάσκεψη, την τελευταία σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Όπως θα γνωρίζετε, έχουμε ε, ήδη κάποιους συγκεκριμένους προσανατολισμούς. Ο πρώτος στόχος ήταν να στηρίξουμε τις προτάσεις που έγιναν από τους Υπουργούς Οικονομικών, προκειμένου να κινητοποιήσουμε πάνω από... 5 για να στηρίξουμε, 54 δις για να στηρίξουμε για να στηρίξουμε ε, τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους πολίτες και όλα αυτά μέχρι τον Ιούνιο. Εδώ βέβαια ξέρουμε ότι και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν αρκούν αυτά. Ξέρουμε ότι το Ευρωπαϊκό αυτό Συμβούλιο ήταν ευκαιρία για να περάσουμε από την διαχείριση της κρίσης ε, βραχυπρόθεσμα ε, σε κάτι μακροπρόθεσμο. Όχι μια κοντόφθαλμη θεώρηση, και να έχουμε συγκεκριμένους προσανατολισμούς για τη στρατηγική ε, ανάκαμψη και για τη στρατηγική μετατροπής του κοινωνικού μας και οικονομικού μας μοντέλου. Κυρίες και κύριοι, αυτή η τέταρτη διάσκεψη ήταν ε, η ευκαιρία για να συζητήσουμε το φύλλο πορείας που ε, θέλαμε να έχουμε μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλαμε δε, λοιπόν εδώ να παρουσιάσουμε τα τέσσερα κεφάλαια που κοιτάζουμε από κοινού και να επικεντρωθούμε κυρίω σε δύο πτυχέ. Δύο πτυχέ των αντικείμενων συζητήσεων και θα πρέπει να μα κινητοποιούν του ερχόμενου μήνε, τι ερχόμενε εβδομάδε. Πρώτο σημείο είναι η ανάγκη να είμαστε διαρκώ ε, σε επαγρύπνηση για την κατάσταση τη εσωτερική αγορά. Πώ μπορούμε δηλαδή να ενισχύσουμε την εσωτερική αγορά και αν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι δυσκολίε, οι προκλήσει που υπήρχαν πριν την πανδημία ε, δεν έχουν εξαλειφθεί φυσικά με την έλευση αυτής της πανδημίας. Η κλιματική, ε, η πράσινη ατζέντα Ξέρετε ότι και πριν από την, ε, το ξέσπασμα αυτή τη πανδημία είχαμε λάβει ιστορικέ αποφάσει, ιδίω στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και με την υποστήριξη του Ευρωκοινοβουλίου, γιατί θεωρούσαμε ότι η κλιματική ουδετερότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι ένα στόχο που να κινητοποιήσει όλου. Θα πρέπει να στηρίξουμε τι επιχειρήσει και τι εταιρείε μα και να επιτρέψουμε την οικονομική μα ε, μεταμόρφωση. Μέσα σε αυτή την ψηφιακή εποχή θα πρέπει λοιπόν να αναλάβουμε κάθε δυνατή δράση προ τη σωστή κατεύθυνση, ε, με την βεβαιότητα ότι το κλίμα θα πρέπει να είναι στο κέντρο τη νέα μα ατζέντα. Η εσωτερική αγορά ήταν επίση σημαντικό στοιχείο τη ε, στρατηγική αυτονομία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ βλέπουμε ότι οι απόψει ε, συμπίπτουν με αυτά που επιθυμεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να αντλήσουμε τα διδάγματα του παρελθόντο και να ενισχύσουμε τι δυνατότητε παραγωγή μα. Στα πλαίσια αυτή τη στρατηγική, και για να πω και αυτό που ανέφεραν ε, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πολύ, ότι εδώ θα πρέπει να ε, πάρουμε τα ενία της Ευρώπης στα χέρια μας ε, και αυτό ακριβώς έδειξε και η πανδημία, αυτή η ιστορική κρίση. Πέραν των δεσμεύσεών μας ε, για την εσωτερική αγορά, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύντομα να υποβάλει έκθεση για τον τρόπο που τα διάφορα ευρωπαϊκά οικοσυστήματα επλήγησαν και επηρεάστηκαν, και αυτό θα συνεχιστεί και τι προσεχεί εβδομάδε, ώστε να ξέρουμε ακριβώ τι έχει συμβεί και να έχουμε χρήσιμε πληροφορίε στα χέρια μα. Δεύτερο σημείο Δεύτερο σημείο είναι η χρηματοδότηση. Είναι ζωτική σημασία να αναπτύξουμε μια φιλόδοξη στρατηγική για να έχουμε περισσότερα μέσα βασιζόμενη σε δύο ισχυρά εργαλεία. Πρώτον, ο ευρωπαϊκός προπολογισμός και τις περασμένες εβδομάδες, τους περασμένους μήνες είχαμε επανειλημμένο συζητήσει για τον προσανατολισμό που θέλουμε να λάβει ο ερχόμενο Ευρωπαϊκό ε, προπολογισμό και περισσότερο από ποτέ θα πρέπει να λάβουμε αποφάσεις και να προσαρμόσουμε τη στρατηγική μας για να προσαρμοστούμε. Να προσαρμοστούμε στι ε, ανίποτε συνέπειες αυτής της κρίσης. Όμως δεν αρκεί ευρωπαϊκός προπολογισμό. Γι' αυτό δεσμευτήκαμε να συνεργαστούμε και να εκκινήσουμε ένα ταμείο ανάκαμψης για να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε περισσότερα κονδύλια, μεγαλύτερα ποσά, έχοντας εντοπίσει ποιε είναι οι προτεραιότητες που θα μας απασχολήσουν στο εγγύς μέλλον. Σε αυτό το πλαίσιο αυτών των δύο εργαλείων που θα πρέπει να κινητοποιηθούν, κάποιοι και εγώ είμαι μεταξύ αυτών, κάλεσαν να προβλεφθεί μια στατικική τύπου σχεδίου Marshall ε, Εγώ θα το έλεγα πρόγραμμα σχέδιο Ντεκάσπερη, ενό από του ε, ε, ιδρυτέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ιταλία, για να ε, κινητοποιηθούμε στα επίπεδα τη χρηματοδότηση. Αυτό πρέπει να συζητήσουμε. Πώ θα χρηματοδοτήσουμε, πώ θα προβλέψουμε το ύψο των ποσών που χρειάζονται και μετά πώ θα προβλέψουμε τη σχέση διάδραση μεταξύ του Ταμείου Αυτού Ανάκαμψη και του ερχόμενου πολιτή δημοσιονομικού πλαισίου, δηλαδή του ερχόμενου Ευρωπαϊκού Προπολογισμού. Πώ θα μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε τα μέσα που χρειάζονται για να πετύχει η οικονομική ανάκαμψη. Και επιπλέον στο περιθώριο αυτές της συζήτησης για την ανάκαμψη, για την ε, μετατροπή, θα πρέπει να συνεχιστεί και η συζήτηση των προτάσεων που ε, θα υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, λόγω αυτής της πανδημίας. Αυτά την ανάγκασαν βεβαίως όλα να προβλέψει νέες ιδέες και προτάσεις που θα συζητηθούν. Εδώ θέλω ας πούμε να Ε, στη σχολιάσω μερικά πράγματα γιατί μου δόθηκε ευκαιρία εδώ να συζητήσουμε τις πτυχές των νέων προτάσεων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βασικό χαρακτηριστικό του ευρωπαϊκού εγχειρήματος από την ε, ε, ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν η ειρήνη και η ευμερία. Αυτά ήταν τα βασικά στοιχεία. Όμως ήταν και η ιδέα ότι με την συνεργασία, με την κοινή μας δουλειά μπορούμε με μια, ένα πνεύμα αλληλεγγύης να αντιμετωπίσουμε τι κοινέ μας προκλήσεις. Και βεβαίως τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες ε, θέμα του ευρωπαϊκού εγχειρήματο ήταν και η σύγκληση, δηλαδή να πάυσουν οι ανισότητες, να πάυσουν οι βαθιές διαφορές αυτό το σημείο είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να συμφωνήσουν τα κράτη-μέλη. Δεν θα πρέπει αυτά λοιπόν να γίνουν δικαιολογία, πρόσχημα, αφορμή για να ε, οξυνθούν οι ανισότητες και οι διαφορές στο ευρωπαϊκό επίπεδο, για να οξυνθούν οι ε, λήψεις ισορροπίας. Θα πρέπει ε, απέναντίας να ενισχύσουμε την κοινή μας βούληση για να υπάρξει περισσότερη συνοχή, περισσότερη συνεργασία και περισσότερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ε, περισσότερο από ποτέ λοιπόν Συμμερίζομαι την άποψη ότι η κρίση αυτή αποκαλύπτει πόσο η λύση που θα πρέπει να βρούμε είναι περισσότερη συνεργασία, περισσότερη ε, ολοκλήρωση, περισσότερη ε, κοινή βούληση και όχι το αντίθετο. Διότι το αντίθετο θα σημαίνει περισσότερη αδυναμία και ε, περισσότερους διχασμούς, πράγμα που το βλέπουμε και σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί εκεί δημιουργούνται δυσκολίε όπου υπάρχουν σοβαροί τριγμοί. Και ένα άλλο σοβαρό σημείο διότι βλέπουμε ήδη τις πολύ σοβαρές συνέπειες στο οικονομικό επίπεδο, λόγου χάρη στον τουριστικό κλάδο ή στις ε, αεροπορικές εταιρείε. Σε πολλούς κλάδους βλέπουμε ότι τις ερχόμενες ημέρες, τις ερχόμενες εβδομάδες θα υπάρξει ανάγκη να εργαστούμε ε, σκληρά βάσει των προτάσεων που θα υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστάσεων που ακόμη και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ε, δουν τι θα κάνουν με τις αποφάσεις τους για τα σύνορα, για τον τουρισμό. Θα πρέπει γρήγορα λοιπόν να υποβληθούν προτάσεις και τα κράτη-μέλη γρήγορα να καθίσουν γύρω από το ίδιο τραπέζι, να ανασκουμποθούν ε, για να μπορέσουμε να ε, καταφέρουμε με τον ίδιο δυναμισμό να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση τη ανάκαμψη. Εγώ καλώ να ανοίξουν τα ευρωπαϊκά σύνορα, μόλι αυτό είναι δυνατό, λαμβάνοντα βέβαια τα μέτρα που απαιτούνται, ε, αλλά να υπάρξει η ελεύθερη κυκλοφορία των ε, πολιτών, κάτι που είναι άκρο σημαντικό. Και θα πρέπει σταδιακά να υπάρξει δυνατότητα να ξανανοίξουν τα σύνορα, κάτι που είναι καθοριστική σημασία και για το κοινωνικό ε, επίπεδο. Ελπίζω λοιπόν τι προσεχεί ημέρε να γίνει πραγματικά πρόοδο, ώστε να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να βρεθούν στο ίδιο τραπέζι και να λάβουν τι κατάλληλε αποφάσει με τρόπο συντονισμένο για να δείξουν πόσο ανθεκτική είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίε και κύριοι, εν τέλει, θα ήθελα να σα πω ακόμη και αν αυτό δεν ε, σχετίζεται ε, απευθεία με τα όσα συζητήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αλλά μου φαίνεται σημαντικό, εφόσον μιλώ στου Ευρωβουλευτέ ε, και το λέω με κάθε επισημότητα ω πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ότι θα υπερισχύσει το ευρωπαϊκό δίκαιο. Θα πριτανεύσει. Είναι ένα θέμα που θα σε μα αποσχολήσει και στο ερχόμενο διάστημα. Πρέπει να προχωρήσουν οι ευρωπαϊκέ ιδέε και τα ιδανικά και βεβαίω η ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Ο ρόλο τη ευρωπαϊκή δικαιοσύνη είναι σημαντική για να υπάρξει και ενιαία ερμηνεία του ευρωπαϊκού δικαίου. Ε, πριν από 70 χρόνια ο Ρόμπερτ Σούμαν ε, εκφώνησε μια δήλωση. Έκανε μια δήλωση που ακόμα και σήμερα είναι ένας από τους θεμέλιους, είναι ένας από τους θεμέλιους λίθους του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Ε, κάτι μάλιστα πολύ καινοτόμο. Ε, ενώ μόλις πριν λίγα χρόνια από τη στιγμή τη δήλωση, τα κράτη πολεμούσαν μεταξύ τους και οδηγήθηκαν σε εθνικές αναδιπλώσει που προκάλεσαν την τραγωδία που όλοι γνωρίζουμε. Ε, δεν θέλω να πω ότι αυτό που αντιμετωπίζουμε είναι πόλεμος, αλλά ο καθένα πρέπει να βρει τι δικέ του δυνάμει για να αντιμετωπίσει τις ε, προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην κάθε χώρα. Όμως τα κοινά σημεία που βρίσκω μεταξύ τη κατάστασης πριν από 70 χρόνια και τη σημερινή είναι ότι έχουμε να κάνουμε μια κρίση παγκόσμια, κρίση βαθιά, κρίση άνευ προηγουμένου. Ε, τότε είχαν χρειαστεί όλοι οι πόροι ε, δημιουργικότητα καινοτομία, ε, θάρρου και ανανέωση, ώστε να φύγει από την, το ο κόσμος και να κοιτάξει πώς θα ανασηκωθεί ε, το ίδιο και με την πολιτική μας γενιά σήμερα. Πρέπει να έχουμε την ίδια τόλμη, την ίδια ε, ε, δυνατότητα δημιουργικότητας και νέα συνεργασίας για να αντιμετωπίσουμε την δυστυχία, το, τις δυσχέρειες και την, την τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τόσε ευρωπαϊκέ οικογένειε, τόσοι ευρωπαίοι πολίτε. Θα πρέπει λοιπόν να δείξουμε ότι είμαστε πολιτικοί άνδρες και γυναίκε που είμαστε σε θέση να ε, σταθούμε στο ύψο της πρόκλησης αυτής, να βελτιώσουμε την κατάσταση της Ευρώπης και να προστατεύσουμε την αξιοπρεπία των πολιτών με ε, κοινωνίες οι οποίες να είναι καλοπροαίρετες στις πολιτικέ που χαράσουν και να, να το μέλλον με... Ευχαριστούμε Πρόεδρε Μισελ, ο Πρόεδρος και τον δώσουμε τον λόγο στην Πρόεδρο της ε, επιτροπή, την κυρία Φοντερ Έχετε το λόγο κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ Σαλ Μισελ, κυρίες και κύριοι, βουλευτές. 70 χρόνια πέρασαν από την ε, διακήρυξη Σούμαν. Κρίσεις, προκλήσεις, αυτά είναι γνωστά στην Ευρώπη. Ακριβώς όπως ορθά είπατε και από πολλές πλευρές πάντοτε η Ευρώπη δεν ήταν μόνο ενωμένοι στη διαφορετικότητα, αλλά ήταν και ενωμένοι μπροστά σε αυτέ τι αντικσότητε και σε αυτήν την περίοδο αντικσότητων δίνουμε κάποιε απαντήσει στι κρίσει. Και η Ευρώπη τώρα περισσότερο από ποτέ χρειάζεται αυτή την αποφασιστικότητα, την ε, ενότητα αλλά και την φιλοδοξία. Οπότε ε, με αυτό το πνεύμα τώρα πασχίζουμε σε σχέση με αυτό το φιλόδοξο σχέδιο Ανάκαμψη, όπω τα είπατε και σήμερα στο κείμενό σα, στο ψήφισμά σας κυρίε και κύριοι. Γνωρίζουμε όλοι γιατί χρειάζεται να αναλάβουμε δράση. Και τις τελευταίες αυτές εβδομάδες με ακούσατε συχνά να ομιλώ για το τι πρέπει να πράξει η Ευρώπη. Σήμερα δε θα σας μιλήσω για το πώς. Και θα σας παρουσιάσω την αρχιτεκτονική, και τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού του φιλόδοξου σχεδίου ανάκαμψη για την Ευρώπη ε, το οποίο επεξεργαζόμαστε αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει πρώτα πρώτα να κατανοήσουμε την ανατομία της ε, ιδιαίτερης αυτής κρίσης και επιτρέψτε μου να σας υποβάλω τρεις παρατηρήσεις πριν προβώ στην ε, ανάλυση. Περάσαμε από υφέσεις οικονομικές και στο παρελθόν, αλλά ουδέποτε είχαμε τέτοιου είδους ε, κλείσιμο της οικονομίας Σταμάτησε η οικονομία, φρέναρε, σταμάτησε ε, η αλυσία των προμηθειών, σταμάτησε η ζήτηση και η αλήθεια είναι ότι ε, ε, δεν θα μπορέσουμε σύντομα να ξαναγυρίσουμε στη συνήθεια ροή των πραγμάτων, στο business as usual. Ανοιγόμαστε σιγά σιγά και βλέπουμε ότι τι γίνεται με τα σχολεία. Ξέρουμε ότι οι περισσότεροι γονείς θα βουλεύουν από το σπίτι και έχουμε και τα μέτρα της απόστασης ασφαλείας. Ορθώς συνεχίζουν και ισχύουν, οπότε οι επιχειρήσεις θα πρέπει να τα σκεφτούν πώς θα λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις τους, ένα λόγες θα ανακάμψουμε, αλλά πρόκειται αυτό να πάρει χρόνο. Και η δεύτερη παρατηρήσή μου είναι η εξή ότι ο ιός είναι ίδιος σε κάθε χώρα. Όμως η δυνατότητα αντίδρασης και απορρόφησης των κραδασμών διαφέρει και ποικίλει. Όλοι γνωρίζουμε χώρες και περιφέρειες όπου η οικονομία ε, βασίζεται στον κλάδο του τουρισμού, του πολιτισμού, στις υπηρεσίες. Ε, αυτοί επλήγησαν πολύ περισσότερο και να μην ξεχνούμε ότι εκείνοι που χτυπήθηκαν πρώτοι από την επιδημία είναι αυτή που συνήθως είναι αυτή που χτυπήθηκαν περισσότερο γιατί είδαμε πόσο οδυνηρά είναι αυτά που γίνανε από την εμπειρία την Ισπανική, την Ιταλική ε, οπότε οι άλλοι μπόρεσαν έτσι να προστατευτούν, να προετοιμαστούν για το κύμα της επιδημίας κάθε κράτος μέλος στήριξε εργαζομένους και τις επιχειρήσεις όσο καλύτερα μπορούσε. Και επίσης, α, ε, ε, ακριβώς επειδή η Ευρώπη ε, ήταν αποφασιστική, ήταν γρήγορη, είχαμε την ε, ρήτρα διαφυγή στα ε, διευθυντικά ταμεία, είχαμε την ευελιξία όσον αφορά τις κρατικέ ενισχύσει. αλλά επίση ισχύει ότι κάθε κράτος μέλος έχει διαφορετική φορολογική πολιτική. Οπότε, και διαφορετική δημοσιονομική αρχιτεκτονική, οπότε είχαμε μεγάλη ποικιλία σε κάθε κράτο μέλο. Οπότε τώρα βλέπουμε ότι θα πρέπει να γίνει κάποιο είδου εξίσωση των όρων παιχνιδιού για την ενιαία αγορά. Οπότε έτσι θα πρέπει να αντιδράσει η Ευρώπη και πραγματικά να έχουμε μια πραγματική ανάκαμψη επί τη βάση των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαδραματίσει πλήρω τον ρόλο του και για μένα αυτό είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει το Κοινοβούλιο να έχει την δημοκρατική ε, λογοδοσία και θα πρέπει να ετοιμάσει αυτό το πακέτο της ανάκαμψης ακριβώς όπως ε, γίνεται και με τον προπολογισμό. Οπότε γι' αυτό σα λέω ότι πρέπει αυτό να συζητήσουμε σήμερα. Για να δούμε τώρα. Για να κάνουμε μια βουτιά σε αυτή τη δέσμη μέτρων τη ανάκαμψη. Δηλαδή ε, έχουμε τα εξή. Πρώτα-πρώτα έχουμε αυτό τον προπολογισμό, έχουμε αυτό το ε, το πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο και είπαμε ότι πρώτα πρώτα θα έχουμε κάποιο μέσο δημοσιονομικό για την ανάκαμψη και θα έχει πάρα πολύ μεγάλη ε, μεγάλη, μεγάλη ευελιξία να μπορεί να ε, δανειστεί από τις αγορές ε, η Κομισιόν στηριζόμενη από τα κρατη και επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε τι γίνεται όσον αφορά το σύνολο των πόρων αυτού του Ταμείου ε, του μέσου ανάκαμψη. και αυτό θα γίνει μέσω του ευρωπαϊκού προπολογισμού, δηλαδή μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και για αυτό είπα και σα επαναλαμβάνω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι θα έχει ε, λόγο στο πώς θα γίνουν οι δαπάνες όπω ακριβώς έχετε λόγο και για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Οπότε για να δούμε πού θα πάνε αυτά τα χρήματα. Αυτά τα χρήματα θα πάνε σε τρει πυλώνε. Ε, πρώτα πρώτα ε, έχουμε έναν πυλώνα που θα υποστηρίξει τα κράτη-μέλη ούτως ώστε να ανακάμψουν, ούτως ώστε να ξεπεράσουν αυτή την ε, κρίση. Και ο κύριος όγκος ενισχύσεων θα πάει σε αυτόν τον πρώτο πυλώνα ε, για να υπάρχει ένα νέο μέσο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Ε, αυτό όμως θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με την υπόλοιπη πολιτική μας. Έτσι νομίζω ότι θα μπορέσουμε να προλιάνουμε το έδαφος για να έχουμε μια Ευρώπη ανθεκτική και με ψηφιακή τεχνολογία αυτό θα γίνει με το ευρωπαϊκό εξάμενο. Και αυτό θα διατεθεί θα προσχεθεί σε όλα τα κράτη-μέλη, είτε ε, ανήκουν στην Ευρωζώνη είτε όχι. Και πρόκειται επίση να επικεντρωθούμε εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είχαμε τα πιο σημαντικά, τα πιο μεγάλα χτυπήματα. Ε, και αυτό είναι ε, ένα βασικό του πρώτου πυλώνα. Τα πάντα και τα περισσότερα χρήματα είπαμε, αλλά εκεί επίσης έχουμε και το θέμα του ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να συμπληρώσει ε, τα ταμεία συνοχής και αυτό θα είναι πέραν των ε, συγκεκριμένων πόρων που διατίθενται. Πρόκειται επομένω όλα αυτά να λαβούν κριτήριο το πόσο σοβαρή ήταν η κρίση. Δεύτερος πυλώνας τώρα. Ο δεύτερος πυλώνας έχει να κάνει με την επανεκκίνηση της οικονομίας και με την ε, βοήθεια προς τις ιδιωτικές επενδύσεις να κινηθούν και πάλι. Δεν πρέπει επομένω να προλάβουμε την κρίση. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις στους τομείς κλειδιά, στο 5G, ε, ε, καθαρά καύσιμα, ε, τεχνητή νοημοσύνη και αυτά τα ξέρουμε αλλά τώρα τι άλλαξε ότι τώρα η ανάγκη είναι πιο μεγάλη από ό,τι στο παρελθόν ε, και για αυτό το λόγο εμείς θέλουμε το Invest EU να αναβαθμιστεί και για πρώτη φορά θέλουμε να υπάρχει ένα μέσο διευκόλυνσης στρατηγικών επενδύσεων ούτω ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τις αλυσίδες αξίας τις πιο σημαντικές για ανθεκτικότητα κλπ. Τα είδαμε αυτά και στην ε, κρίση ε, πόσο, πόσο από την αλυσίδα προμήθειας επομένως θα πρέπει η Ευρώπη να μπορεί να παραγάγει τα πιο σημαντικά των φαρμάκων, αλλά επίσης χρειάζονται και κάποιες εταιρείες υγιείς, εύρωστες για να μπορέσουμε να κάνουμε τις επενδύσεις. Και αυτό επομένως θα καλυφθεί από τον δεύτερο αυτόν πυλώνα. Εκεί θα δούμε ένα νέο ε, όργανο του, του, να υπάρχει αξιόχρεος εταιρείε και έτσι να δούμε τι κίνδυνοι υπήρξαν λόγω του εγκλισμού, λόγω των περιοριστικών μέτρων μάλλον και στη συνέχεια έχουμε στον τρίτο και τελευταίο πυλώνα, ε, εκεί έχουμε το θέμα του πώ θα μπορέσουμε να αντιλήσουμε τα πρώτα συμπεράσματα από την κρίση, γιατί το τελευταίο μήνα καταλάβαμε ποιο είναι το πιο σημαντικό, τι πήγε καλά και τι πρέπει να βελτιωθεί. Οπότε και εμεί πρέπει να θωρακίσουμε κάποια προγράμματα, αυτά τα οποία βοηθάνε για την κρίση, το Rescue, ε, το Horizon Europe και επίσης ε, θα έχουμε ένα πρόγραμμα υγείας, ειδικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα εξασφαλίσουμε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε τους εταίρου μας με το που θα θωρακίσουμε αυτά τα μέσα πολιτικής γειτονίασης, διεθνή συνεργασία και κάποιο είδου προενταξιακή αρρωγή, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, με λίγα λόγια έτσι πρόκειται να είναι αυτό το σχεδίο ανάκαμψη. Πρόκειται να εστιάσουμε την προσοχή μα εκεί που το χρειάζονται περισσότερο, εκεί που θα πιάσει τόπο περισσότερο και πρόκειται για κάτι βράχη πρόθεσμο. Και επίση θα επικεντρωθούμε όσον αφορά τα πρώτα χρόνια τη ανάκαμψη. Πρόκειται να περιλάβει κάποιε χορηγήσει πόρων. Ε, θα έχουμε front loading ε, όσον αφορά ε, δηλαδή το πώ θα καλύψουμε τι επενδύσει από φέτο. Θα χρησιμοποιήσουμε κατά των μελών και δεν ξεκινούμε από το μηδέν, αυτό είναι σημαντικό, γιατί αυτό το μέσο ανάκαμψη πρόκειται να συμπληρώσει αυτά τα τρία δίκτυα ασφαλεία που αναφέρθηκαν και συμφώνησαν τον Απρίλιο οι ηγέτε. Το, το, το πρόγραμμα SOAR τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, ε, ό,τι προέρχεται από το Ταμείο Επενδύσεων και αυτή είναι, η απάντηση που απαιτεί και χρειάζεται η Ευρώπη και επίσης θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τους ίδιους πόρους, αυτούς που χρειάζεται ο προπολογισμό, ακριβώς ό,τι προτείναμε το 2018 ε, είναι μια απάντηση που λαμβάνει υπόψη τις κοινέ ε, αξίες και λαμβάνει υπόψη το κράτος δικαίου, είναι κάτι το οποίο το χρειαζόμαστε, είναι κάτι το οποίο είναι σχεδιασμένο για το μέλλον. Στα γερμανικά. Μία απάντηση που θα προκύψει από την κρίση, αλλά θα μας επιτρέψει να επενδύσουμε στο μέλλον. Και μιλάμε για αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών και των ανθρώπων, αλλά και αλληλεγγύη μεταξύ των διαφορετικών γενεών. Κυρίες και κύριοι, αργά ή γρήγορα οι οικονομολόγοι και οι επιστήμονες θα βρουν ένα εμβόλιο για τον κορονοϊό. Όμως για την κλιματική αλλαγή δεν υπάρχει εμβόλιο και θα πρέπει η Ευρώπη να επενδύσει σε ένα καθαρότερο μέλλον. Οι επενδύσεις μας για την ανάπτυξη, για την ανάκαμψη θα πρέπει να κοιτάξουν το θέμα του αυξανόμενου χρέους. Σε ό,τι αφορά και τα χρέη τα οποία θα χρειαστεί να πληρούν τα παιδιά μα στο μέλλον, το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να επενδύσουμε τα χρήματα αυτά σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση τη αλλαγή του κλίματο, σε ό,τι αφορά την μείωση τη επιβάρυνση του κλίματο για να μην υπάρξει επιπλέον επιβάρυνση. Και γι' αυτό σε ό,τι αφορά την κρίση και σε ό,τι αφορά την έξοδο από την κρίση, δεν μπορούμε να επανέλθουμε στις ε, παλιές, ε, στα παλιά συστήματα, στα συστήματα του χθε. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τη σημερινή ευκαιρία λοιπόν για να δημιουργήσουμε μια πιο καθαρή, πιο υγιή οικονομία, η οποία θα αποτελέσει το μέλλον, την εγγύηση για το μέλλον των παιδιών μας. Κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επουλώσει όλες τις πληγές που θα αφήσει πίσω της αυτή η κρίση, αλλά θα αναλάβουμε το τμήμα της ευθύνη που μας αναλογεί. Και αυτό το κάνουμε σήμερα, εξισορροπώντας την επιβάρυνση των κρατών μελών και εκ παραλλήλου διασφαλίζοντας ότι αυτή η τεράστια προσπάθεια θα έχει κάποιο θα έχει κάποια αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά το, από το μέλλον των νέων γενιών. Σας ευχαριστώ πολύ και ε, ζήτω η Ευρώπη. Ευχαριστούμε Πρόεδρε Φόντερ Λάιν και τώρα. Να ακούσουμε τους πρόεδρους των πολιτικών ομάδων, ο πρόεδρος Βέμπερ. Συνήθως ξεκινάω κατευθείαν ε, τις πολιτικές μας ε, παρεμβάσεις με τεχνικές ε, παρατηρήσεις. Αλλά σήμερα θέλω να μιλήσω πρώτα για τον κόσμο, για τα προβλήματα της αυτά που ανησυχούν τον ε, κόσμο. Η Μαδρίτη, για παράδειγμα, μία νοσοκόμα η οποία μολύνθηκε όσο βοηθούσε τον κόσμο. Ένα γιατρό στο Πέργαμο που καθημερινά παίρνει αποφάσεις ζωής και θανάτου όλοι αυτοί που βοήθησαν για την ανακοπή τη πανδημία. Αναφέρω τα παράδειγματα αυτά για να καταδείξω ότι οι ήρωε τη κρίση αυτή δεν είναι οι πολιτικοί, οι μάνατζερ, αυτοί που δουλεύουν στα μέσα ενημέρωση. Είναι τα εκατομμύρια Ευρωπαίοι οι οποίοι βοήθησαν να φροντίσουμε όλου εκείνου που χρειάστηκαν τη φροντίδα μα. Σα ευχαριστούμε από το βάθο τη καρδιά μα, όλου σα. δεν αρκούν τα λόγια για να σα ευχαριστήσουμε για τη δέσμευσή σα. Και τώρα έρχεται η στιγμή να κάνουμε και εμεί τη δουλειά μα ω πολιτικοί. Είναι η σειρά μα. Ως ΕΛΚ υποστηρίζουμε το γενικότερο σύστημα που προτείνεται σε ό,τι αφορά το πουδουπού και την προσανατολισμό στο μέλλον και το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο θα δώσει απάντηση στις ε, απαιτήσει του μέλλοντος. Αυτός ο μηχανισμός για μας ως ΕΛΚ το βασικό στοιχείο αυτό είναι να υπάρξει ένας δημοκρατικός ε, προπολογισμό, ο οποίος θα καθοριστεί από τον κόσμο που θα βασιστεί στην αλληλεγγύη μεταξύ εθνών και λαών. Ένας προπολογισμό που θα είναι τίμιο προ τον κόσμο και ο οποίο θα φροντίσει τον κόσμο. Θέλουμε να υπάρχει επικυριαρχία. Αυτό ήταν το βασικό ε, μήνυμα, ένα από τα βασικά μηνύματα της εκστρατείας του Brexit. Αυτό θεωρώ ότι αποτυπώνει το γεγονός ότι ο κόσμος δεν αισθάνεται ότι συμμετέχει στην διαδικασία της ε, Ευρωπαϊκή Ενοποίησης. Το θέμα λοιπόν είναι να καταλάβουμε ότι δεν αποφασίζει μια εξωτερική δύναμη για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι, ο βουλευτής μου είναι αυτός ο οποίος αποφασίζει για το μέλλον της Ευρώπης. Κανένας προπολογισμό λοιπόν χωρίς νομι... νομιμότητα. Δημοκρατική νομιμοποίηση. Αυτό είναι ευρωπαϊκό τρόπο ζωή και αυτή η υπόσχεση δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει έρθει λοιπόν σήμερα η στιγμή να ανταποκριθούμε στην υπόσχεση αυτή έχει έρθει η στιγμή να εξασφαλίσουμε και από πλευρά του Συμβουλίου με Δημοκρατική Ευρώπη για το μέλλον της Ευρώπης. Ένα δεύτερο θέμα που μας απασχολεί ο ΕΛΚ είναι ότι ο κόσμος δεν ανησυχεί για την ε, διαδικασία, μόνο για τα αποτελέσματα. Και έτσι το πνεύμα της αλληλεγγύης με τις τελευταίες εβδομάδες θα πρέπει να επικρατήσει. Θα πρέπει να κοιτάξουμε αυτού που έχουν πληχθεί ιδιαίτερα και κυρίως για τους νέους. Αυτού θέλουμε να βάλουμε στο επίκεντρο, στο δεύτερο σημείο μα. Τα τελευταία 12 χρόνια έχουμε ήδη ζήσει μια χαμένη γενιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκατομμύρια νεαροί οι οποίοι είναι καλά εκπαιδευμένοι, καλά προετοιμασμένοι, δεν είχαν ευκαιρίες να πετύχουν στην αγορά εργασίας. Και εδώ θέλω να υποστηρίξω το εξή η Ευρώπη δεν μπορεί να επιτρέψει και πάλι να υπάρξει μια χαμένη γενιά η οποία θα ατενίζει το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον τρόπο αυτό. Γι' αυτό χρειάζονται λοιπόν επενδύσεις η Ευρώπη. Θα πρέπει να δώσει στη νέα γενιά ελπίδα. Τρίτο σημείο που θέλω να υπογραμμίσω. Θα πρέπει να είμαστε ε, ειλικρινεί σε ό,τι αφορά το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και σε ό,τι αφορά τι υποσχέσει που δώσαμε στου εκλογεί μα πριν από πέρσι. Σωστά υπογράμμισε η Ουρσουλά von Το θέμα είναι οι επενδύσει στο κλίμα, το ψηφιακό κόσμο, ε, η έρευνα, η καταπολέμηση του καρκίνου, του κρονοϊού. Όλα αυτά λοιπόν προϋποθέτουν κοινή δράση. Να μην ξεχάσουμε επίσης και τις περιφερειές μας, τους αγρότες μας, το υπογραμμίζω, να είμαστε δίκαιοι προς όλους. Η συνοχή και η αγροτική πολιτική είναι ένα από του κλάδου όπου επιδεικνύουμε ήδη σήμερα αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει σωστή χρηματοδότηση. Και τέλο, τελευταίο σημείο, θα ήθελα να υπογραμμίσω το εξή. Θα πρέπει να φροντίσουμε την προετοιμασία για τι μελλοντικέ καταπήγουσε καταστάσει που θα αντιμετωπίσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε να υποσχεθούμε ότι θα καταφέρουμε να αποφύγουμε στο μέλλον μια τέτοια πανδημία. Κανεί δεν μπορεί να το υποσχεθεί αυτό, αλλά μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη θα είναι πιο καλά προετοιμασμένη για την επόμενη πανδημία, για την επόμενη κρίση. Χρειαζόμαστε ευελιξία, ιδίου πόρου. Θα πρέπει να υπάρχουν εργαλεία για να υπάρχει σωστή, δέουσα αντιμετώπιση μια μελλοντική κρίση. Μετά την κρίση, λοιπόν, θέλουμε να δούμε μια ευνομένη Ευρώπη όπου όλα τα τμήματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανακάμψουν. Μετά την κρίση θα θέλουμε να διαπιστώσουμε ότι η Ευρώπη θα επενδύσει σε μελλοντικά project, τα οποία θα δημιουργήσουν ένα μέλλον οικονομικό για τη μελλοντική γενιά. Και θέλουμε σε παγκόσμιο επίπεδο επίσης να υπάρξει μια Ευρώπη η οποία θα βγει ως πρώτη από την κρίση. Αυτός είναι ο στόχο μας και αυτή είναι μάλλον η στιγμή Σούμαν ε, της γενιά μας αυτής. Ε, για να χρησιμοποιήσω τα λόγια σας, θα πρέπει να μας δίνει θάρρος, το θάρρος και η τόλμη που είδαμε από τους νοσοκόμες, από τους γιατρούς, από όλους όσοι βοήθησαν τις τελευταίες εβδομάδες. Αυτούς πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ως παράδειγμα και να δράσουμε τώρα. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Πρόεδρε Γκαρθία Πέρεθ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρώτα-πρώτα θα ήθελα να σας πω ότι ε, είμαι ευγνώμων ότι μπορώ να βρίσκομαι εδώ τώρα και να τα συζητούμε γιατί περάσαμε δύσκολε ώρε σε όλε τι χώρε. Πάρα πολλοί από του συμπολίτε μα έχασαν τη ζωή του και πάρα πολλοί από αυτού ήταν αγαπημένοι μα, ήταν συγγενεί μα και τώρα έχουμε εκατομμύρια που έχουν μπροστά του τον, τον, τον φόβο για το μέλλον και πέραν αυτών των ε, δύσκολων στιγμών μπόρεσε το Κοινοβούλιο να συνεχίσει το έργο του με υπευθυνότητα χάρη στον πρόεδρο Σασόλη ο οποίος κατάφερε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είναι παράδειγμα ελεγγύης και χάρη στους υπαλλήλου του Κοινοβουλίου. Ε, την ώρα αυτή έχουμε επίγνωση της ιστορικής μας ευθύνης και όταν ο κόσμος ε, θεωρεί ότι τον έχουμε αφήσει στην τύχη του, ε, τότε υπάρχει εφορέδαφος για τον λαϊκισμό, τις εύκολες λύσεις, για τον ε, εθνικισμό. Οπότε αυτός που βγαίνει χαμένος είναι η δημοκρατία. Ε, γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική η απόφαση που θα λάβουμε τις αμέσως επόμενες μέρες και παρά την αρχική αντίδραση του Συμβουλίου. Γιατί φαινόταν ότι οι αργοί κρατών και κυβερνήσεων και ότι οι υπουργοί έριχναν το μπαλάκι ο ένας τον άλλο γιατί δεν θέλαν να αποφασίσουν. Αλλά τελικά στις 23 Απριλίου είχαμε ένα μήνυμα. Είχαμε κάτι που το πήρε ο κόσμος ως μήνυμα, δηλαδή αυτό το πρόγραμμα ανάκαμψης με αντίστοιχο δημοσιονομική κάλυψη, δηλαδή ούτως ώστε να αλλάξει το νέο ΠΔΠ. Οπότε τώρα αυτό το οποίο θέλουμε, ζητάμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φανεί φιλόδοξη, να έχουμε αυτό το κοινό κείμενο και τα μηνύματα να είναι ξεκάθαρα. Πρώτα-πρώτα, μήνυμα ενότητας, γιατί εμεί μπορούμε να ξεπεράσουμε τις ιδεολογικές διαφορές και τις εθνικές διαφορές, ούτω ώστε να μπορέσουμε να πασχίσουμε για το κοινό συμφέρον. Οπότε χρειάζεται αυτό το σχέδιο ανάκαμψη στα πλαίσια του ΠΔΠ, του, του δημοσίου κανονισμού, αυτά τα οποία εδώ αποφασίζουμε, οπότε και εμεί να αποφασίσουμε επίση ω με το Συμβούλιο. Οπότε τώρα κάτι άλλο, ένα άλλο μήνυμα είναι η φιλοδοξία, θα πρέπει η βιωσιμότητα, θα πρέπει η σύγκληση. Αυτά να είναι οι μπούσουλε που θα έχουμε, να δούμε πώ θα πιάσει τόπο αυτό το χρήμα, γιατί αυτό το ζητάει η κοινωνία, οι νέοι που μα λένε ότι δεν θα πρέπει να θυσιάσουμε το μέλλον του με το που να, παρα, να παρετηθούμε από μια πράσινη Ευρώπη, από μια βιώσιμη Ευρώπη. Το ζητάνε τα κοινωνικά δίκτυα, έχουμε την πρωτοβουλία We Move Europe. Οπότε αυτό θέλει η κοινωνία των πολιτών. Θέλει να συνεργαστεί μαζί μα για μια καλύτερη Ευρώπη, διότι η Ευρώπη Κυρίες και κύριοι, δεν είναι ε, κάτι που είναι η διοκτησία μας θα πρέπει τώρα να εκμεταλλευτούμε κάθε στάλα ενέργειας που έχουμε. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τους πιο δύνατους οπότε. Ο βασικός άξονας μας θα πρέπει να είναι η κοινωνική πολιτική. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τους πιο ευάλωτους και θα πρέπει να δώσουμε εγγύσεις για απασχόληση και δεν θα πρέπει να παραιτηθούμε από τέτοιες πρωτοβουλίες. Επίσης θα πρέπει να επενδύσουμε σε κάποιο είδους μετασχηματισμό ψηφιακό με δικαιοσύνη. Οπότε να δούμε τι πιο επίγουσες πολιτικές. Ο θα πρέπει να δοθούν 2 ευρώ. Βέβαια είναι δύσκολο τώρα να ζητήσουμε με χρήμα από τα κράτη, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να δούμε τι θα γίνει με το 2% για τους ιδίους πόρους, 2% του ΑΕΠ, να δούμε μήπως μπορούμε να έχουμε αυτά τα κορονομόλογα και επίσης θα πρέπει να έχουμε τις ε, ενισχύσεις, να πρέπει να υποστηρίξουμε τα δάνεια, θα πρέπει να είναι μακροπρόθεσμα αυτά τα δάνεια για να μπορούμε να βοηθήσουμε την οικονομική ανάκαμψη. Κυρία Φοντερ ε, ε, σωστά λέτε για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και δεν ξέρω αν το Συμβούλιο θα δεχθεί ότι το το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο συνδέεται με τόσο φοβερά θέματα όπως τη βιωσιμότητα για το περιβάλλον, τα κοινωνικά και όπως τους στόχους για την βιωσιμότητα. Ε, βέβαια, θα θυμάστε τι έγινε στο παρελθόν. Θα πρέπει να το θυμόμαστε στο παρελθόν για να αντιλήσουμε συμπεράσματα και έτσι να, ε, να ταινίζουμε το μέλλον. Και θέλω να πω σε Κομισιόν και Συμβούλιο ότι αυτή τη στιγμή ε, έχουν σημαντικέ ευθύνε. Το δέκινο Βούλιο. θα σα στηρίξει. Θα σα στηρίξει και θα προχωρήσουμε χέρι-χέρι, θα βάλουμε πλάτη. Αλλά θέλουμε να έχετε φιλοδοξία και θέλουμε να δώσετε προτεραιότητα στο κοινό συμφέρον και όχι στα, στα εθνικά καλέσματα. Άρα ε, θάρρος, γενναιότητα και φιλοδοξία. Αυτό θέλουμε. Ευχαριστούμε. Πρόεδρε Σόλος, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, Πρόεδρε Μισελ, Πρόεδρε Φοντερ Λάιον. Ο Σούμαν είπε πριν από 70 χρόνια ότι η Ευρώπη δεν θα χτιστεί μέσα σε μια νύχτα, αλλά βήμα το βήμα, λιθαράκι το λιθαράκι. Η υγειονομική κρίση του COVID-19 δείχνει ότι μπαίνουμε σε μια τεράστια οικονομική κρίση και η εμπειρία των τελευταίων 70 ετών δείχνει ότι η Ευρώπη έχει προχωρήσει ε, ιδίως ιδίω όταν αναγκαζόταν και εξαναγκαζόταν να βρει λύσεις σε κρίσεις. Εδώ λοιπόν δεν θα πρέπει να μα απασχολήσει μόνο πώ θα ανακάμψει η οικονομία μετά την κρίση, αλλά θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε κάθε δυνατότητα για να ανοικοδομήσουμε, να εκμεταλλευτούμε όλε τι τεχνολογικέ λύσει που υπάρχουν. Δεν μπορούμε να πάμε πίσω στην οικονομία του 20ου αιώνα. Πρέπει να θέσουμε νέα θεμέλια, δίνοντα μεγάλη σημασία στο περιβάλλον, την ψηφιοποίηση και στρατηγικού τομεί όπω ε, η υγειονομική περίθαλψη. Αυτά θα είναι στην καρδιά τη ανοικοδόμηση τη ε, οικονομία που θέλουμε θα πρέπει να φροντίσουμε, να προστατεύσουμε εκατομμύρια πολίτες που έχασαν ή χάνουν ε, τις δουλειές τους ή εκατοντάδες εταιρείε που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες. Ε, τόσους ανθρώπους ε, που δυσκολεύονται λόγω του υπερφορτωμένου νομικού μας συστήματος και σε τομείς όπως ο τουρισμός, οι μεταφορές ή η γεωργία ε, άνθρωποι που αντιμετωπίζουν εργασιακά προβλήματα. Θα πρέπει να πάυσουν οι διχασμοί της Ευρώπης ανατολικά, δυτικά ή μεταξύ βορρά και νότου. Θα πρέπει να κοιτάξουμε να υπάρξει ένα πρόγραμμα ανάκαμψης με φρέσκο χρήμα. Αυτό θα είναι η μεγαλύτερη δημοκρατική ενέργεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μια πρωτοβουλία που εμείς ως άμεσα εκλεγμένοι από τους πολίτες θα θέσουμε για το μέλλον ως ένα κοινό όραμα, όχι μόνο για τα κονδύλια και το χρήμα. Ε, θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε. Θα πρέπει να γίνει η οικονομία μας ε, μια οικονομία που να λειτουργεί όσο το δυνατόν συντομότερα. Διότι οι κοινωνίες μας θα πρέπει να επανεπινοήσουν τους εαυτούς τους μετά την κρίση. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να μας απασχολήσει και οι δικαιούχοι θα πρέπει να ζήσουν τη διαφορά, να καταλάβουν στην πραγματική οικονομία ότι του υποστηρίζουμε. Οι άνθρωποι έχουν κάνει τι δουλειέ του, οι εταιρείε και οι επιχειρήσει έχουν πτωχεύσει χωρί να φταίνε. Εμείς πρέπει να τους υποστηρίξουμε και εμείς θα πρέπει να πολεμήσουμε για να υπάρξουν οι απαραίτητοι πόροι. Οποιαδήποτε άλλη πρόταση που δεν προβλέπει επαρκή πρικοδότηση για του ερχόμενου προπολογισμού και το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να απορριφθεί. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε του αναγκαίου πόρου και από τον πολιτή προπολογισμό, ώστε να υπάρχει σταθερότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρί να πιέζονται οι εθνικοί προπολογισμοί. Επίση, η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώ και το κράτο δικαίου θα πρέπει να παραμένουν για μα πραγμάτευτα και αναπαλωτρίωτα. Θα πρέπει λοιπόν και η ομάδα Renew, όταν γκριθεί το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο να ε, βεβαιωθεί ότι η Ευρώπη δεν θα βασίζεται σε λαϊκισμού ούτε σε εξτρεμισμού, αλλά θα συνεχίσει να προστατεύει αξίε το κράτος δικαίου και μια εύρυθμη ε, δικαιοσύνη, ένα σύστημα δικαιοσύνη που θα λειτουργεί. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε τώρα τη σωστή επιλογή. Μια επιλογή που ελπίζω ότι θα έχει μία και μόνη απάντηση. Και η απάντηση αυτή είναι μαζί. Μαζί από κοινού μόνο μπορούμε να δώσουμε θαραλές τολμηρές απαντήσεις στις αγωνίες των πολιτών πολίτες που μας εξέλεξαν μόλις πριν από ένα χρόνο, ε, ενάμιση χρόνο. Θα πρέπει λοιπόν να τους δείξουμε ότι έχουμε το θάρρος, αυτά που υποσχεθήκαμε στις προεκλογικές μας εκστρατείε όταν τους απευθυνθήκαμε και τους ε, μιλήσαμε για μια δικαιότερη Ευρώπη, τώρα θα πρέπει να γίνουν πραγματικότητα. Η Ευρώπη θα πρέπει να βασίζεται σε μια πραγματική αλληλεγγύη και όχι δηλώσεις. Ευχαριστούμε για την ομάδα ID, ε, ταυτότητα και δημοκρατία. Ο συνάδελφος κ. Φαναντρίσσα, αξιότιμοι συναδελφοί, όπως και στο Τσέρνομπιλ, ένα κομμουνιστικό καθεστώς προσπάθησε να κρύψει την αλήθεια για τα όσα είχαν γίνει και να αρνηθεί την ευθύνη της και να αρνηθεί ε, αυτά που της αναλογούσαν σήμερα, θα πρέπει να δούμε κάτι ανάλογο. Τα ευρωπαϊκά ε, κράτη ε, χρειάστηκε να ε, ζητήσουν, να κλειπαρίσουν για να υπάρχει σωστή ε, προετοιμασία και προστασία. Στην Κίνα αντιμετώπισαν dumping, διάφορες μεθόδους κατάχρησης της αγοράς και την αφέλεια των δυτικών πολιτικών. Και σήμερα έχουμε 146 δις ευρώ ζημία και έχουμε επίσης ε, ένα κίνδυνο οικονομικής απεικιοκρατία, από μια ε, κομμουνιστική δικτατορία. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τη σχέση μας με την Κίνα. Θα πρέπει στρατηγικούς τομείς να τους προστατεύσουμε από τις επιθετικές ε, κινέζικες κινήσεις. Θα πρέπει να πούμε γεια στην αφέλεια κατά της Κίνας και να κάνουμε μια νέα βιομηχανοποίηση της Ευρώπης και κυρίως μετά την μεταναστευτική κρίση και την οικονομική κρίση δεν μπορεί να είναι και πάλι ο πολίτης ο οποίος θα πληρώσει την κρίση. Θα πρέπει να δούμε σε ό,τι αφορά και τους ε, φόρους ε, κορονοϊού στις κινησικές επιχειρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σίρντουμπαν. Λάμπερτ, συγγνώμη. Δεν το θεωρώ ντροπή μου να με ονομάζετε Σέντεβαν, αλλά εν πάση δεν είμαι. αυτοί που βοηθούν σε, σε κάθε μέτωπο, στη, στο, στα νοσοκομεία, στο δρόμο, αυτοί που βοηθούν κατοίκον, όλοι αυτοί ε, κάνουν τη ζωή τους, όλο αυτό μας δείχνει την ελληνική, αυτούς που έχουν ε, ε, απομονωθεί και θα πρέπει όμως να υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες εδώ και ε, τρεις μήνες υπάρχει ευθύνη ε, αλλά ε, ανυπομονούν και έχουν δίκιο γιατί ε, ρωτάνε τι, τι, γίνεται, τι, τι, τι κάνουν οι ηγέτες. Συμφωνώ, θα πρέπει να έχουμε αλληλεγγύη και θα πρέπει να μειωθούν οι αποκλήσεις στην Ευρώπη, αλλά όταν βλέπουμε το τι, γίνεται, πώς αντιδρούν οι, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, τότε βλέπουμε ότι καθυστερούν και ότι ο καθένας κοιτάει την πάρτη του. Οπότε αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να δούμε τι, τι συμπεράσματα θα αντιλήσουμε γιατί ξέρουμε ότι ε, υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί. Είναι βέβαια σε Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα δεν ήταν πάντοτε τέ, τέλεια αλλά ούτε και στις ε, κάτω χώρες ήταν πάντοτε τέλεια. και επίσης ε, η Γερμανία πάντοτε υπερασπίστηκε την αυτοκινητοβιομηχανία που είχε κάνει ε, τόσες ε, αμαρτίες και ε, ταυτόχρονα βλέπουμε ότι η Ελλάδα, Ισπανία και η Ιταλία κάνανε πολύ περισσότερα για το μεταναστευτικό από όσο τους αναλογούσε και όλα τα κράτη-μέλη ε, έχουν στιγμές επιλήψιμες ε, και όλοι μπορούν να βάλουν το λιθαράκι τους για να προχωρήσουμε. Οπότε να αφήσουμε τις ηθικολογίες. Αυτό το οποίο τώρα διακυβεύεται είναι ε, όλη αυτή η διαδρομή των 70 ετών. Είναι θεμέλιο η αλληλεγγύη, το κοινό συμφέρον. Να υπάρχει μια ευημερία βιώσιμη για τους συμπολίτε μας και έτσι να μπορέσουμε ε, μαζί να ε, ανταποκριθούμε στα προβλήματα και έτσι να δούμε πώς μπορούμε να σκεφτούμε και να υλοποιήσουμε μια στρατηγική για την οικονομική ανάκαμψη και ε, η βασική αρχή είναι ο καθένας όσο μπορεί προς όποιον όσο χρειάζεται. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς θα χρηματοδοτήσουμε αυτή την προσπάθεια και μόνος χρειάζεται ένα κοινό προπολογισμό, ε, θα πρέπει να γίνει επανεκκίνηση στην οικονομία, χρειάζεται κάποιο είδους άλμα ποιοτικό, κοινοτικό, ε, γιατί θα πρέπει να το καταφέρουμε αυτό με την ε, νομισματική πολιτική μας και έκανε ο κόσμος ό,τι μπορούσε και τώρα οι ηγέτες θα πρέπει Τώρα εσείς να κάνετε αυτό που σας αναλογεί, είναι ε, ιστορικές στιγμές, κανείς δεν θα συγχωρήσει αν δεν κάνετε ό,τι πρέπει. Ευχαριστώ Πρόεδρε Λάμπερτ. Ευχαριστούμε Πρόεδρε Λάμπερτ, ο κύριος Φανόβερτφελτ για τους ε, συντηρικούς και μεταρρυθμιστές. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, Πρόεδρε. Ε, συνάδελφοι, κοιτώντα τι τελευταίε εβδομάδε, δεν εμπόζει ότι μπορούμε να πούμε ότι η, Ευρώπη είχε σωστή και έγκυρες αντιδράσεις στην πανδημία, αλλά μπορούμε να αντισταθμίσουμε τα πράγματα τις επόμενες εβδομάδες σε ό,τι αφορά τη συζήτηση για το πολιτισμό πλαίσιο και το σχέδιο ανάκαμψης που θα ψηφιστεί αύριο και το οποίο θα περιλαμβάνει σαφείς ενδείξεις για τα αυτά που χρειάζονται και θα υποστηρίξει και η ομάδα μου. Θα μιλή, μιλάμε για πολλά χρήματα το οποίο είναι και φυσιολογικό γιατί η έκταση και η σοβαρότητα της κρίσης αυτή προϋποθέτει σημαντική οικονομική, δημοσιονομική ε, επέμβαση, αλλά θεωρώ ότι συχνά χάνουμε την προσοχή μας ε, για πράγματα τα οποία δεν κοστίζουν χρήματα και τα οποία μπορούν να έχουν ε, μεγάλη επίδραση για την καταπολέμηση της πανδημίας και για την οικονομική ανάκαμψη. Τα ανέφερε αυτά και η Επίτροπος Φοντερ σε ό,τι αφορά τη σημασία της ενιαίας αγοράς. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το τονίσουμε παρκώς αυτό, το πόσο σημαντική είναι αυτή η ιστορική ενιαία αγορά για τις οικονομικές δραστηριότητε. Δεύτερο σημείο, οι επενδύσεις. Φυσικά είναι πολύ σημαντικές ε, δημόσιες και ιδιωτικέ επενδύσεις και πιστεύω ότι πρέπει πλέον να αφήσουμε πίσω μας τους πολύ αυστηρούς ε, κανόνες του Eurostat σε ό,τι αφορά τις δημόσιες επενδύσεις, το οποίο αποτρέπει τη σωστή λειτουργία της οικονομίας. Τρίτο σημείο, και νομίζω ότι ένα σημείο το οποίο είναι όλο και πιο σημαντικό σήμερα, είναι η ανάγκη να υπάρξει γεωπολιτική προστασία. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν ε, διεθνείς ομάδες και επενδυτικά ταμεία τα οποία ε, καθημερινά κερδίζουν δισεκατομμύρια Υπάρχει ένας ε, πόλεμος ε, ρευστότητας, αλλά υπάρχει και ένας ε, πόλεμος στις αγορές. Θα πρέπει να λάβουμε λοιπόν αυστηρά μέτρα σε ό,τι αφορά τις επιθετικές αναλήψεις. Τέλος, χρειάζεται αποφασιστικότητα για να ξεπεράσουμε τον φαύλο κύκλο της ασάφειας και του φόβου, γιατί αυτό θα έχει επιπτώσεις στην ανακαμψή μας τις επόμενες εβδομάδες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, ο πρόεδρος Σύρδεβον. Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Και δεν ήταν τόσο άσχημα αυτά που μας είπε ο Φίλιπ. Θα μπορούσα να συμφωνήσω και εγώ με κάποια από αυτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε ένα μπροστά σε, ένα, σε μια διχάλα. Κατά πόσον θα συνεχίσει την πολιτική αυτή που ασκούσε ως τώρα και θα αποτύχει ή θα μεταφραστεί σε ένα πραγματικά μεγάλο έργο αλληλεγγύης τόσα χρόνια μετά την διακήρυξη Σούμαν. Και βλέπουμε ότι ο Ευρωπαίος, ο Ευρωπαϊκός λαός περίμενε ένα σαφές μήνυμα της αλληλεγγύης και της ενότητας. Παράλληλα όμως τα κράτη-μέλη τσακώνονται και ο κύριος Μισελ επί εβδομάδες και όλη αυτή την περίοδο διαπιστώνουμε ότι αυτοί που πληρώνουν τελικά το τίμημα με κακούς ε, μισθούς και κακές συνθήκες εργασίας τόσα χρόνια δεν έχουν επαρκές ε, υποδομές. Αυτοί λοιπόν οι εργαζόμενοι χρειάζονται όχι μόνο τις ευχαριστίες μας κύριε Βέμπερ αλλά και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Βλέπουμε τον ευρωπαϊκό ε, μηχανισμό ο οποίο δίνει 240 δισεκατομμύρια ω πιστώσεις. Τι γίνεται όμως όταν θα επανέλθουν ε, οι κανόνες για τα χρέη. Δεν θα υπάρξουν νέε κρίσει ε, χρεών, υπερχρέωση στα κράτη-μέλη. Και τι θα κάνουμε για να υπάρχει ένα σύστημα για να δούμε τι γίνεται στις συντάξεις, στους μισθούς. Ε, θα κληθούν όλοι να τους περικόψουν και ποιοι τελικά θα επιβαρυνθούν από την κρίση του κορονοϊού. και η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου δεν σημαίνει τίποτα παραπάνω παρά από ιδιωτικοποίησει και περικοπέ σε ό,τι αφορά και τι επενδύσει τι απαραίτητε υποδομέ. Να σταματήσουν και τα έργα εκείνα τα οποία χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ψηφιακή καμπή, το νέο πράσινο σύμφωνο, όλα αυτά χρειάζονται. Έχει έρθει λοιπόν στιγμή να θέσουμε εκτό λειτουργία επιτέλου διαπαντό το Σύμφωνο Σταθερότητα και Αναπτύξη σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση τη εντετεκοσποίηση και όλες αυτές τις τάσεις οι οποίες θα ανατραπούν. Είμαστε λοιπόν αντιμέτωποι με μεγάλα ερωτήματα σε ό,τι αφορά την οικονομική ανάκαμψη της Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς μπορούμε να την πετύχουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο, μάλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έλαβε το δύσκολο έργο από το Συμβούλιο να βρει ένα, όχι γεωμετρικό, ε, μια γεωμετρική λύση, μια πολιτική λύση, μια τολμηρή λύση. Χρειάζονται λοιπόν σημαντικά ίδια μέσα, χρειάζονται ένας ψηφιακός φόρος, ένας φόρος δημοσιονομικών συναλλαγών και από φορολόγηση των μεγαλύτερων ε, περιουσιών των Ευρωπαίων. Και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα και το μερίδιό τους ε, που τους αναλογεί για την ε, οικονομική ανάκαμψη. Τα μέσα αυτά θα χρησιμοποιηθούν ως επιχορηγήσεις, ως πιστώσεις προς τα κράτη-μέλη δεν ήταν σαφές από την ομιλία σας. Αν είναι πιστώσεις, αυτό θεωρώ ότι αυξάνει πρετέρω την ε, πιθανότητα μια μελλοντικής ε, κρίσης ε, υπερχρέωσης των κρατών μελών μετά τον κορονοϊό και μετά πώς θα βρούμε τα βήματα για μία έκτη η οποία θα υποστηρίζει άμεσα την ευρωπαϊκή οικονομία. Χρειάζεται λοιπόν τόλμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τα πού θα κινηθεί προς τον οδό της λιτότητας ή της αλληλεγγύης. Εμείς έχουμε αποφασίσει από πλευρά της ομάδας μου. Θέλουμε με τον ευρωπαϊκό λαό να ακολουθήσουμε τον δρόμο της αλληλεγγύης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ με την προσοχή σας. Ευχαριστούμε ο κύριος Καστάλντο, μη εγγεγραμμένος. Ευχαριστώ πρόεδρε, πρόεδροι, συνάδελφοι. Ο χρόνος δεν έχει τιμή, αλλά δεν έχει και ε, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει αξία. Δεν μπορεί κανεί να τον κρατήσει, αλλά δεν μπορεί και να τον δαπανίσει. Μόλι τον ξοδέψει κανεί, δεν μπορεί να τον πάρει πίσω. Χρειάζεται λοιπόν ε, χρόνος και από όσα έχουμε προβλέψει αυτό το χρόνο που πέρασε, ε, μόνο ένα θα έχει σημασία, το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε στην δημοκρατική επιλογή της έγκρισης του πολιτισμού δημοσιονομικού πλαισίου, όπω είπε και η πρόεδρος Φόντερ Λάιεν, θα πρέπει να φροντίσουμε να έχει τις κατάλληλες ε, κατευθύνσεις ε, το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να μην ζητήσουμε στα ε, κράτη που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση λόγου χάρη να συμβάλλουν περισσότερο από ό,τι παλιότερα. Όπω είπε και το Κοινοβούλιο, χρειάζονται νέοι ε, ήδη πόροι. Χρειάζονται ε, υποψηφιακό φόρο, ε, ο φόρο για τι εκπομπέ του αερίου του θερμοκηπίου και θα πρέπει η πρότασή μα να είναι έτοιμη μέσα στο καλοκαίρι, με τόλμη. Διότι οι γιατροί μα ε, έχουν δείξει την τόλμη του. Αναλόγω πρέπει και εμεί να δείξουμε τη δική μα τόλμη για να σώσουμε ζωέ. Δεν μπορούμε να παραμένουμε στι εθνικέ εγωπάθειε αν θέλουμε να ξεφύγουμε από κοινού ε, από αυτή τη μεγάλη κρίση. Αυτή είναι η στιγμή τη αλήθεια. Ευχαριστούμε. Στο τέλος αυτού του γύρου ζήτησε ξανά το λόγο ο πρόεδρος Μισελ, ότι θα πρέπει να ε, εξέλθει ε, και θα ήθελε να κάνει κάποιες παρατηρήσεις πριν την αποχώρησή του. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Ευχαριστώ για όλα τα μηνύματα που απευθύνθηκαν ως τώρα. Μερικές σύντομες παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, ε, ό,τι και αν λένε, η αντιρρησίες, ε, λαϊκιστές, δημαγωγοί ε, και εξτρεμιστές που καταφέρονται κατά της Ευρώπης έδειξαν παρόλα αυτά ότι η Ευρώπη μας έχει μια αξία ανεκτήμητη για την προστασία του κράτους δικαίου, των δικαιωμάτων, της ευημερία των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτό το ευρωπαϊκό κεκτημένο πέρα από τους λαϊκισμούς και τους εξτρεμισμούς πρέπει να το προσπιζόμαστε. Και έπειτα το είπατε, ο καθένας, κάθε μια από εσά, το είπατε με διαφορετικούς τρόπους, όλοι ερχόμαστε αντιμέτωποι με τα προβλήματα και τώρα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις ευθύνες μας αυτήν την στιγμή που είναι καθοριστική για τη γενιά μας. Πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Σωστά το είπατε κύριε Βέμπερ. Δεν είναι η στιγμή να κάνουμε ανταγωνισμό του ποιος νομιμοποιείται περισσότερο από άλλους. Τα θεσμικά όργανα της Ευρώπης είναι νομιμοποιημένα όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που εκλέγεται απευθείας από τους Ευρωπαίους πολίτες και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όπου έρχονται οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις κάθε εβδομάδα και εδώ και δεκαετίες, χρόνια λαμβάνουν τις αποφάσεις των λαών που τους ανέθεσαν την την αρμοδιότητα αυτή. Και βεβαίω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να είναι κινητήριο δύναμη για όλα αυτά. Για την ε, πολιτική διάσταση αυτού του αγώνα και για τον δυναμικό χαρακτήρα που θα πρέπει να έχει. Ναι, είστε πεπισμένοι ότι από τη δική μου την πλευρά θα κάνω όσα χρειάζονται με τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ώστε ε, να μην έχουμε μια στήρα ε, αντιπαράθεση σε θεσμικό επίπεδο, αλλά να ανασκουμποθούμε, να πιάσουμε τη δουλειά και να στρωθούμε σε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Ποιο είναι το ποσό για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, ποιο είναι για το Ταμείο Ανάκαμψη, ποιο είναι ο τρόπο να χρηματοδοτηθεί, ποιο είναι ο τρόπο να γίνει ο επιμερισμό των πόρων και των κονδυλίων, για να βεβαιωθούμε ότι θα υπάρχει πολιτική συμβαστική λύση που θα εξυπηρετήσει του Ευρωπαίου πολίτε. Πώ θα προχωρήσει η ψηφιακή ατζέντα, πώ θα ε, γίνουν ε, όλα αυτά σωστά. Τα προβλήματα του παρελθόντο δεν έχουν εξαλειφθεί. Όμω θα πρέπει τώρα να βρούμε ε, έναν τρόπο να προσφέρουμε ξανά ελπίδα, αισιοδοξία. Διότι στην Ευρώπη έχουμε και ταλέντα και ε, πόρου και οι βασικοί μα πόροι είναι Ευρωπαίοι πολίτε, άντρε και γυναίκε. Γι' αυτό τώρα πρέπει να σταθούμε στο ύψο των περιστάσεων και να είστε βέβαιοι ότι την ε, χείρα που απευθύνεται από το Κοινοβούλιο προ το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα την ε, ανταποδώσουμε και θα φροντίσουμε να συνεργαστούμε στενά για να αντιμετωπίσουμε την κοινή μας πρόκληση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ευχαριστούμε Πρόεδρε Μισελ. Ευχαριστούμε Πρόεδρε Μισελ. Να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας ο κύριος Μουρεσάν. Έχετε 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι. Απ' την αρχή αυτή της κρίση η Ευρωπαϊκή Ένωση βοήθησε όπου χρειαζόταν ε, γιατρούς, προσωπικό, εκεί όπου χρειαζόταν ε, υλικά, ε, φάρμακα να πάνε εκεί όπου χρειαζόντουσαν περισσότερο. Και ε, επίση και οι κοινοτικοί πόροι θα πρέπει αντίστοιχα να κατανεμηθούν. Ε, προτείναμε μέτρα, συμφωνήσε το Κοινοβούλιο, τώρα θα πρέπει να προετοιμαστούμε για το μέλλον και για να μπορέσουμε να έχουμε τις πιο σωστές αποφάσεις θα πρέπει όλα τα ε, ευρωπαϊκά όργανα να είναι κοντά στον κόσμο, εκεί όπου οι τοπικές αρχές γνωρίζουν το τι συμβαίνει. Θέλουμε να εμπλακεί το Κοινοβούλιο όσον αφορά ε, το σχέδιο ανάκαμψης σχεδιασμός έγκριση και υλοποίηση αυτού του σχεδίου. Έτσι θα είναι καλύτερα. Ε, παντού προτείνει η κυβέρνηση και το κοινοβούλιο εγκρίνει. Πάντα γίνεται αυτό για τον προπολογισμό και σήμερα πέντε πολιτικές ομάδες έχουμε πρόταση ψηφίσματος όποτε θέλουμε να είναι φιλόδοξο αυτό το σχεδίο ανάκαμψης, δάνεια, χορηγίες, ε, να βοηθήσουμε, να κάνουμε τη διαφορά και έτσι να προσπαθήσουμε να ελαφρώσουμε το βάρος των κρατών μελών εκεί ε, ε, όπου θα πρέπει να επιστρατεύσουμε τους ίδιους πόρους μας και επομένως να μπορέσουμε να έχουμε ένα πι, δέλτα πι προσανατολισμένο προς το μέλλον. Να μην παραλείπουμε να προσέξουμε αυτές τις προτεραιότητες που έχουμε τάξει. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, συνάδελφε Μούρισαν. Και τώρα 1,5 λεπτό το λόγο έχει ο κύριο Ερτούγκ. Το μικρόφωνο σας, αν θέλετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχά να ξεκινήσω ε, με τις ευχαριστίες μου προς ε, όλους εκείνους τους γιατρούς ε, και νοσοκόμους και να μην ξεχνάμε και τους γονείς εκεί έξω αγαπητοί συνάδελφοι που εδώ και μήνες φροντίζουν τα παιδιά τους στο σπίτι προσπαθούν να διδάξουν τα παιδιά τους δεν έχουν όλοι τους κήπους που χρειάζονται και θα πρέπει να του ευχαριστήσουμε και αυτός και σε τέτοιες εποχές ε, κοινωνική απόσταση. Είναι σημαντικό να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και ευχαριστώ την κυρία Πρόεδρο για τους στόχους που περιέγραψε. Νομίζω ότι θα είναι μία αναστρέψιμο το γεγονό ότι τα κράτη-μέλη εδώ θα πρέπει να βάλουν το χέρι βαθιά στην τσέπη γιατί Λυπάμαι που έφυγε και νωρίς ο κύριος ε, Μισελ. Τουλάχιστον 2% του, ε, των ίδιων πόρων ως ανατολόριο είναι σωστό. Και νομίζω ότι σήμερα είναι καθοριστικό οι στόχοι που περιγράψαμε με τους σωστούς ε, μηχανισμούς να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Μιλήσατε για την ψηφιοποίηση, πολύ σωστό. Χρειαζόμαστε μια νέα κινητικότητα, επενδύσεις εκεί που χρειάζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και να μην ξεχνάμε επίσης να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το γεγονός αυτό, για τον δρόμο που χάραξε σήμερα για να ανοίξει τα σύνορα σταδιακά και για την ενίσχυση του τουρισμού. Θεωρώ ότι και αυτό θα έχει αποτέλεσμα. Γι' αυτό λοιπόν σα εύχομαι μεγάλη επιτυχία, κάθε επιτυχία για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα για δύο λεπτά ο κύριος Γκαρικάνο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρία Φαντερ Λάιεν. Όπως βρισκόμαστε και καταπολεμούμε την πανδημία αυτή, Αντιμετωπίσουμε τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση των τελευταίων 100 χρόνων. Όταν θα βγούμε, για να βγούμε από την κρίση αυτή θα χρειαστεί να κινητοποιήσουμε μεγάλο όγκο επενδύσεων, δημόσιων επενδύσεων, γιατί έχουμε πολλά κράτη που είναι υπερχρεωμένα και πολύ επιφαρημένα για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Η Ευρώπη λοιπόν θα πρέπει να άρθει στον ύψο των περιστάσεων για να χρησιμοποιήσουμε αυτό το σχέδιο να μου επιτρέπετε να το α, περιγράψω έτσι. Μιλάμε για ένα πακέτο ανάκαμψη 2-3 από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από ομόλογα ανάκαμψη, θα μας επιτρέψει να επενδύσουμε στον ιατρικό κλάδο, στο πράσινο σύμφωνο, στην ψηφιοποίηση, σε όλες αυτές τις προτεραιότητες. Το βασικό ερώτημα είναι το πώ θα χρηματοδοτηθεί ένα τέτοιο σχέδιο. Εδώ στο Κοινοβούλιο έχουμε πέντε ομάδες οι οποίες ε, κάνουν μία ε, προσφέρουν μια συμφωνία προς τα κράτη-μέλη. Λέμε ότι καταλαβαίνουμε ότι βρίσκεστε σε δενή κατάσταση και ότι είναι δύσκολα τα πράγματα για σας. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι θα πρέπει αυτές οι μακροπρόθεσμα δάνεια για το σχέδιο αυτό θα πρέπει να ε, πληρωθούν με ίδιους πόρους. Αυτοί που δεν πληρώνουν αυτά που τις αναλογεί, οι μεγάλοι τυπαίνοντες, οι ψηφιακές εταιρείε που δεν ε, δίνουν αυτά που τους αντιστοιχούν. Αυτό το σχέδιο είναι οικονομικά ορθό γιατί χρειάζονται αυτές τι επενδύσεις. Είναι πολιτικά εφαρμόσιμο. Θα το δείτε αυτό αύριο. Θα μετρήσετε τις ψήφους αυτές. Είναι εφικτό να έχουμε ένα τόσο φιλόδοξο σχέδιο και είναι και οικονομικά εφικτό γιατί οι πολίτε μα. Ε, αναζητούν καλά οχήματα επενδύσεων για το μέλλον. Χρειάζεται αυτά. Υπάρχει ζήτηση. Πριν από 70 χρόνια, αγαπητέ Πρόεδρε, συνάδελφοι, ο Ρόμπερτ Σούμαν είπε ότι θα πρέπει να έχει συγκεκριμένη διάσταση και διαμόρφωση η Ευρώπη. Αυτή είναι η στιγμή λοιπόν να οικοδομήσουμε συγκεκριμένα το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Γκαρικάνο. Για 1,5 λεπτό η κυρία Ντονάτου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι ίδιοι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα ε, αποτελούν τον ευρωπαϊκό προπολογισμό είναι εθνικές συνεισφορές από το φόρο προστατέμενης αξίας και ε, το φόρο επί του ΑΕΠ. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει απευθεία τον ευρωπαϊκό προπολογισμό σε αντίθεση με άλλες εθνικές τράπεζες, ούτε υπάρχουν δυνατότητες για άλλους ίδιους πόρους που να μεταφράζονται και δεν θα πρέπει να γίνει αυτό σε περισσότερους φόρους για τους Ευρωπαίους πολίτες. Το εργαλείο στο οποίο θα πρέπει να βασιστούμε και να βασιστεί η Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη, το Ταμείο για την Ανάκαμψη. Δηλαδή θα πρέπει να ε, μην είναι απλώ κέρδη για κάποιου και σκέτε απώλειε ε, για του ε, υπόλοιπου. Θα πρέπει όσοι μπορούν να χρηματοδοτήσουν μόνο του την οικονομία του, που αρνούνται την οποιαδήποτε ευελιξία για τα ευρωομόλογα ή για την διαφορετική μεταχείριση των υπόλοιπων προπολογισμών και του εθνικού χρέου, να μην συνεχίσουν ακάθεκτοι. Θα πρέπει Ευρωπαίοι πολίτες που δεν έχουν καμία ευθύνη και καμία ενοχή σε όσα συμβαίνουν να μην συνεχίσουν να πλήττονται, ούτε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να συνεχίσει το ρόλο του παρελθόντος. Μέχρι τώρα ε, ποιο θα μπορεί να παράγει το απαραίτητο κέρδος για να αποπληρωθεί το οποιοδήποτε χρέος εάν οι πολίτες δεν μπορούν να πάνε στις δουλειές τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν δεν μπορεί να συνεχίσει να κραδένει συνθήματα και σλόγγαν χωρίς να φέρνει συγκεκριμένα τα αποτελέσματα. Πρέπει να υπάρξει μια άρδιν ε, μεταρρύθμιση και ανανέωση Ένωση και στον ίδιο την εντολή τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εάν δεν γίνει κάτι τέτοιο, όσα λέμε θα παραμένουν μόνο συνθήματα και δεν θα έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Θα είμαστε τελείω μέτροι, διότι πολλοί θα είναι οι πολίτε που θα έχουν μείνει εκτό τη όλη πρόοδου. Ευχαριστούμε. Και για δύο λεπτά ο συνάδελφο Έκχαουτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους. Ακούσαμε ξανά ότι χρειάζεται ανάληψη δράση προηγούμενο και ότι μια τέτοια βαθιά κρίση δεν έχουμε βιώσει ποτέ στο παρελθόν και τώρα χρειαζόμαστε λύσει. Ε, πολύ συχνά η Ευρώπη δίνει πάρα πολύ μεγάλε υποσχέσει, αλλά όχι αποτελέσματα όταν μιλάμε για αλληλεγγύη και συνεργασία. Αυτή τη φορά αυτό δεν επιτρέπεται. Οπωσδήποτε η δράση αναβάλλεται. Τα προγράμματα και η ανάληψη δράση αναβάλλονται εβδομάδα τη βδομάδα. Όμω μαζί αυξάνονται και οι απαιτήσει μα και εμεί Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να οδηγήσουμε στο σωστό δρόμο. Δείξαμε ότι με πέντε πολιτικές ομάδες από όλες τις πλευρές και τις παρατάξεις του Κοινοβουλίου προτείνουμε λύσει. Το συνυπογράφουν μέλη χωρών από τη Ρουμανία μέχρι τη Γερμανία και από την Ιταλία μέχρι τι κατοχώρε, από την Ισπανία μέχρι το Βέλγιο. Αυτό αποδεικνύει ότι εμεί μπορούμε να υπερβούμε τι διαφορέ μα και να βρούμε λύσει που να κάνουν διαφορά, να έχουν πολιτικό νόημα και οικονομικό νόημα. Αυτό που προτείνουμε είναι ομόλογα και με τα ομόλογα αυτά μπορεί κανεί να χρηματοδοτήσει ένα σχέδιο ανάκαμψη και ένα ε, ταμείο α, ε, μετατροπή διαφοροποίηση τη ευρωπαϊκή οικονομία. Και αυτό είναι σημαντικό. Δεν θέλουμε να συνεχιστεί ό,τι γινόταν στο παρελθόν. Θέλουμε ίδιου πόρου και ίδιου πόρου που να καλύπτουν όχι μόνο του ντόπου, αλλά και την αποπληρωμή. Αυτό εννοούμε εμεί ε, πραγματική κοινή ανάληψη ε, και των ευθυνών. Και επίση θα πρέπει να κοιτάξουμε να υπάρχει μια πραγματική πράσινη συμφωνία. Εάν δούμε όλα τα προγράμματα από τα οποία θα πρέπει να περάσουν από το δημοκρατικό μα έλεγχο, θα πρέπει να σκεφτούμε και να θυμηθούμε τη Συμφωνία των Παρισίων, την ε, ισότητα των φύλων. Θα πρέπει να απευθυνθούμε στου ανθρώπου που έχουν χτυπηθεί και έχουν πληγεί ε, δρυμύτερα από την κρίση. Γιατί βρίσκονται σε συνθήκε φτώχεια, ε, γιατί είναι εργαζόμενοι καταναλωτέ και οικογένειε. Και τελευταίο επιχείρημα, λέμε ότι οι κανόνε για την κρατική βοήθεια πρέπει να ευθυγραμμιστούν παντού. Και εκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θυμηθείτε ότι παρατείνατε τι κρατικέ βοήθειε μέχρι το τέλο του Ετου χωρί καμία ε, προπόθεση. Πολύ κακό σημάδι, πολύ κακό μήνυμα. Θα πρέπει λοιπόν να συγκεντρώσουμε όλα τα κονδύλια που μπορούμε και να ενώσουμε και τι δυνάμει μα για να έχουμε μια ισχυρότερη ανανεωμένη οικονομία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Εκχάουτ. Για ένα λεπτό ο κύριο Φιντάντσα. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε καθήκον να πούμε την αλήθεια. Ε, πάρα πολλέ εταιρείε θα κλείσουν. Καταστροφή κοινωνική και είναι ένοχοι για την καθυστέρηση και βλέπουμε ότι υπόσχονται τρεις που δεν υπάρχουν οπότε ε, διστάζεται γιατί βλέπετε τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λίγα και αργά θα δοθούν Επίσης, όσον αφορά την αιρεσιμότητα του Ταμείου Διάσωσης, υπάρχουν πολλές σκιέ. Άρα θα πρέπει να γίνουν όλα με διαφάνεια, να σταματήσουν τα δάνεια επιδανείων. Έτσι ε, κατεστράφει η Ευρώπη. Θα πρέπει να βοηθήσουμε το εμπόριο, να σταματήσει η επιθετική φορολογία, ε, να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει ε, να κάνετε κάτι για τους γίγαντες ε, του ίντερνετ θα πρέπει να σεβαστούν τα ευρωπαϊκά στάνταρ, το περιβάλλον κλπ. Να βοηθηθούν επίσης φορολογικά οι ΜΜΕ, γιατί αυτοί πληρώνουν την ε, νύφη με καινούργια Ευρώπη. Ναι, μην επιμένετε στο να υπεραμείνεστε τη χθεσινής Ευρώπη του παρελθόντο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, συνάδελφε ε, Φιντάντσο. Κύριε Σομορζάκη, ένα μισή λεπτό. Merci. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, δεν μπορούμε σε αυτή τη συζήτηση να φέρνουμε ε, το αδιέξοδο σε σχέση με το Συνταγματικό Δικαστήριο, το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο, γιατί δεν είναι δυνατόν ε, ούτε εσείς ούτε εμείς να αποκαταστήσουμε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Επρόκειτο για μια απόφαση πάρα πολύ σοβαρή. Κανείς, κανεί λαό στην Ευρώπη δεν είναι δυνατόν να δεχθεί να αναλάβει τον ε, ρόλο ε, του να του υπαγορεύει ένα ξένο συνταγματικό δικαστήριο το τι ισχύει στην Ευρώπη. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε για να κάνουμε το επόμενο βήμα 27 αποφάσεις από 27 συνταγματικά δικαστήρια. Αυτό είναι η αρχή του τέλους της Ευρώπης, συνάδελφοι, η οποία χρειάζεται ένα μεγάλο σχέδιο για ανάκαμψη. Έτσι ε, θα πρέπει να στραφούμε προς την αρχή της συνοχής. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυθεντικά είναι ευρωπαϊκή. Αυτό χρειάζεται. Όχι, δεν χρειάζεται να έχουμε μια τράπεζα η οποία να είναι ε, προσκολλημένη και να, και να διευθύνεται από το Βερολίνο. Αυτό θα πρέπει να γίνει για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε το σχέδιο ανάκαμψης. Αυτή η απόφαση το περιορίζει το σχέδιο ανάκαμψης. Είναι απαράδεκτο. Ούτε η Άγγελα Μέρκελ ε, μπορεί να, να, να το δεχθεί. Θα πρέπει ξεκάθαρα να το πει. Άρα θα πρέπει το Συμβούλιο αύριο να αγνοήσει, να απορρίψει αυτή την απόφαση και να προχωρήσει με συνοχή και αλληλεγγύη ακριβώς όπως διατυπώνουμε στο κοινό μας ψήφισμα το οποίο και υποστηρίζω. Ευχαριστούμε κύριο Μαρζέ. Για ένα λεπτό ο κύριος Πεστεμόνη Καζαμάχο. Ευχαριστώ όλες τα γερμανικά, στα αγγλικά υπάρχει κίνδυνος. Κίνδυνος να σταματήσει να είναι χρήσιμη η Ευρωπαϊκή Ένωση αν δεν μπορέσει να προσφέρει κάποιες λύσεις. Οι λύσεις θα πρέπει να είναι και οικονομικές αλλά και κοινωνικές. Όταν υπάρχει γκρέμισμα της οικονομίας τότε θα πρέπει να κινητοποιούνται κάποιοι πόροι και αυτό να αποδώσει. Παρ' όλα αυτά, όταν έχουμε αποδυνάμωση των δικαιωμάτων και σύγνωσή τους, τότε ποιο πρέπει να την ήθει. Τα ανθρώπινα δικαιώματα απειλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερο σήμερα από ποτέ και ε, ακόμη έχουμε πολιτικούς κρατουμένους. Αυτοί θα πρέπει να απελευθερωθούν. άμεσα ο Ασάντζο αλλά και οι ε, Καταλανοί ηγέτε για την εξαρτησία οπότε επιβάλλεται να, ο Τζόρντι Κουσάρ και ο Τζόρντι Σάντσα να απελευθερωθούν, να αποφυλακιστούν. Υπάρχει κάποιο σχέδιο από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση για να σωθεί έτσι η δημοκρατία ε, εκεί που έχει καταπατηθεί σοβαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον συνάδελφο κύριο Πιτζεμόν Καζαμάχο και τώρα το έχουμε τον συνάδελφο τον κύριο Φέρπερ για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, όταν έχει πέσει το σπίτι στο κεφάλι, δεν ξεκινάμε από το να κοιτάμε τα χρώματα για τα κεραμίδια, ξεκινάμε από τον αρχιτέκτονα για να βάλουμε τα σωστά θεμέλια. Αυτό που μου λείπει από τη συζήτηση είναι μια απάντηση στην ερώτηση του ποια είναι η ευρωπαϊκή ημεραξία την οποία μπορούμε να δώσουμε. Πέρα από αυτά που έχουν ξεκινήσει να κάνουν δικαίω τα κράτη-μέλη, προκειμένου στην τελική ανάλυση να μην υπάρχει αντίφαση, αλλά να ταιριάζουν τελικά όλα αυτά τα κομμάτια. Αυτό θα πρέπει να είναι το πρώτο στο θέμα. Κατά δεύτερον, θα πρέπει να ασχοληθούμε με το ποια είναι τα σωστά εργαλεία, τα σωστά μέσα. Το λέω ευθύ εξ αρχή. Δεν ακούω κάτι καινούριο. Εδώ και πολλά χρόνια μιλάμε για τα πράγματα αυτά. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι με κάποιους ε, φορολογικούς, κάποιες φορολογικές διαφορές θα καταφέρουμε να λύσουμε τα προβλήματα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ε, μπορεί να αποτελέσει αυτό λοιπόν τη βάση τη σωστή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να έχουμε ρεαλιστική αντιμετώπιση. Και τρίτον, αγαπητοί συνάδελφοι, έχω την αίσθηση ότι και εδώ στο ψήφισμα το θέμα είναι πώς μπορούμε να δώσουμε όσο πιο γρήγορα, όσο πιο πολλά χρήματα γίνεται υπό ε, χωρίς όρους στα κρατημέλη. Δεν είναι και αυτό λύση, γιατί δεν μπορούμε να ανοίξουμε τους ασκούς του αιώλου. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν αύριο πώς θα αποφασίσουμε ένα σωστό χρονικό διάγραμμα για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ συνάδελφε Φέρμπερ και τώρα έχουμε την κυρία Καρτίδη Σαμπάλ Ρουμπιάλ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, η αλήθεια είναι ότι στις διαπραγματεύσεις για το ψήφισμα είχαμε πολλές δυσκολίες γιατί υπήρχαν πολλές πιθανότητες αποτυχίας αλλά τα καταφέραμε και θα πρέπει να ευχαριστήσω για την επικοδομητική στάση όλους με όσους κάνουμε διαπραγματεύσεις. Ο στόχος ήταν να σωθεί η αξιοπρέπεια της Ευρώπης αλλά να σωθούν και οι ζωές. Ε, είναι στο ψήφισμα σύντομο και αυτό πάντοτε ήταν δύσκολο να το κάνουμε εδώ σε αυτό το κοινοβούλιο αλλά τέλος πάντων θα πρέπει το Συμβουλίο να λάβει υπόψη ότι συμφωνήσαμε πέντε κόμματα. Ε, άρα θα πρέπει να τα συμφωνήσουν και οι του Συμβουλίου. Ε, ακούσαμε την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν θα πρέπει να φοβάστε να ζητείτε κινητοποίηση ε, ε κρατικών πόρων. Χρειαζόμαστε επομένω ένα στεγανό, θωρακισμένο ε, πλαίσιο δημοσιονομικό και θέλουμε επίσης μεγάλες ε, επενδύσεις κόντρα στο χρέος. Μιλάμε για αυτά τα δισεκατομμύρια για να μπορέσουμε να αλλάξουμε την κοινωνία αυτό το 2%, 2% του ΕΠ και έτσι να έχουμε ε, μια επανάσταση φορολογική που χρειάζεται και θα βεβαίω και σημαντικό είναι να γίνει αυτό πρέπει να γίνει αλλά να γίνει καλά άρα να, δώσουμε μια ευκαιρία σε αυτή την ελπίδα και να λάβουμε υπόψη ότι τα πράγματα επίγουν αλλά και τα πράγματα είναι και σοβαρά τώρα το μήνυμα προς τον κόσμο είναι ότι έχουμε επίγνωση της κρίσης και ξέρουμε πόσο άσχημα πήγαν τα πράγματα στην προηγούμενη κρίση, δεν θα πρέπει τα λάθη να επανεληφθούν και εμεί είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται, να σώσουμε τον κόσμο, γιατί τελικά περί αυτού πρόκειται. Σωτηρία ανθρώπων. Ευχαριστούμε κύριε Καρδιά Θραμπάλε Ρούμπιελ. Για δύο λεπτά ο συνάδελφος σε Ζουρνέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, συνάδελφοι. Πραγματικά δεν ικανοποιήθηκα μετά την παρουσίαση τη Πρόεδρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι ε, προτάσει που μα έκανε. Ε, τον περσμένο μήνα το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε με μεγάλη πλειοψηφία ένα ψήφισμα για την απόκρισή μα στην πανδημία COVID. Και αναλάβαμε τι ευθύνε μα. Ε, δείξαμε ότι η αλληλεγγύη θέλουμε να είναι βασική προπόθεση ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρίσκεται στο ύψο των περιστάσεων και των προκλήσεων και να βοηθήσει όλου του πολίτε ανεξαιρέτω. ανεξαιρέτως. Η αλληλεγγύη αυτή είναι μια απέτηση, απέτηση και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για την ποιότητα του ψηφίσματος αυτού, διότι το Ευρωκοινοβούλιο άκουσε τους ευρωπαϊκούς λαούς. Προσφέραμε λύσεις ε, έτοιμες, ε, κομμένες και ραμμένες για το Συμβούλιο και δεν τα άκουσα καν στην ομιλία της ε, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τις ιδέες που εμείς είχαμε συμπεριλάβει στο δικό μας το ψήφισμα. Πραγματικά, βάσει τις αρχές της αλληλεγγύης είχαμε συντάξει συντάξει το ψήφισμα αυτό και ε, αυτό μας είχε προσχολήσει, ήταν γνώμονάς μα. Το Συμβούλιο συμφώνησε και όλος ο κόσμος εδώ αναφέρει τον Σούμαν, τον ιδρυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως η αλληλεγγύη είναι μια αλληλεγγύη, είναι ένα θέμα ευρωπαϊκό βεβαίω, μια ευρωπαϊκή αξία, αλλά πρέπει να φαίνεται και στις πράξεις, στις πράξεις και στα γεγονότα. Και αυτό θα πρέπει να φανεί για τα κράτη που περισσότερο πλήγησαν από τον κορονοϊό. Ό,τι και αν λένε οι εθνικές αρχές, ε, εδώ πρέπει να σκεφτούμε τι λέμε. Ε, μεταφορές, ποσά, κονδύλια, τι πρόγραμμα ανάκαμψη, μια μετάβαση που να βρίσκεται στο ύψο των περιστάσεων με την Πράσινη Συμφωνία, τα κορονομόλογα, την αλληλεγγύη, νέοι ήδη πόροι. Μα δεν άκουσα κάτι. Δεν άκουσα πολλέ εξηγήσει και λεπτομέρειε για το τι θα γίνει σε σχέση με αυτού του νέου ίδιου πόρου. Πραγματικά λοιπόν ήθελα να πω στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πραγματικά δεν πρέπει τώρα να φοβάστε και το να μην σας κρατάνε τα γόνατά σας. Ε, το είδαμε από τους συναδέλφους μας ε, τους, στις, στα εθνικά κοινοβούλια και τις εθνικές ε, συνελεύσεις. ο κόσμος καταλαβαίνει ότι δεν θα είναι εύκολο, θα πρέπει να εργαστούμε σκληρά για να βρούμε λύσεις. Στο εμικύκλεμο αυτό βλέπουμε ότι η ιστορία, και το έχουμε ξαναδεί, είναι ένας κριτή χωρί ήκτο. Οι αδυναμίες και Πρόεδρος Διακόπτη, ευχαριστούμε κύριε Σεζουρνέ. Ο κύριος Κούς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι. Αυτό που μας έδειξε η κρίση πάνω απ' όλα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένας καλός διαχειριστής κρίσεων. Είδαμε ότι οι περιοχές που αντιμετωπίζαν μεγάλο πρόβλημα ε, περιορίστηκαν πολύ αργά με τα σύνορά τους να κλείνουν και είδαμε ότι χρειάζεται αλληλεγγύη ε, για να αντιμετωπιστεί το κλείσιμο των συνόρων και όσα προκάλεσε η κρίση. Εδώ βλέπουμε πόσε πολλέ είναι οι επιπλοκέ τη κρίση και ε, μιλάτε για γιγαντιά ποσά και ε, υποσχέσει. Εδώ οι προσδοκίε μα φαίνεται να φτάνουν στα ύψη και πραγματικά ε, φαίνεται να θέλετε να χρηματοδοτήσετε τα κράτη όχι 30% αλλά 100% ε, σε σχέση με το ΑΕΠ και το τίμημα που έχουν πληρώσει. Αυτό δεν μπορεί να είναι η λύση. Θα πρέπει ε, να σκεφτούμε μήπως δημιουργήσουμε περισσότερα χρέη και αυτομάτως αυτό επιβαρύνει τα παιδιά μας πολύ περισσότερο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που ανέφερε και η κυρία Φοντερ Λάιεν. Δηλαδή, εάν θέλουμε αυτή τη στιγμή να φορτώσουμε με χρέη τον οργανισμό των παιδιών μας για το μέλλον, α το σκεφτούμε. Τα ε, ομόλογα θα βοηθήσουν τα παιδιά μας να ξαναπάνε στο σχολείο. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε κύριε Κού και για ένα λεπτό ο κύριο Άντερσεν. Ευχαριστώ. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη κρίση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και οι Ευρωπαίοι ε, αγωνίζονται για να ζήσουν, να χάνουν τι δουλειέ τους, αρρωσταίνουν. Ο κορονοϊός δεν του πλήττει όλου με τον ίδιο τρόπο. Αυτοί που πλήττονται πιο πολύ είναι οι αδύναμοι και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δικαστή από την κρίση θα χάσουν όλοι και όλοι θα αποδυναμωθούν. Θα πρέπει να δράσουμε τολμηρά λοιπόν. Θα πρέπει να δείξουμε εδώ στο Κοινοβούλιο ότι με ευρεία υποστήριξη μπορούμε να ψηφίσουμε ένα ψήφισμα. Ζητάμε λοιπόν ένα σχέδιο δύο Δεν πρέπει να επαναλάβουμε τα λάθη της Ευρώπη κρίσης με τα προγράμματα λιτότητα. Αντί για αντιδικοποίηση, θα πρέπει να επενδύσουμε στο σύστημα υγειονομική περίθαλψη. Αντί να προωθήσουμε αυτούς που ρηπαίνουν θα πρέπει να έχουμε μια πολιτική η οποία θα είναι δική προς το κλίμα και γι' αυτό ζητώ από την ε, κυρία Φοντερ Λάιεν να βρείτε μια λύση όχι όμως μια λύση η οποία θα δώσει χρήματα για δύο χρόνια και μετά θα προχωρήσει σε περικοπές. Δεν θα λύσουμε έτσι την κρίση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα λεπτό ο συνάδελφος κ. Σούγκα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι. το δράμα της πανδημίας αυτής παραδόξως ενδεχομένως να μας προχωρήσει, να μας ε, προχωρήσει πιο μπροστά. Να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τι πάει στραβά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία να καταπολεμήσουμε την φοροδιαφυγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει επίση να φροντίσουμε το θέμα των κρατικών επιδοτήσεων. Έχουμε τεράστιε διαφορέ μεταξύ των κρατών και αυτό βλάπτει την ε, κοινή αγορά την ενιαία αγορά. Θα πρέπει να καταργήσουμε τους φορολογικούς παραδείσους. Και οποιασδήποτε επιστροφές, γιατί μιλάμε για μεγάλη πηγή χρημάτων, την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να αξιοποιήσουμε. Έχουμε την ευκαιρία επίσης να δώσουμε δάνεια και επιχορηγήσεις, αλλά δεν μπορούμε να ξεχνάμε και την συνοχή από τον τομέα των μεταφορών, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τη γεωργία. Αυτό αποτελεί τη βάση για την μελλοντική επιτυχία και την ανάκαμψη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα για ένα λεπτό η κυρία Κουντουρά. Κύριε Πρόεδρε, ο Σούμαν πριν από 70 χρόνια είπε ότι η Ευρώπη δεν θα δημιουργηθεί με τη μία ούτε σε ένα συνολικό οικοδόμημα. Θα διαμορφωθεί μέσα από συγκεκριμένα επιτεύγματα που θα δημιουργήσουν πρώτα μια πραγματική αλληλεγγύη. τα λόγια του λοιπόν είναι πιο επίκαιρα από ποτέ σήμερα. είμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και επιβάλλεται να διαλέξουμε το δρόμο της αλληλεγγύης γιατί κινδυνεύουμε να χάσουμε ό,τι χτίσαμε τα τελευταία 70 χρόνια. αυτό που βιώνουμε σήμερα στην ευρώπη είναι εθνικά συμφέροντα εθνική επιβολή όχι με πόλεμο αλλά μέσω οικονομικής δύναμης. ο νόμος της απόλυτης υπερίσχυσης του πιο δυνατού. πρέπει να μπει ένα τέλος και η απάντησή μας σε αυτή την κρίση πρέπει να είναι ένα γενναίο σχέδιο ανάκαμψης πραγματική στήριξη αυτών που το έχουν ανάγκη με επιδοτήσεις και όχι με νέα χρέη νέα εργαλεία για ίδιους πόρους της ευρωπαϊκής ένωσης ώστε να μην αποφασίζει ο πιο πλούσιος για όλους τους υπόλοιπους και τέλος πραγματική δημοκρατία με ισότιμη συμμετοχή του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου στη λήψη αποφάσεων για το σχέδιο της ανάκαμψης. ευχαριστώ πολύ. κυρία ε, Μπεγίν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συνάδελφοι, είναι πάρα πολύ σημαντικό το σχέδιο ανάκαμψη για να μπορέσουμε να έχουμε ανασυγκρότηση τη οικονομία. Οπότε θα πρέπει έτσι να έχουμε κάποια αξιόγραφα να χρηματοδοτήσουμε ε, την υπόθεση από τι και έχουμε 2,5 δι ευρώ προ τούτο. Αλλά θα πρέπει όμω πάνω απ' όλα να μπορέσουμε ε, να ε, βοηθήσουμε και με πόρου και όχι μόνο με δάνεια. Ε, και έχουμε αυτούς τους ε, φόρους πάνω στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, στις μεγάλες εταιρείες. Άρα αυτό θα πρέπει να γίνει άμεσα χωρίς να περιμένουμε να τελειώσουν μακρές διαπραγματεύσεις και οπότε θα πρέπει και αυτό το επταετές σχέδιο να αλλάξει το ΠΔΠ να προσαρμοστεί στην κατάσταση δεν θέλουμε να υπάρχει ε, κάτι το οποίο είναι προσαρμοσμένο στην πανδημία και έτσι θέλουμε να δούμε πώς προσωρινά θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτές τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο ε, να αυξηθεί η συγχρηματοδότηση να πάει στο 90-95% εκεί που χρειάζεται και ε, πρόεδρε ε, συναδελφοί μας διδάσκει στο της Ευρώπης ότι κάθε κρίση μπορεί να γίνει μια ευκαιρία αν έχουμε τη σωστή διαχείριση και σήμερα 70 χρόνια μετά την διακήρυξη του Σούμαν έχουμε την ε, ευκαιρία, έχουμε την ε, ευθύνη και έχουμε και την τιμή να μπορέσουμε να δώσουμε μια απάντηση που δεν θα έχει προηγούμενο προς τον κόσμο και επομένως με λίγα λόγια να ενώσουμε την Ευρώπη να δείξουμε στον κόσμο τι μπορούμε να καταφέρουμε όλοι μαζί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Μπεγκίν. Για 1,5 λεπτό η κυρία Νίμπλερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής, συνάδελφοι. Ο κορονοϊός και οι επιπτώσεις του θα είναι μια ιστορική πρόκληση που βεβαίως θα επηρεάσει και τον πολιτή μας προπολογισμό και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλα εγκαίρως. Θέλω να κάνω τις εξής παρατηρήσεις. Πρώτον, λόγω της κρίσης θα πρέπει να μην ξεχάσουμε ότι υπάρχει και ένα απότερο μέλλον μετά την περίοδο του κορονοϊού. Οι προτεραιότητε μα στην έρευνα και την ανάπτυξη, στην ψηφιοποίηση, σε ε, μια ε, οικονομικά ε, σωστά οικοδομημένη πράσινη συμφωνία, θα πρέπει να είναι στοιχεία που θα τα αντιμετωπίσουμε και στην περίοδο μετά τον κορονοϊό. Επίσης, θα πρέπει να μην ε, προβλέψουμε τις απαραίτητες δυνατότητες για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό μόνο από τις συνεισφορές των κρατών μελών. Θα πρέπει να υπάρξει και πραγματική στήριξη από την οικονομία. Και βεβαίως χρειάζεται και διαφάνεια. Χρειάζεται δημοκρατική ε, αλληλεγγύη και αυτό και στην ε, συνεισφορά την οικονομική μας για την αντιμετώπιση της κρίσης. Καταλαβαίνω ότι χρειάζεται έγκαιρη αντιμετώπιση τώρα και με τα ευελικτότερα μέσα. Όμως θα πρέπει να σκεφτούμε στις δεδομένες σημερινές συνθήκες ότι τώρα, ε, όσοι βρισκόμαστε εδώ, ε, έχουμε και την ευθύνη να λάβουμε αποφάσεις δημοκρατικές και που να τους εκπροσωπεί όλους και βεβαίως τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουν τα κράτη να είναι και ανάλογα με τις δυνατότητές τους. Αυτό το ζητώ και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από όλους τους συγκεντρωμένους συναδέλφους του Ευρωκοινοβουλίου. Ευχαριστούμε κυρία Νίμπλερ. Για 1,5 λεπτό ο συνάδελφος Φερνάντες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Στι 6 Μαου όφιλε να παρουσιάσει την πρόταση και έτσι να προβλέπετε το νέο πιδελταπή και να μπορέσουμε εδώ να έχουμε την πρόταση για το σχέδιο ανάκαμψης. Δεν το έκανε και σήμερα ε, είχε κάποιες προτάσεις οπότε ε, γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια οριστική πρόταση μέχρι τέλος του μηνός πρέπει να σας πω ότι αυτό είναι απαράδεκτο και είναι απαράδεκτο οπότε το Κοινοβούλιο συμφωνεί ότι πρέπει να υπάρχει ε, αυτό το ψήφισμα. Ομόφωνα το κατεβάσαμε. Χρειάζεται απόκριση αλληλέγγυα, χρειάζεται άμεση για την κρίση και επίσης να σχεδιαστεί μια στρατηγική ανάκαμψης τουλάχιστον δύο ε, δις και με πόρους που να πάνε στην ε, πραγματική οικονομία με άμεσες πληρωμές. Τι σας λέμε και το τονίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα ε, έπρεπε να, μην, ε, να κάνει αυτό το οποίο έκανε, δηλαδή να μας έχει κάποιου προπλασιαστέ που είναι φαντάσματα. Μα αυτό είναι πάρα πολύ κακό, όχι μόνο για την Κομισιόν, αλλά για το σύνολο του ευρωπαϊκού οράματο δεν θα πρέπει να περιμένετε το Συμβούλιο ούτως ώστε να κατεβάσετε μια πρόταση προς εμάς. Εμείς ε, ομόφωνα είπαμε ότι είμαστε δίπλα σας για να πάμε στο Συμβούλιο να διαπραγματευτούμε. Αυτό είναι το ε, συμπέρασμα από την προηγούμενη θητεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, συνάδελφε Φερνάντες. Για δύο λεπτά ο κύριος Φερχόφστατ. Πρόεδρε, να σας πω ότι μετά την ε, ε, παρέμβαση της κυρίας Φόντερ Λάιεν βλέπω να συνεχίζονται τα πράγματα όπως τα ξέραμε και πριν. Πραγματικά ελπίζω να πέφτω έξω. Αλλά Είδα και τα πρώτα έγγραφα που κυκλοφορήσαν στο επίπεδο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πραγματικά είναι business as usual. Ε, είναι ό,τι γινόταν συνήθω. Μια νέα συσκευασία βρήκανε, πολύ ωραίε διατυπώσει και μετά κάτι πολλαπλασιαστέ. Πολλαπλασιαστέ που Πού θα του βρει να του χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με συντελεστή 45 ακόμα και ο Ισού στην καινή διαθήκη. Δεν ήταν εύκολο να τα πολλαπλασιάσει τα ψωμιά και το κρασί επί 45. Ε, δεν το κατάφερε για τα ψάρια και το ψωμί. Ε, η Ευρωπαϊκή λοιπόν εδώ Επιτροπή Όπω συνήθω με τα γραφειοκρατία τη, με τη διοίκησή τη και τη διοικητική διοργάνωση, έτσι δουλεύει. Το εξήγησε η κυρία Φοντερ Λάιν. Θα τα καταφέρουμε. Θα ε, υψώσουμε λίγο τώρα το τόριο και θα ζητήσουμε περισσότερε εγγυήσει από τα, κρατη... τα μελη Μα αυτό ακριβώ δεν πρέπει να κάνουμε. Όλα τα κράτη-μέλη μα αυτή τη στιγμή θα έχουν έλλειμμα και χρέη. Δεν μπορούμε να αυξήσουμε τώρα τι εθνικέ ενισφορέ των κρατών μελών, που ζητάνε και να ζητήσουμε και περισσότερε εγγυήσει στο μέλλον. Ε, αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να υπάρξει ένα νέο κεφάλαιο. Ήδη πόροι, νέοι διπόροι. Δεν είναι καμία επιστημονική φαντασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα βασιζόταν στου ίδιου πόρου. Το φόρο προστιθέμενη αξία, ειδικού τελωνικού φόρου, ψηφιακό φόρο έχουμε προτείνει εμεί και άλλου φόρου κατά τη ρήπανση. Είναι λόγω τη συζήτηση που είχε ε, γίνει με αφορμή την Μάργαρετ Θάτσερ και τότε είχαμε προσπαθήσει να σταματήσουμε τα δημοκρατικά δημοσιονομικά με τον τρόπο που γινόντουσαν προηγουμένω. Ε, έτσι τα σταματήσαμε τότε και τώρα πρέπει να πάψουμε. Πρέπει να υπάρξει πραγματική χρηματοδότηση για αυτή την ένωση. Το πρόβλημα λοιπόν κύριε Πρόεδρε δεν είναι πού θα γίνουν οι δαπάνες. Το πρόβλημα είναι πού θα βρούμε το χρήμα. Και κύριε Σεφτκοβίτς αύριο στη συνάντηση τη Επιτροπή, αυτό ζητάω να σκεφτείτε. Νέες λύσεις να ζητήσετε και αυτό που σας προτείναμε και εμεί στο ψήφισμά μας. Ευχαριστούμε συνάδελφε Φερχόφστατ. Και τώρα για ένα, λεπτό ε, ο συνάδελφος Ρινάλντι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πραγματικά αυτά που είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση ως συνθήματα για την αντιμετώπιση της ε, πανδημίας είναι τελικά μόνο ένα αυτό που φαίνεται να καταφέραμε το όρος έτε και μη. Ε, δηλαδή μόνο η ΕΣΜΑ είναι ο μηχανισμός ε, της σταθεροποίησης ήταν κάτι που θα μας προσέφερε υποτίθεται κάτι αλλά και το Ταμείο της Ανάκαμψης δεν φαίνεται να μας χρησιμεύει σε τίποτα σήμερα. Είναι χρηματοδοτήσεις με μηδενικούς ε, τόκους και θα παίρνει υποτίθεται ε, κάποιος τις συνεισφορές των ε, κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως τους ξέραμε σήμερα και τους αυξάνει με ένα πολλαπλασιαστή ή θα έχουν απαλλάξει στο μέλλον. Αυτά που μας είπε η κυρία Γιούροβα για να λειτουργεί το 2021 είναι περισσιόδοξα. Πώς θα λειτουργεί και πώς θα υπάρχει μόχλευση από το πρόγραμμα Juncker του 2014, το περίφημο εκείνο 300 ευρώ που ποτέ δεν είδε το φως της ημέρας. Εδώ λοιπόν ακριβώς αυτό θα είναι ένα αντίγραφο του προγράμματος στρατηγικών επενδύσεων, τίποτε παραπάνω. Θα χάσουμε πολύτιμο χρόνο αναβάλλοντας αποφάσεις και εντωμεταξύ επιχειρήσεις και κυρίως Ευρωπαίοι πολίτες θα έχουν γονατίσει. Θα έχουν γονατίσει και θα ε, έχουμε περάσει από μια κατάσταση παρόμοια με πόλεμο, αλλά θα συνεχίσουμε να ψάχνουμε εμεί με πείσμα τα κατάλληλα εργαλεία βάσει των συνθηκών και τη γραφειοκρατία, λε και βρισκόμαστε σε καιρού ειρήνη. Επιτέλου πρέπει να έχουμε το δόλο και τη θάρη, να λάβουμε αποφάσει εξαιρετικέ και έκτακτε, όπω την εντολή τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που πρέπει να αλλάξει, πρέπει να δράσουμε. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφε Ρινάλτη. Και τώρα ο συνάδελφο ο κ. Κορμό. Έχει το λόγο για ένα λεπτό. Αγαπητοί φίλοι, το ξέρουμε όλοι ότι το θέμα τη χρηματοδότηση ποτέ δεν είναι θέμα ε, οικονομικό, είναι και πολιτικό θέμα. Και η κρίση αυτή λοιπόν μας φέρνει ε, αντιμέτωπο σε αυτό το βασικό θέμα. Εμείς είμαστε λοιπόν αυτοί που θα πρέπει να προσπαθήσουμε για την ευρωπαϊκή αυτή κρίση. Χωρίς τους ίδιου πόρους αυτό που θα κρυθεί. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν γιατί η Ευρώπη δεν ε, μπορεί να χάσει ένα οικονομικό έτος. Θα πρέπει να δούμε τους ιδίους πόρους στην πραγματικότητα. Θα πρέπει να έχουμε τους πολιτικούς πόρους για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση, την περιβαλλοντική, την οικονομική, την κοινωνική. Χρειαζόμαστε ίδιους πόρους για να ε, χρηματοδοτήσουμε ένα σχέδιο ανάκαμψης ε, και σε ό,τι αφορά τους πόρους, σε ό,τι αφορά τον φόρο συναλλαγών κτλ θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να φροντίσει να υπάρξει μια δίκαιη μετάβαση στο παγκόσμιο προσκήνιο. Χωρίς ιδίους πόρους δεν θα μπορέσει να το πειράξει αυτό. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Κορμά και τώρα για ένα λεπτό το λόγο έχει ο κύριος Τζαμπάσκι. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο και τους συναδέλφους. Είναι σαφές ότι θα χρειαστεί μετά το γενεζικό ιό μία α, μεταρρύθμιση του οικονομικού πλαισίου. Αλλά αυτό δεν θα πρέπει να είναι εις βάρος του φορολογούμενου. Ακούμε διάφορες περίεργες ιδέες για νέους φόρους. Μεταδεχόμαστε αυτά. Σκοπός θα πρέπει να είναι να μειωθεί η γραφειοκρατία σε διεθνές επίπεδο. Υπάρχουν πολλές παράλογες ιδέες σε αυτή φορά το πράσινο σύμφωνο, το πακέτο κινητικότητας. Όλα αυτά θα καταστρέψουν τις θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη. Το πράσινο σύμφωνο είναι προς το συμφέρον της Κίνας. Η βιομηχανία θα συνεχίσει να μετακαταστάται στην Κίνα. Αυτό πρέπει να το καταπολεμήσουμε. Οι πολίτες θα πρέπει να βλέπουν διευκολύνσεις ε, αντί να εργαζόμαστε επί περίεργων ιδεών όπως το Πράσινο Σύμφωνο. Τέλος, να ε, ζητήσουμε ευθύνε από την Κίνα για την διάδοση του ιού αυτού. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, συνάδελφε Τσαμπάσκη, για ένα λεπτό, ο κ. Μποτέγκα. Ευχαριστώ πολύ. Μιλάμε για επενδύσεις και σε κάποια φάση όμω κάποιο θα πρέπει να τα πληρώσει όλα αυτά. Και εκεί θα πρέπει να δώσουμε προσοχή. Βρήκα λεφτά όμω στην Ευρώπη. Δεν θα ζητήσουμε καν από τον Γερμανό εργαζόμενο να πληρώσει τον Ιταλό εκατομμυρίουχο που θα βάλει τα χρήματά του στο φορολογικό παράδεισο που είναι η Ολλανδία. Όχι, θα δούμε. Στη Forbes, ο Λίστα, Μπερναναρνό, Λουί Βιτών, 70 δις ε, ευρώ. Δεν ξέρετε αν τα κάνει. Ορτέγκα από την, τα καταστήματα Ζάρα, 50 δις. Τι να τα κάνει, τι να τα κάνει. Χέρμαν Τίλερ, ο δισεκατομμυριούχος χώρο τη Λουφτχάντζα, ο οποίο σήμερα θέλει να πωλήσει ε, τόσου πολλούς ε, στο Βέλγιο δισεκατομμυρίουχο κι αυτό. Έχουμε χρήματα. Α βάλουμε λοιπόν ε, ένα φόρο στου δισεκατομμυρίουχου αυτού. Έχουμε χρήματα. Οι εκατομμυρίουχοι να πληρώσουν. Αυτό θα έχει τη διαφορά. Τι περιμένουμε λοιπόν. Ευχαριστώ. Για ένα μισή λεπτό τώρα. Κομίνιο Λιβέρες. Euh, euh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτή η κρίση έχει φέρει τριγμού στα θεμέλια τη συζήτηση για το ΠΔΠ που ξεκίνησε εδώ και μήνες. Ε, τώρα, ε, το θέμα δεν είναι ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόκειται για του ίδιου πόρου. Εκεί θα στηριχτεί το σχέδιο ανάκαμψη, τα ευρωομόλογα, τα οποία επίση πρόκειται αυτό το ταμείο, αυτό το σχέδιο να το υποστηρίξουν. Άρα έχουμε αυτό το 2% του ΑΕΠ που θα μας βοηθήσει να κάνουμε αυτό το άλμα και θα πρέπει να δούμε πώς θα ε, έχουμε 1% περιθώριο, αλλά βέβαια όλα αυτά είναι πενταροδεκάρες λόγω της κατάστασης. Επομένως, η συζήτηση είναι ολοένα και πιο ε, σημαντική, δηλαδή ε, θα πρέπει να έχουμε διαφορετικούς ίδιους πόρους για να τα καταφέρουμε. Το είπαν αυτό πολλοί συνάδελφοι σήμερα. Δεν ήρθε η ώρα να έχουμε κάποιο είδους φόρους, φόρους στα πλαίσια ε, των δασμών στα πλαίσια των ιδίων πόρων. Ε, κάποιους φορούς να βοηθούν το Green Deal ε, να σταματήσουν οι ανισότητες και επίσης να δούμε το ότι υπάρχουν άδικοι φόροι σε πολλές χώρες. Επομένως, μας έδωσε την αφορμή για τέτοια κουβέντα η πανδημία. Να βρούμε ένα πραγματικά ευρωπαϊκό φορολογικό σύστημα. Να είναι το Κοινοβούλιο και όχι το Συμβούλιο πρωτοπόρο στη συζήτηση ή τώρα ή ποτέ. Ευχαριστούμε κύριε Κομίνιο Ολιγέρες. Τώρα για ένα λεπτό ο κύριος Ντέλη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η κρίση του κορονοϊού έδειξε ότι τώρα αυτό που θα είναι καθοριστική σημασία για την οικονομική ανάκαμψη στην περίοδο μετά την κρίση είναι να έχουμε ένα προπολογισμό ικανό και φιλόδοξο. Μετά την κρίση θα χρειαστεί ένα τέτοιο πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δεν θα ε, αντλεί από τι παραδοσιακέ ευρωπαϊκέ πολιτικέ. Η πολιτική συνοχή και η γεωργική πολιτική λόγω χάρη πρέπει να ενισχυθούν. Η πολιτική συνοχή είναι το σημαντικότερο εργαλείο χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση και από αυτό κερδίζουν όλα τα κρατη Πρέπει λοιπόν να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει η απαραίτητη ευελιξία και αποτελεσματικότητα στη χρήση αυτών των κονδυλίων. Εγώ βεβαίω ω Ούγκρο βουλευτή θα δώσω ιδιαίτερη προσοχή στην ίση κατανομή των κονδυλίων και στην πολιτική της συνοχής πρέπει να πούμε ότι σίγουρα έχουμε δει να καλύπτει το χάσμα ανισότητα μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. 5% ήταν η αύξηση του εισοδήματο στην Ουγγαρία για πολλού επί σειρά ετών χάρη στην πολιτική συνοχή. Έχουν δημιουργηθεί θέσει εργασία. Ελπίζω λοιπόν ότι οι νέε μα λύσει δεν θα θέσουν ένα αμφιβόλο αυτά που ήδη έχουμε πετύχει. Δεν θέλουμε ε, να πληγεί η πολιτική συνοχή ε, από αυτά τα νέα προγράμματα. Θα πρέπει όλα τα τη μελη βεβαίω να υποστηριχθούν ανάλογα με τι ανάγκε του και την αξία του. Ευχαριστούμε, συνάδελφε Ντέιλε, για ένα λεπτό. Ο συνάδελφο Τάνγκ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και μετά ε, την απομόνωση, το lockdown, ε, πρέπει να α, ε, βγούμε. Πώς τρεις τρόπους. Καταρχάς ανακάψει για όλους. Θα πρέπει να δούμε ότι μια, ένα πρόβλημα για μια χώρα είναι πρόβλημα για όλους. Δεν έχουμε. Λοιπόν, δεν είναι στιγμή να κατηγορήσουμε με τους ΔΕΣ. Θα πρέπει όλοι να βγούμε από την κρίση. Και εδώ θα μας εξυπηρετήσει το ψήφισμα κατά δεύτερον. Θέλουμε να μπει στο στην πρώτη θέση το περιβάλλον. Θα πρέπει λοιπόν κάθε επένδυση να μην βλάψει το περιβάλλον και τον κόσμο. Κατά τρίτον, θα πρέπει να μπει ένα τέλος ε, στην ε, προδιαφυγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, οι μεγάλες επιχειρήσεις να συμβάλλουν ε, στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Αυτή είναι τρεις επιλογές για να καταφέρουμε να βγούμε με τον καλύτερο τρόπο από την κρίση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα ο κύριος Κέρνερ για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι σημαντικό νομίζω στην κρίση αυτή να δώσουμε μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση. Και γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουμε ένα ισχυρό πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και να προσέξουμε να υπάρχει ενίσχυση στο που, το που τα προγράμματα των προγραμμάτων αυτών που χρειάζεται να μην πάνε όλα στην ανάκαμψη. Πώς θα ξοδέψουμε τα χρήματα αυτά. Πού θέλουμε να δαπανηθούν τα χρήματα αυτά, γιατί είναι τεράστια πόσα. Θέλουμε να αναγνωρίσουμε την ε, ψηφιοποίηση. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δοθεί μια έμφαση στην ψηφιοποίηση προκειμένου να είμαστε ανταγωνιστικοί μετά την κρίση. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα μας βοηθήσουν οι φόροι. Σε αυτή την ε, κρίση θεωρώ ότι είναι δηλητήριο αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ένας ψηφιακός φόρος ε, σημαίνει ότι οι Αμερικανοί και ο Τραμπ θα ξεκινήσουν να τα διαλύουν όλα. Δεν θα μας βοηθήσουν αυτά για να εξέλθουμε από την κρίση. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι χρειαζόμαστε έναν προπολογισμό που θα επενδύσει στο μέλλον και που θα δώσει χρήματα σε αυτούς που α, σέβονται το κράτος δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα ο κύριος Μαριάννη για ένα λεπτό. Ο μήνα του Απριλίου είναι ένα μήνα δακρύων. Στη Γαλλία, στην Ελσατία, στην Ισπανία και στη Λομπαρδία οι Ευρωπαίοι όλοι μιλούσαν την διαφωνή και έγιναν δάκρυα. Και περιμέναμε να τοποθετηθεί η Ευρώπη. Στι 23 Απριλίου μα είπε ο κ. Μισελ για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι είμαστε ευτυχεί για το φιλοπορία, για την ανάκαμψη. Μια δήλωση που φαίνεται να είναι πραγματικά άτυχη στη στιγμή που η ανεργία, η δυστυχία, η τεράστια φτώχεια δεν φαίνεται να αφήνουν ευτυχία τυχή ε, ελπίδε για την ανάκαμψη. 500 δι είναι ελάχιστα για την ανάκαμψη και βεβαίω όπω είπαμε και οι προηγούμενοι ομιλητέ ε, μα έχει αφήσει πάντοτε να περιμένουμε ένα πιο συγκεκριμένο και λεπτομερέ πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η γραφειοκρατία ε, και η καθυστέρηση, το πόσο χρόνο τριβεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σίγουρα για κάποιου είναι ευχάριστο. Όμω δεν βλέπουμε πού θα είναι το νέο χρήμα, πού θα είναι αυτό το νέο ταμείο που θα έχει την απαραίτητη ευελιξία και θα μπορέσει ε, να απελευθερώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση από τα ίδια στενόμυαλα κεφάλια που έκλεισαν την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το πνεύμα ε, γραφειοκρατία. Ευχαριστούμε για ένα λεπτό ο κύριος Χάν, η κυρία Χάν, συνάδελφοι, με την ανάκαμψη μετά την, Ευρωπαϊκή, μετά την κρίση του κορονοϊού. Δεν χρειάζονται μόνο χρήματα, αλλά θα πρέπει να δούμε τι δομέ που υπήρχαν από το παρελθόν. Ούτε με την κρίση του κορονοϊού, ούτε με την κλιματική κρίση φαίνεται ότι έχουμε την, ε, το, τη λήψη των μοιρών αποφάσεων. Χρειαζόμαστε ένα ε, νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και να θέσουμε στα θεμέλια την Πράσινη Συμφωνία. Για να υπάρξει ανοικοδόμηση της οικονομίας μας. Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε στις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίε ή τι αεροπορικές εταιρείε, αλλά θα πρέπει να δούμε και τι πολλέ τις εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίε επιχειρήσεις που είναι ο κρογόνες λέω των ε, τη οικονομία μα και τη ενεργειακή απόδοση. Χρειαζόμαστε μια αποβιομηχανοποίηση ε, με τέτοιο τρόπο που να επιτρέπει την κάλυψη και των εργασιακών και των κοινωνικών αναγκών. Θα πρέπει να υπάρχει και ένα ταμείο δίκαιη μετάβαση. Τώρα είναι μεγάλη ευκαιρία να θέσουμε τι σωστέ προποθέσει και τα θεμέλια για μια ε, ισχυρή, αηφόρο και ε, σταθερή οικονομική ανάπτυξη τη Ευρώπη. Τότε θα έχουμε πάρει ε, ω καλή ευκαιρία την κρίση. Ευχαριστούμε, συνάδελφε Χάν. Για ένα λεπτό, ο συνάδελφο Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, τα εξή θέλω να σας πω. Πρώτα-πρώτα, να σας τονίσω ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η πολιτική συνοχή. Είναι ο πιο αποτελεσματικό τρόπος να γεφυρώσουμε τις διαφορές όσον αφορά την ανάπτυξη Επίσης, η κοινή γεωργική πολιτική, οι γεωργοί μας, μας εξασφάλισαν την διατροφή κατά την πανδημία, οπότε θα πρέπει να συνεχιστεί η κοινή ε, γεωργική πολιτική και πρέπει να τους ενισχύσουμε γιατί έχουν τώρα ευξημένες υποχρεώσεις οι γεωργοί μας. Επίσης, αυτό το σχέδιο ανάκαμψης θα πρέπει να στηριχθεί σε κάποιες χωριές, και όχι σε ε, δάνεια. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλέ χώρε, ιδίω στον Νότο, που δεν αντέχουν περισσότερο χρέο. Κατά τέταρτο λόγο, θα πρέπει να ε, πούμε ότι είναι θετικά τα όσα είπε η Ευρωπαϊκή Τροπή για τι κρατικέ ενισχύσει. Όμως ε, αυτή η βοήθεια είναι πολύ διαφοροποιημένη, φέρνει στρεβλώσεις, είναι πρόβλημα για την κοινή αγορά. Σας ευχαριστώ. Μονσεράτ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι. Πριν από 70 χρόνια ο Σούμαν ξεκίνησε μετά από αυτόν τον σκληρό πόλεμο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα όμως ο εχθρός είναι η πανδημία, αργήσαμε, ο καθένας έκανε τα δικά του, αλλά έτσι μάθαμε, τώρα είμαστε εδώ ενωμένοι. Ξεπεράσαμε ιδεολογικά σύνορα και γραφικά σύνορα φτάσαμε στο να εγκρίνουμε αυτό το κείμενο που περιμένει ο κόσμος από εμά. Να είμαστε ενωμένοι και όχι διερημερινά το ε, μήνυμα προς Κομισιόν και Συμβούλιο. Υπάρχει η Οδύνη για χιλιάδες ε, απολειών, για εκατομμύρια ανέργων, κλείσιμο ΜΜΕ. Ε, πρέπει να παλέψουμε για την ανάπτυξη στην Ευρώπη και άρα να μην ξεχνούμε ότι αυτό το κείμενο θα πρέπει να ωφελήσει όλους τους Ευρωπαίους. Οπότε θα πρέπει να δείξουμε υπευθυνότητα όσον αφορά την αξιοποίηση των πόρων και έτσι να μπορέσουμε να προωθήσουμε, να, να τον κόσμο να προχωρήσει, να αφήσουμε κανέναν απ' έξω. Να έχουμε κάποιες προσαρμοσμένες πολιτικές ε, ατζέντε και έτσι να, η Ευρώπη να αντιμετωπίσει τη νέα πραγματικότητα του 21ου αιώνα. Νομίζω ότι αυτό ε, ήταν ε, επιτάχυνση ε, ήταν ένα κίνητρο το COVID. Τουρισμός, πράσινη οικονομία, θωράκιση συστήματος υγείας και να μην ξεχνούμε ποτέ ελευθερία, ισότητα, αλληλεγγύη. Θα πρέπει να ξαναβρούμε εκείνη την υπερηφάνεια ότι ανοίγουμε στην Ευρώπη που μας προσέχει, μας στέλνει στην ανάπτυξη. Το ε, διετράνωσε ο Σούμαν και αυτό θα πρέπει να τηρήσουμε και σήμερα. Ένα λεπτό Μπενιφέη. Αυτή τη φορά δεν έχετε μικρόφωνο κύριε Μπενιφέη. Αυτή τη φορά δεν έχει μικρόφωνο κύριε Μπενιφέη. Το μικρόφωνο σας του λέει ο πρόεδρος. Τώρα, τώρα το ανάψατε. Αυτή τη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν κόλλησε για, χρόνια αντέδρασε γρήγορα, βοήθησε τα κρατημέλη, ούτω ώστε να δαπανηθούν ό,τι χρειάζεται για να νικήσουμε ε, την πανδημία. Χρειάζεται ακόμα ένα βήμα. Αυτό το σχεδίο ανάκαμψη με τα κορονοομόλογα να είναι ξεκάθαρο το μήνυμα για όλο τον κόσμο ότι υπάρχει η Ευρώπη. Θέλει να έχει συνοχή, ελευθερία, ενωμένη, προσιλωμένη για πολιτικές ελευθερίες, και για το κοινωνικό ευρωπαϊκό πρότυπο. Ε, να τα κάνουμε αυτά να προκαταλάβουμε τις εξελίξεις. Έχουμε ε, ε, να δώσουμε εκατομμύρια εκατομμυρίων. Δεν είναι θέμα τη αλληλεγγύη μόνο, είναι το κοινό μα μέλλον. Διότι κανεί κανείς δεν μπορεί να ευημερήσει εάν καταρρεύσει η κοινή αγορά, εάν δεν υπάρχουν λυσίδε αξιών. Δεν θα πρέπει αλλού να δοθούν ενισχύσεις και αλλού να μην δοθούν. Άρα θα πρέπει να βρούμε το σωστό δρόμο, να μην προδώσουμε τις βασικές αρχές μας που είναι το θεμέλιο της Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε συνάδελφε Μπενιφέη. Για ένα λεπτό ο συνάδελφος Σαστέλ. Πρόεδρε, συνάδελφοι, το Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να είναι ένας από τους πρωταγωνιστές της οικονομικής ανάπτυξης και των δημοτεύσεων του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου. Θέλουμε να είναι ε, σαφείς οι αποφάσεις μας σε ένα ε, πλαίσιο οικονομικής κρίσης. Θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι, αλληλέγγυοι και αξιόπιστη στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε ιδίου πόρου και δυνατότητε επενδύσεων από κοινού. Στο πρόγραμμα ανάκαμψη θα πρέπει να βρούμε χρηματοδότηση με φρέσκο χρήμα, κυρίω με ε, τα ομόλογα τη ανάκαμψη που θα καλύπτει ο ευρωπαϊκό προπολογισμό. Θα πρέπει να υπάρχει σωστή εξισορρόπηση μεταξύ δανείων και επιχορηγήσεων. Θα πρέπει, συνάδελφοι, να σκεφτούμε ότι εδώ μπορούμε να ορίσουμε μια νέα πορεία. Μια νέα πορεία για την οικονομία μα που να είναι φόρος να ε, βεβαιωθούμε ότι υπάρχει ανεξαρτησία τη Ευρώπη και καλύπτονται τα στρατηγικά μα συμφέροντα. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στι δαπάνε του μέλλοντο και ε, να κοιτάξουμε και τι κλιματικέ προκλήσει αλλά και την ε, στρατηγική μα βιομηχανία. Περισσότερο από ποτέ είναι κεφαλαίο σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργηθούν προποθέσει για μια Ευρώπη βιώσιμη, ανθεκτική και αλληλέγγυα. Ευχαριστούμε. Και τώρα για 1,5 λεπτό η συνάδελφος το Βαλιέρη. Ευχαριστώ. Είμαι Ιταλίδα και απογοητεύομαι με τα μέτρα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσουμε την οικονομική κρίση μετά την πανδημία. Ε, είναι καθυστερημένα, τσαπατσούλικα και επικίνδυνα για τη χώρα μα, διότι είναι από τι χώρε που συνεισφέρουν στον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση ω ε, βασική χώρα και δεν έχει ποτέ τι ε, ίδιε ωφέλειε με τα άλλα Εδώ με το Ταμείο Ανάκαμψη και το Ευρωπαϊκό Ευρωπαϊκού προπολογισμό βλέπουμε ότι τα κονδύλια, ακόμη και αν διατεθούν για την ανάκαμψη, δεν θα φτάσουν πριν του χρόνου. Θα είναι ήδη πολύ αργά. Χρειάζονται τώρα πόροι. Και μάλιστα όχι στη μορφή ε, δανείων. Διότι εάν τώρα δανειστούν χρήματα σε δεν μπορούν να τα αποπληρώσουν, δεν είναι ούτε κίνηση αγάπη, ούτε χειρονομία αλληλεγγύη. Είναι πραγματικά κερδοσκοπικό και το κοβλευτικό. Εδώ λοιπόν μα είπατε για το μηχανισμό ε, που θα μα σώσει, αλλά ε, χωρί προποθέσει υποτίθεται. Θα πρέπει όμω μετά τη συμφωνία του Eurogroup να δούμε τι έγινε. Ξεκίνησε από το μηδέν. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τα τέσσερα δις ετησίω που η Ιταλία πρέπει να καταβάλει ε, και ε, έχει οδηγήσει σε καταστροφή το υγειονομικό σύστημα. Εδώ λοιπόν οι Ιταλοί δεν πιστεύουν πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δείξτε μα εσύ γιατί πρέπει να πιστεύουμε. Δεν θέλουμε να έρθουμε σε μερικά χρόνια και να έχουμε πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα έρθει στην Ολομέλεια και θα πει ότι προθύστερα επέβαλε έβαλε μια λιτότητα για να γίνει η ανάκαμψη όπως παλιότερα είχε γίνει με τους Έλληνες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε συνάδελφε το Βαλιέρη και τώρα για ένα λεπτό ο συνάδελφος Ουρτασούν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχουμε τώρα ένα σταυροδρόμι να περάσουμε ή όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε την πανδημία ε, ή θα πρέπει να πάνε στον ε, λανθασμένο δρόμο τα θεσμικά όργανα. Ε, έχουμε όλη αυτή την ολοκλήρωση που είναι προηγούμενες γενιές και θα πρέπει όλες οι χώρες να προχωρήσουν μαζί, μην έχουμε τους καλούς και τους κακούς από να έχουμε αυτή την ευθύνη, όπω έγινε δημοσιονομικά τα τελευταία χρόνια. Ε, να έχουμε αυτά τα δύο δι τουλάχιστον για την ανασυγκρότηση, αυτά να γίνουν με μεταφορέ πόρων, να μην επιβαρύνουν περαιτέρω τα κράτη-μέλη και να υπάρχει ένα σύστημα ιδίων πόρων που να εξασφαλίζει ε, την ε, επιστροφή των οφειλωμένων και να καλύπτει και το θέμα των τόκων. Όχι, δεν θέλουμε να, να μας παρουσιάζεται κάποιο είδου δίθεν μαγικούς πολλαπλασιαστέ. δεν μας πάνε πουθενά αυτά. γραστείτε, αυτά τα οποία λέμε ε, και να περάσει αυτό αυτή τη βδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, συνάδελφε Ορτασόν. Ευχαριστούμε. Για, ένα λεπτό, ο συνάδελφο ε, κ. Ρούισεν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, τα πιο πολλά που ακούσα εδώ δεν με βρίσκουν σύμφωνο η, κορονο... η κρίση του κορονοϊού ε, ζητά αλληλεγγύη. Η συνοχή θα πρέπει να δημιουργηθεί με διαφορετικό τρόπο, πιο στοχευμένα. Αλλά αυτά που ζητάμε είναι πολύ παραπάνω από αυτό. Τεράστια αύξηση του προπολογισμού, νέου ευρωπαϊκού φόρου, ε, ε, κρατική χρέωση, τη οποία θα αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση αντί για τα κράτη-μέλη. Πρόκειται για μια μεγάλη κίνηση προ μια ένωση μεταφορών, η οποία προκαλεί διχασμό των πολιτών. Και στο μεταξύ με το ευρώ έχουμε χάσει το πιο σημαντικό μέσο για το, την οικονομική ανάκαψη, την ε, υποτίμηση της εθνικού νομίσματος. Σε κάποιες περιπτώσεις θα ήταν καλύτερο να επανέλθουμε στα εθνικά μας νομίσματα αλλά θα πρέπει να προβλέψουμε τι θα γίνει στην περίπτωση αυτή. Καλό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το αντιμετωπίσει αυτό και να προετοιμαστεί, γιατί θεωρώ ότι είναι πιο σκόπιμο και πιο σκόπιμη η κατεύθυνση παρά σε σχέση με τις προτάσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή επιτάπητος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Ένα μισή λεπτό ο Μπελαμή. Κύριε Πρόεδρε, Όλες οι κρίσεις αποκαλύπτουν διάφορα πράγματα και αυτή η κρίση θα αποκαλύψει διάφορα πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βγαίνει από την εμπειρία αυτή με δεδομένη την ευαλωτότητά τη. Σήμερα λοιπόν θα πρέπει να αντιδράσουμε και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα μια νέα αλληλεγγύη. Αυτό, στη συζήτηση αυτή για τον προπολογισμό και για το πρόγραμμα ανάκαμψη. θα πρέπει να ξεκινήσουμε ε, τους σκοπούς που προσκεφτούμε τα μέσα. Έχουμε ακούσει πολλά μεγάλα πόσα, αλλά αυτά τα χρήματα τι θα σκοπό θα εξυπηρετήσουν, πού χρειάζονται πραγματικά, πώ μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι. Αυτό είναι το ερώτημα από το οποίο θα πρέπει να ξεκινήσουμε το επόμενο καιρό. Θα πρέπει να αντιδράσουμε γρήγορα και γι' αυτό λοιπόν μου προκαλεί έκπλεξη το γεγονό ότι μιλάτε για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο ενώ μιλάμε για ανακάμψη ανακάμψης ε, έκτακτης ανάγκη που χρειάζεται. Πώ θα περιμένουν οι επιχειρήσει ε, και πώ θα λειτουργήσουν σε πλήρη σύγχυση. Και τέλος, αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει αύριο να δημιουργήσουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία θα δώσει μια απάντηση στην παγκοσμιοποίηση και αυτό είναι το διακύβευμα μακροπρόθεσμα. Θα πρέπει να παράγουμε αυτά που χρειάζουμε, να δημιουργήσουμε μια Ευρώπη η οποία θα δώσει ε, τη δυνατότητα στους ε, πολίτες της να έχουν μάσκες, στου νοσοκόμους, σε όλους αυτούς. Αυτό περιμένουν οι πολίτες. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη και ελπίζω να έρθουμε στο ύψος των περιστάσεων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε στην αδελφέ Μπελαμή. Η κυρία Φαμπρέμπτ έχει το λόγο. Είναι λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση σε αυτή τη μεγάλη κρίση υγείας και οικονομική και κοινωνική κρίση είναι η μεγάλη λυγγύη μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών. Η ίδια συλλελεγγύη θα πρέπει να αποτυπωθεί και στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο πρόγραμμα ανάκαμψης. Αλληλεγγύη σημαίνει να κοιτάξουμε και τη οικογενειακή ε, δικαιοσύνη και την κοινωνική ε, δικαιοσύνη βασιζόμενη στο Πράσινο Σύμφωνο και στον κοινωνικό πυλώνα. Ένας δεύτερος λόγος για την αλληλεγγύη είναι το μεγάλο πρόγραμμα επενδύτησης ε, το οποίο ζητάμε από όλο το Κοινοβούλιο βασίζεται σε ομόλογα, όπως και να τα αποκαλέσουμε, σε ομόλογα, αλλά, αλλά το τονίζω αυτό και σε μια δίκαιη και αλληλέγγυη οικονομική διαμόρφωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτό είναι κρίσιμη σημασία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, συνάδελφε Φαμπρέμπτ. Και τώρα για ένα λεπτό, ο κύριος Τούρβαλτς. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αυτές οι τελευταίες λέξεις, τις τελευταίες ε, εβδομάδες ε, ε, είχαμε παραδείγματα λοιπόν, Ευρωπαϊκής Ελληνικής. Πώς θα αντιμετωπίσουμε λοιπόν τα θέματα αυτά προκειμένου να μην ξαναξεκινήσουμε από εκεί που ήμασταν στην αρχή, πριν την κρίση. Το ακούσαμε αυτό ήδη σήμερα. Τι συζητάμε λοιπόν σήμερα, συζητάμε τον προπολογισμό και πώς μπορεί να υπάρχει συγκατανομή των ε, επιβαρύνσεων και των ευθυνών. Να μην ξεχνάμε ότι ένας ευρωπαϊκός ε, προϋπολογισμός, ο οποίος είναι 30 φορές ε, πάνω από τον προϋπολογισμό της Βουλγαρίας, δεν είναι απόλυτα αλληλεγγύης. Δεν έχω να προσάψω τίποτα στη Βουλγαρία. Αλλά αυτό που χρειαζόμαστε είναι να χρησιμοποιήσουμε τους απαραίτητους ιδίους πόρους όπως έχει γίνει και στο παρελθόν, να έχει προσταθεί και στο παρελθόν. Αυτή είναι η καλύτερη αντιμετώπιση της κρίσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Τόρβαλτς, ένα λεπτό, κύριε Σολιβιέ. Θα σας αναφέρω ένα ταμπού εδώ στο Κοινοβούλιο η απόφαση της 5ης ε, Μαΐου του Στεγματικού Δεστήριου της Γερμανίας σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα τώρα δεν μπορούμε να μπούμε ούτε σε νομική ούτε σε ε, συζήτηση για τα οικονομικά αλλά τι λέει αυτή η απόφαση αυτή η απόφαση είναι ένα τελεσίγραφο. Υπάρχει μια συγκεκριμένη παράδοση ε, όσον αφορά την εξουσία της δικαστικής ε, αρχής. Ε, τι έκανε. Έκανε κάτι πάρα πολύ εθνικιστικό το δικαστήριο της ε, Καλσρούης. Ότι δεν υπάρχει ομοσπονδιακή δομή, ότι ο καθένας θα πρέπει να φροντίζει τους συμπατριώτες του και όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι υπερέχει το κοινοτικό του εθνικού δικαίου όμως ε, ε, να τι, τι έγινε. Καθόμαστε και συζητούμε για την Μακεδονία και το Κόσοβο ενώ ταυτόχρονα υπάρχει ένα δράμα και πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη. Βλέπουμε το ότι συνεχίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αγνοεί αυτά όλα τα μηνύματα που της έρχονται. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ολιβιέ, η συνάδελφος Κίζερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε συνάδελφοι, καλωσορίζω το γεγονό ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα κάνουν άνευ προηγουμένου προσπάθειε για να μετατρέψουν αυτή την κρίση σε ευκαιρία και να βεβαιωθούν ότι τα κάτι μελη που έχουν πληγεί περισσότερο θα έχουν τι ίδιε δυνατότητε για να ανακάμψουν οικονομικά. Όμω φοβάμαι ότι δεν δίνονται ίδιε ευκαιρίε στο μισό ευρωπαϊκό πληθυσμό που έχει πληγεί περισσότερο από όλου, δηλαδή τι γυναίκε. Εκείνε δουλεύουν στου κλάδου που έχουν πληγεί περισσότερο και δική του ανεργία έχει φτάσει στα ύψη. Μιλάμε για ένα πακέτο τόνωση τη οικονομία μα και περισσότεροι σκέφτονται τι επενδύσει, τι βαριέ υποδομέ και την ψηφιακή μετατροπή. Αυτό είναι σωστό. Όμω ακριβώ το μερίδιο τη γυναικεία απασχόληση σε αυτού του κλάδου είναι πολύ χαμηλό. Οι γυναίκε πολλέ φορέ εργάζονται χωρί να αμείβονται για τα κλειστά, λόγω των, σκληρών, των κλειστών σχολείων, συγγνώμη, λόγω τη φροντίδα που προσφέρουν στα παιδιά. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να σκεφτούμε τι θα κάνουμε, γιατί οι γυναίκε σα κοιτάζουν, οι γυναίκε οργανώνονται και να βεβαιωθούμε ότι το Ταμείο Ανάκαμψη θα προσφέρει ένα φωτεινό μέλλον και μεγάλε επενδύσει για να έχουν το σωστό εισόδημα και οι γυναίκες οπωσδήποτε όπως και οι άντρες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Κίζε για ένα λεπτό η συνάδελφος Ζαλεύσκα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κάποιος εδώ είπε προηγουμένως ότι βρισκόμαστε σε μια στιγμή που είναι κρίσιμη, είναι μια καμπή. Εγώ θα έλεγα ότι είναι η τελευταία ευκαιρία, η τελευταία δυνατότητα που θα έχουμε να αποδείξουμε ότι τα ιδανικά και οι ιδέε του Σούμαν ήταν δίκαια και σωστά. Είναι η τελευταία ευκαιρία που θα έχουμε να πούμε στου πολίτε ότι εδώ είμαστε στο πλευρό μα. Στο πλευρό του, συγγνώμη. Η πανδημία χτυπάει τώρα. Δεν μπορούμε να του πούμε σε ένα χρόνο και σε τρία χρόνια και σε πενήντα χρόνια ότι θα του βοηθήσουμε. Δεν είναι αυτά σκέψεις ε, και ιδέες. Τι να πούμε στον κόσμο που αυτή τη στιγμή ε, ζει στα προάστια του Παρισιού και δεν έχει να φάει. Τι να πούμε στον κόσμο που ε, δουλεύει ε, χωρίς πραγματική σύμβαση και ξαφνικά ε, βρέθηκε και στο πουθενά. Πρέπει να υπάρξει αναδιοργάνωση του πολιτέ δημοσιονομικού πλαισίου και του προπολογισμού μα. Πρέπει τώρα να στηρίξουμε τους Ευρωπαίου πολίτες. Χρειάζεται αυτού του είδου ελεγγύη. Όλα τα άλλα θα πρέπει να υποβάλλονται και να είναι υποκείμενα στην υποστήριξη των δεδοχθείς τους πολίτες. πολίτε. Μην διστάτε από τα κράτη-μέλη να βρουν περισσότερα κονδύλια. Θα πρέπει να βρούμε το φρέσκο χρήμα με ίδιου πόρου. Ευχαριστούμε κυρία Ζαλεύσκα. Για 1,5 λεπτό η κυρία Σπυράκη. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αντιπρόεδρε Σεύκοβιτ, το γεγονό ότι η κυρία Φοντερ παρουσίασε εδώ στο σώμα το νέο Ταμείο Ανάκαμψη μα γεμίζει ελπίδα. Είναι ένα ταμείο εμπροστοβαρέ, ένα ταμείο επενδυτικό με βάση τι προτεραιότητε του Green Deal, ένα ταμείο αναλογικό για τι ανάγκε των κρατών μελών ωστόσο αυτό το νέο υπερόπλο που έχει καθυστερήσει αρκετά οφείλει να μην επιβαρύνει υποχρεωτικά με επιπλέον χρέος χώρες όπως η πατρίδα μου η ελλάδα που ήδη χτυπήθηκαν από την κρίση χρέους και την προηγούμενη δεκαετία έχασαν 25% του αεπ τους. να δίνει τη δυνατότητα να υποστηρίζονται οι οικονομίες κυρίως με επιχορηγήσεις mostly grants όπως ακριβώς λέμε στο κείμενό μας το οποίο θα ψηφίσουμε αύριο με ευρύτατη πλειοψηφία εδώ στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο να συνδυάζεται με όλα τα άλλα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία την ποσοτική χαλάρωση της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας το επενδυτικό πρόγραμμα της ευρωπαϊκής τράπεζας επενδύσεων και τα πολύ χαμηλού επιτοκίου δάνεια του μηχανισμού στήριξης καθώς και με έμεσες ανάγκες των εθνικών συστημάτων υγείας που πρέπει οπωσδήποτε να χρηματοδοτηθούν το βέβαιο είναι ότι η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε αυτή την περίοδο είναι μια πρόκληση υπαρξιακή για την ευρωπαϊκή ένωση και θα ήθελα να καταλήξω ως εξής είμαστε όλοι ξέρετε στο ίδιο καράβι. εάν δεν λειτουργήσει η ενιαία αγορά εάν δεν ενισχυθούν με ρευστότητα οι επιχειρήσεις μας εάν δεν διατηρήσουμε τη συνοχή των κοινωνιών μας και δεν αντιμετωπίσουμε το κύμα της ανεργίας που έρχεται κανένας μας δεν θα διασωθεί ούτε θα ταξιδεύει ούτε θα αγοράζει ούτε τεχνολογικό εξοπλισμό θα έχει ούτε αυτοκίνητα ούτε τουλίπες. σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Σπυράκη. Για ένα λεπτό ο συνάδελφος Λαρουτούριου. Κυρία Φόντερ Λάιεν, σε Τρει μόλι μέρε, ένα εκατομμύριο πολίτε συνυπέγραψαν την επιστολή τη ΑΒΑΖ που λένε ότι υπολογίζουν σε εσά για ένα πραγματικό προπολογισμό για το κλίμα και την απασχόληση. Ω εισηγητή για τον προπολογισμό, πιστεύω ότι μια από τι λύσει για να χρηματοδοτηθεί ε, ένα προπολογισμό είναι ένα φόρο για τι χρηματοοικονομικέ συναλλαγέ. Όταν αγόρασα αυτό το τηλέφωνο, πλήρωσα φόρο ΦΠΑ 19%. Για τα βασικά τρόφιμα είναι 5,5% ΦΠΑ. Όμω και οι πιο φτωχέ οικογένειε πρέπει να το πληρώσουν αυτό το 5,5% για να συμβάλλουν στι κοινέ προσπάθειε. Ωστόσο, αυτοί που αγοράζουν μετοχέ στι χρηματοοικονομικέ ε, αγορέ πληρώνουν φόρο 0,0%. 0,0% σα λέω. Είναι πιο φτωχοί και από του φτωχού. Προφανώ και όχι. Είναι λοιπόν επίγον να δημιουργηθεί ένα φόρο χρηματοπιστωτικών ε, συναλλαγών. Ήδη το 2011 η Επιτροπή Μπαρόζο είχε συντάξει μια οδηγία που ήταν ένα σχέδιο θα μπορούσε σήμερα να παράγει 500 ευρώ. Αυτό έχει συνταχθεί, υπάρχει ω κείμενο και παρά την κρίση την οικονομική, αυτό, παρά το Brexit θα μπορούσαμε να έχουμε 500 δι. Τι περιμένουμε, θα είναι 10 ε, φορέ παραπάνω από τον φόρο το ψηφιακό. Πρέπει λοιπόν τώρα ε, να ε, κάνουμε κάτι, κυρία Φοντερ Λάιεν, για την ζωή των πολιτών, για το σύμφωνο του κλίματο και τη απασχόληση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, συνάδελφε Λαρουτουρού, και τώρα για ένα λεπτό συνάδελφο Κόβαρικ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε η κατάσταση αλλάζει από πανδημία, γίνεται οικονομική κρίση, θα πρέπει να αντιδράσουμε ταχαίως στην Ευρώπη τώρα. Δούμε τον νέο προπολογισμό. Ε, αυτό θα πρέπει να είναι η απάντησή μας. Θα πρέπει επομένω να προσέξουμε να βρούμε προγράμματα τα οποία αποδίδουν και να υπάρχουν κάποια προγράμματα συνοχής αποδοτικά. Επίσης να προσέξουμε τις επενδύσεις. Πολύ θετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, σε σχέση με το ότι χρειάζονται νέα επενδυτικά πιο αποφασιστικά προγράμματα επενδύσεων, αλλά να δούμε επίσης πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις ε, μικρές επιχειρήσεις, να βοηθήσουμε την απασχόληση, να καλύψουμε ε, τις περιφέρειες, την καινοτομία, την ε, καινοτομία στην τεχνολογία και επίσης να μπορέσουμε να βοηθήσουμε να υπάρχουν ε, περισσότερες δυνατότητες από πλευρά εσωτερικής ε, αγοράς. α πρέπει να δράξουμε την ευκαιρία. Σας ευχαριστούμε κύριε Κόβαρικ. Μπόρκια, ένα μισή λεπτό. Οι γραφειοκράτες εδώ είναι, είναι ταχυδακτηλουργοί της ε, οικονομίας. Μιλάμε για δισεκατομμύρια τα οποία επιβάλλουν. Αλλά αυτό με φύγει άμεσα. Βλέπουμε εδώ τι λένε οι Financial Times για το ε, Ταμείο Ανάκαμψης. Λένε ότι αυτό θα είναι μια κίνηση χωρίς ε, νόημα σε σχέση με αυτά που χρειάζεται ο κόσμος. Δεν θα πρέπει να έχουμε ε, ε κάποιους ψευδεστήσεις γιατί αυτά που ανακοίνωσαν ως δισεκατομμύρια βοήθειας δεν θα κάνουν τίποτα. Ε, δεν ε, ε, είναι σωστό το να κατηγορούνται και να πληρώνουν την ύφη πιο αδύνατη. Θα πρέπει επομένως να ληφθεί υπόψη ότι αυτά όλα που λέει η Ευρώπη για ε, την κρίση και για τις κρατικές επιχορηγήσεις είναι πράγματα ανεφάρμοστα. Άκουσα τι είπε ο Σαλ ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, στρατηγική αυτονομία της Ένωσης. Θα πρέπει να μπορούμε να παράγουμε εδώ τα βασικά αγαθά. Όχι, όλα αυτά είναι μια ένα πισωγύρισμα ε, νεοφιλελεύθερο και εμείς όλα αυτά τα καταγγέλουμε. Ευχαριστώ και τώρα ο λόγος στον συνάδελφο Τόμας Βάιτς. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βρισκόμαστε λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο όλοι μεταξύ μας σε μια συλλογική κρίση και αυτό μας δίνει μια πρόγευση του τι επέκειται σε ό,τι αφορά την κλιματική κρίση. Όλους λοιπόν εδώ το Κοινοβούλιο και στις εθνικές κυβερνήσεις που προσπαθούν να επωφεληθούν από την κρίση αυτή και να υπονομεύσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, ήθελα να τους πω το εξή ότι θα πρέπει να ε, αποδώσετε ευθύνε στην επόμενη γενιά. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν ένα καλά χρηματοδοτούμενο σύστημα και να δούμε τι ιδιωτικοποίησεις. Όποιοι θέλουν ιδιωτικοποίηση σήμερα και δεν καταλαβαίνουν ότι χρειάζεται ένα καλό σύστημα υγείας σε όλη την Ευρώπη δεν έχει μάθει τίποτα από το πάθημα του COVID. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και τώρα ο λόγος στον κύριο Βέιμερς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολλοί Ευρωπαίοι ενδεχομένως να μην γνωρίζουν ε, την, ε, το κινητικό τελειτουργικό που σήμερα σημαίνει να δείχνουμε μεγάλο σεβασμό σε κάποιον ε, υψηλό βαθμό. Η ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία στο Πεκίνο αποδέχθηκε υπερβολική λογοκρισία και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε τον ε, ιό του Χαν στο τελευταία συνάντηση, αλλά δεν αναφέρθηκε ούτε στην Κίνα, ούτε στο Κομμουνιστικό ε, Κόμμα, ούτε για την ανάγκη για μια διεθνή έρευνα. Αυτός είναι ο κόσμος ε, του ΕΛΚ. Σφραγίστηκε το Γουφάν, αλλά επιτρέπηκαν οι πτήσει ε, στην υπόλοιπο κόσμο. Να σταματήσει λοιπόν αυτή η τελειτουργική επίδειξη σεβασμού. Ευχαριστούμε πολύ και τώρα ο λόγος στον κύριο Κόβατσεφ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι Ευρωπαϊκή Ένωση Αλληλεγγύης σε καλούς και χαλαπούς καιρούς. Απευθύνω λοιπόν έκκληση για να επιδείξουμε αλληλεγγύη τώρα για να εξέλθουμε από την κρίση. Πρέπει να βοηθήσουμε αυτούς που πλήττονται πιο έντονα στον τουρισμό, όχι όμως τους βάρων, τις βάρος της πολιτικής συνοχής. Θα πρέπει να επενδύσουμε και να δημορφώσουμε ένα πιο φιλόδοξο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και ένα ταμείο ανάκαμψης όπου θα υπάρχουν επιδοτήσεις, όχι όμως ή το ένα ή το άλλο. Δεν θα πρέπει να επιλύσουμε τα καταπήγοντα προβλήματα του σήμερα υποσκάπτοντας το μέλλον μας. Αυτό θα σήμαινε ακόμα μεγαλύτερες ε, διαφορές στο μέλλον. Κύριε Σεύκοβιτ, σας καλώ λοιπόν και την Πρόεδρο Φόντερ Λάιεν να απευθυνθείτε στους πολίτες τηλεοπτικά, να εκφράσετε τη συμπόνια μαζί τους και να πληροφορήσετε για τα μέτρα. Να μην επιτρέψουμε θεωρίες, συνωμοσίε να προκαλήσουν διχασμό στον κόσμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Και τώρα ο λόγος στον κύριο Ούσακοφ. Πρόεδρε, συνάδελφοι, είναι αλήθεια το να ξοδεύουμε δισεκατομμύρια από το χρήμα των Ευρωπαίων φορολογουμένων δεν πρέπει να πάει χαμένο. Θα πρέπει να, επικρί... να επενδύσουμε στην ψηφιακή οικονομία, την πράσινη οικονομία και την ελεγγύη. Θα πρέπει να κοιτάξουμε λοιπόν τι ακριβώ κάνουμε. Εγώ έρχομαι από την ε, Λετωνία, από τι χώρε τη Βαλτική. Η χώρα μα έχει πληγεί πάρα πολύ και η οικονομική μετάβαση που περάσαμε τη δεκαετία του 90 ήταν πολύ δραματική από τον ε, κομμουνισμό στην ε, ελεύθερη αγορά. Χρειάστηκαν από το μηδέν λύσει. Χρειάστηκε οι παραδοσιακοί κλάδοι να καταρρεύσουν για να ξαναχτιστούν τα πάντα. Και ήταν δεκάδε χιλιάδε οι Λετωνοί που έχασαν τη δουλειά του και δεν μπόρεσαν να ξαναφτιάξουν μπουν, να ξανέχουν πρόσβαση στην ε, αγορά εργασία. Ε, γιατί ε, παρόλο που πήραν νέα μόρφωση, νέε δεξιότητε, δεν ζητούνταν οι δεξιότητέ του. Τώρα το Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει ένα φιλόδοξο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, ένα φιλόδοξο ταμείο ανάπτυξη, ανάκαμψη, συγγνώμη. Θα πρέπει όμω να εξυγχρονίσουμε την οικονομία μαζί με, δεξι... με τι δεξιότητε και μαζί με του εργαζομένου που θέλουν να δουλέψουν σε κλάδου που δεν θα υπάρχουν πια. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε συνάδελφε Ούσακοφ για ένα λεπτό ο συνάδελφος Ντάντι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιτέλους αποφάσισε ένα σοβαρό πρόγραμμα παρεμβάσεων για να αντιμετωπιστεί η κρίση του κορονοϊού. Βεβαίως, θα έπρεπε αυτό να έχει γίνει νωρίτερα Τώρα περιμένουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει μια πρόταση που να μπορεί να λειτουργήσει για τα Ταμείο Ανάκαμψη. Μια πρόταση η οποία να είναι στα σωστά επίπεδα από την άποψη των μεγεθών και να είναι ποιοτική. Εδώ δεν θα πρέπει να γίνει το παθή η Ευρώπη, αλλά ανθεκτική και να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο διάλυση. Διότι αυτό πραγματικά τροφοδοτείται από τι ε, εξωευρωπαϊκέ χώρε. Πρόεδρε, συνάδελφοι, αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να παράγουμε μόνο στο οικονομικό επίπεδο για να υποστηρίξουμε με τις χώρες και τους ε, πληθυσμούς που έχουν πληγεί. Θα πρέπει να αποδώσουμε πίσω στους Ευρωπαίους το όνειρο, το όραμα και τα ιδανικά τους. Έχουμε κάνει πολλές φορές επιλογές δύσκολες και αντιφατικές, αλλά πραγματικά να μην αναρωτιόμαστε μόνο τι ε, πρέπει να κάνουμε, αλλά και πώς και γιατί. Θα πρέπει να βρούμε το όραμα, τη θεώρηση για το μέλλον που χρειαζόμαστε και το θάρρος για να αντιμετωπίσουμε τους δύσκολους καιρούς που ε, κληθήκαμε να βιώσουμε. Ευχαριστούμε συνάδελφε για ένα λεπτό, ο συνάδελφος ε, Πέρεκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και θα ήθελα να αναφερθώ στη συζήτηση της 21ης Απριλίου σε ό,τι αφορά τις ε, ε, εξορίξεις της Τουρκίας κυπριακά χωρικά είδατα. Ζήνουμε σε εποχές Τώρα θα πρέπει να αποδείξουμε όμως την πράξη την αλληλεγγύη μας προς ένα κράτος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τουρκική κυβέρνηση απέδειξε ότι δεν ενδιαφέρεται για την τήρηση του διεθνούς δικαίου και αυτές οι διαδικασίε εξόριξης ε, με ε, παραβίαση του ε, εμπάργου για τα όπλα στη Λιβύη αποσταροποιεί όλη την περιοχή και σίγουρα θα είδατε την κοινή δήλωση Ελλάδας και Κύπρου Κύπρου, ε, Αιγύπτου, Γαλλία, στην οποία καταδικάζονται οι τουρκικέ αυτέ δραστηριότητε. Αυτό είναι ένα καλό και σημαντικό βήμα, αλλά σίγουρα χρειαζόμαστε πιο πολλέ ε, υποστηρίξει ε, μεγαλύτερη υποστηρίξη προ την Συρία. Η Τουρκία λοιπόν είναι αντίθετη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό δεν μπορούμε πλέον να το ανοιχτούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, συνάδελφε Μπέρκ. Και τώρα για ένα λεπτό το λόγο έχει η κυρία Μουστκαναυσικά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σήμερα τα κράτη-μέλη μας, οι πολίτες μας, οι επιχειρηματίες, οι οικογένειες μας ζητούν μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία θα δράσει κατά της πανδημίας και κατά της οικονομικής κρίσης. Θα πρέπει να επιτύξουμε ευελιξία σε ό,τι αφορά τη χρήση των πόρων και να εξασφαλίσουμε και νέους πόρους για την Ευρώπη. Το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο αποτελεί το νέο κρογωνιό λίθο για την ανάκαμψη. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την κρίση γιατί η οικονομική κρίση σημαίνει ότι θα δούμε να πέφτει κατά 7% το ΑΕΠ μας. Η οικονομία μας λοιπόν είναι τρινή θέση και θα πρέπει να προετοιμάσουμε τις επιχειρήσεις μας, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν μπορούμε να τις ξεχνάμε. Ούτε μπορούμε να ξεχάσουμε Η οικονομία μας πρέπει να διασωθεί. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη φοροδιαφυγή και πρέπει να αντιμετωπίσουμε και την έλλειψη φορολογικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τους φορολογικούς παραδείσους και θα πρέπει να ε, δούμε τι θα κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε την εμφάνιση αυτών των ε, περιπτώσεων. Ευχαριστούμε κύριο Ντόρφμαν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πραγματικά παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον τις συζητήσεις που γίνονται για το μελλοντικό πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και το Ταμείο Ανάκαμψης. Φρονώ ότι θα πρέπει το Ταμείο Ανάκαμψης να δούμε μήπως το έχουμε αναβάλει και παραγωνίσει για να πάει ε, και να παραπεμφθεί στα του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Και τα κράτη-μέλη να μην θέλουν να λάβουν τι ευθύνε του. Νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι σε σχετισμό δυνάμεων είναι πολύ σαφέ. Εδώ λοιπόν με αυτή την πολιτική βλέπουμε στο πολιτισμό συνομικό πλαίσιο να δημιουργούνται μια σειρά από προβλήματα σε καιρού ε, COVID, εκεί που οι γεωργοί μα και οι κτηνοτρόφοι μα μας έχουν εξασφαλίσει τα τρόφιμα για να τρεφόμαστε. Ουσιαστικά έχουμε 80 ε, ε, εκατομμύρια ευρώ για τα 23 κράτη-μέλη υποστήριξη ενώ ε, έχουν μείνει 19 ε, δις ε, στη διάθεσή μας θα πρέπει να τα διαθέσουμε μετά. Αυτή την πολιτική λοιπόν, την Κυριακή πρέπει να υποστηρίξουμε πάνω απ' όλα γιατί θα πρέπει να δράσουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα, να βρούμε το χρήμα που χρειάζεται και για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο να φροντίσουμε να βρεθεί λύση. Και σε αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να φροντίσουμε να υποστηρίξουμε τόσα συμβαίνουν. Ευχαριστούμε μετά τον κύριο Ντόρφμαν Λοιπόν ο κύριος Μορένο Σάντσες για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί κύριοι, τώρα έχει έναν ε, μεγάλο πρόβλημα η Ευρώπη. Μία πρόκληση, πιο μεγάλο δεύτερο πόλεμο. Χρειάζεται πολιτικό, πολιτικό θάρρο. Χρειάζεται η τόλμη που έδειξαν οι ιδρυτέ Ένωση. Να σταματήσουμε να προσιλωνόμαστε στα παλαιά νομικά και πολιτικά δόγματα. Να βρούμε το θάρρο με αλληλεγγύη να χτίσουμε μια νέα Ευρώπη. Πιο αλληλέγγυα και για αυτό το Κοινοβούλιο θα πρέπει να διαδραματίσει έναν βασικό ρόλο προσανατολισμού πολιτικού και ε, καινοτομία στα δημοσιονομικά. Να γίνει έτσι ο μετασχηματισμός και να βρούμε ένα καινούριο ΠΔΠ. Ε, χρειάζεται ένα νοπό χρήμα με το ΠΔΠ, να μην υπάρχουν τίποτε ε, κόλπα δημοσιονομικά, να καλυφθούν οι χώρες που χρειάζονται πολύ αυτή την ενίσχυση. Το είπε ο Αντενάουερ. Όλοι είμαστε κάπου τον ίδιο ουρανό, αλλά ο καθένας έχει διαφορετικό ορίζοντα. Άρα για να βρούμε ε, το κοινό μας μέλλον τον ίδιο ορίζοντα θα πρέπει να ε, ενεργήσουμε, να δείξουμε ότι είναι ισχυρό το κοινοβούλιο. Όλοι, όλες να ψηφίσουμε υπέρ του κοινού ψηφίσματος. Ευχαριστούμε κύριε Μορένο Σάντσες και τώρα για ένα λεπτό ο συνάδελφος Περέιρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πριν από λίγες μέρες ε, στα πλαίσια αυτής της πανδημίας γιορτάσαμε και την Ευρώπη. 70 χρόνια ενός προγράμματος ειρήνης και ένωσης των Ευρωπαίων. Ένα εγχείρημα που ε, μας θύμισε και ο Σούμαν δεν θα χτίσουμε την Ευρώπη σε μια μέρα, ούτε με, σε ένα ε, και μόνο οικοδόμημα. Όντως βρισκόμαστε όλοι στα ίδιο καράβι. Και από τη δική μου την πλευρά δεν θα υποστηρίξω ότι η Ευρώπη θέλει να βυθιστεί. Η στρατηγική για την οικονομική ανάκαμψη από την πανδημία αυτή θα πρέπει να βασιστεί στα πρόσωπα τους Ευρωπαίους, τους νέους που αντιμετωπίζουν αντιμετωπίζουν ήδη τη μεγαλύτερη κρίση τη ζωή του, για του επιχειρηματίε που καθημερινά δίνουν αγώνα για να πληρώσουν μισθού, στου ανέργου που ζουν στιγμέ μεγάλη δυσκολία αυτοί όλοι ε, όντω ε, μα οδηγούν να βρούμε ένα καινούριο πρόγραμμα για να εξυγχρονιστούν οι οικονομίε μα. Δεν είναι το Κοινοβούλιο, αλλά είναι το Συμβούλιο που μπλοκάρει τι απαντήσει που τόσο κατεπηγόντω χρειαζόμαστε. Αυτή τη στιγμή πρέπει να λάβουμε τι δικέ μα ευθύνε, να φροντίσουμε η Ευρώπη να έχει περισσότερο μέλλον μπροστά τη από ό,τι είχε παρελθόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Περέιρα και τώρα για ένα λεπτό ο συνάδελφος Φεραντίνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Κυρία Φόντερ Λάιεν, σα ζητούμε να προβλέψετε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που να ανταποκρίνεται στι ε, προσδοκίε των πολιτών και των επιχειρήσεων που πλήγησαν από την πανδημία COVID. Θα αντιμετωπίσουμε μια οικονομική καταστροφή χωρί προηγούμενο. Το ψήφισμα που βάλουμε σήμερα είναι μια σαφή απόδειξη τη ευθύνη και τη συμπόνια που δείχνουμε σε μια τόσο δυσχερή στιγμή, αλλά και διεκδίκηση του κεντρικού ρόλου που θέλουμε να έχει το Κοινοβούλιο. Δεν μπορούμε να είναι όμοιρο των κυβερνήσεων η Ένωση. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε τώρα για να υπάρξουν κατάλληλε παρεμβάσει για του πολίτε και τι επιχειρήσει. Όχι όπω το 2008 όταν κοιτάξαμε να σώσουμε τι τράπεζε. 200, μάλλον 2.000 δι μόλι παρκούν για να σώσουμε την οικονομία ε, ε, τις οικονομίες των κρατών μελών. Δεν θέλουμε να είναι καινονοήματο ε, το Ταμείο απάντηση στον COVID. Θα πρέπει να βρούμε πράσινε λύσει στην οικονομική αντίσταση κάποιων. Οι Ευρωπαίοι πολίτε χρειάζονται τώρα απαντήσει Ο τουριστικός κλάδο, του αθλητισμού, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή των εστιατορίων. Όλοι χρειάζονται τώρα μια απάντηση, διότι τώρα θα αντιμετωπίσουμε τη χειρότερη οικονομική κρίση. Και τα οικονομικά μέτρα δεν πρέπει να τα πάρουμε με περικοπέ από τα διευθυντικά ταμεία θα πρέπει να βρούμε άλλες λύσεις. Ευχαριστούμε πολύ, συνάδελφε Φεραντίνο. Και τώρα για ένα λεπτό ο συνάδελφος Τομπέ. Ε, Κύριε Πρόεδρε, η Ευρώπη τώρα για να αντιμετωπίσει την κρίση από την εποχή της τελευταίας οικονομικής κρίσης βρίσκεται στη χειρότερη θέση. Χρειάζεται να υπάρξει ένας προϋπολογισμός σύγχρονος που να βοηθά την ανταγωνιστικότητα. Χρειάζεται όμως και μια οικονομική πολιτική με υπευθυνότητα. Αυτή η δέσμη μέτρων διάσωσης ε, δεν αφορά μόνο κάποιες ε, άμεσες καταβολές και επιχορηγήσεις θα πρέπει να υπάρξουν και κάποια δάνεια, δάνεια που να επιστραφούν ε, γιατί να έχουμε μια δημοσιονομική πολιτική ε, που να μην βασίζεται σε φόρους αλλά σε μεταρρυθμίσεις. Η ευρωπαϊκή ε, συνεργασία είναι το ίδιο με την αλληλεγγύη. Δεν είναι δυνατόν εμείς να συμφωνήσουμε με ένα τέτοιο ψήφισμα. Ευχαριστούμε για ένα λεπτό η κυρία Γιονγκέριος. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ένα στου δέκα Ευρωπαίου πρόκειται να μείνουν χωρίς δουλειά φέτος λόγω της πανδημίας. Αυτή είναι η πρόβλεψη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και βέβαια ε, στατιστικά κρύβουν πραγματικούς ανθρώπους με ουσιαστικές ανάγκες. Αυτές όλες οι ανάγκες τους τώρα ε, θα, ε, θα γιατί θα, δεν θα έχουν δουλειά. Άρα πρέπει να ξαναβρούν τη δουλειά τους και θα πρέπει επομένως να ενεργοποιήσουμε ε, τον κοινωνικό πυλόν. Γι' αυτό όμως χρειάζονται χρήματα κάποιες βιώσιμες της απασχόλησης ε, και η καταπολέμηση της φτώχειας επίσης δεν γίνεται χωρίς ε, ε, χρήματα. Ναι, είναι ωραία είναι να βγαίνουμε και να χειροδούμε στα μπαλκόνια, αλλά χρειάζονται περισσότερα, να επενδύσουμε περισσότερο στο κοινωνικό ταμείο, στην πρωτοβουλία για την ανεργία των νέων. Επομένως, ας επενδύσουμε στον άνθρωπο τώρα και έτσι θα γλιτώσουμε τα χειρότερα. Ευχαριστούμε κυρία Γιονγκέριους. Ακολουθεί για ένα λεπτό ο κύριος Λούτκεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ την Πρόεδρο Φόντερ Λάιεν και τον Πρόεδρο Μισελ που επιβεβαίωσαν τη βούλησή του να δημιουργήσουν μια πράσινη συμφωνία και να την εντάξουν στο πρόγραμμα ανάκαμψη. Αυτό το πρόγραμμα ανάκαμψη θα πρέπει να προβλέπει μια πράσινη σύγκληση και την ε, αυτάρκεια τη Ευρώπη τομεί τόσο στρατηγικού όπω αυτό τη υγεία. Το ανέφεραν κάποιοι, αλλά και σε άλλου κλάδου. Όπω τη επιστημιστική ασφάλεια για του γεωργού και κτηνοτρόφου. Για να υπάρχει μια στρατηγική ανεξαρτησία και αυτονομία. Γιατί και στην ενέργεια το χρειαζόμαστε αυτό. Θα πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραμμα ανάκαμψη που να προβλέπει να είμαστε στο το δυνατόν πιο ανεξάρτητη σε θέματα ενέργεια. Να υπάρχει ευρωπαϊκή ε, κυριαρχία και ε, ασφάλεια στα θέματα τα ψηφιακά. Θα πρέπει να ξεκινήσει η πράσινη οικονομία ε, και να προασπιστούμε την άμυνα και την ασφάλειά μα ταυτόχρονα. Βεβαίω, ω Ευρωπαίο συνηγορεί υπέρ και του να έχει η Ευρώπη επιτέλου ίδιου πόρου με την φορολόγηση τη βενζίνη, με τη φορολόγηση και άλλων συναλλαγών, ώστε να έχουμε επιτέλους τη διάθεσή μας τα μέσα που χρειαζόμαστε για την οικονομική μας αυτάρκεια και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε συνάδελφε Λουτκέν και για ένα λεπτό ο συνάδελφος Μάρκες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, συνάδελφοι. Ε, το, Βούλιο αυτό χαιρετίζει το σημαντικό βήμα που έγινε στο προηγούμενο Συμβούλιο, στη Ευρωπαϊκή Ένωση να υπολογίζει το χρέο τη ε, ελαστικά, ώστε να, χωρίς να τιμωρούνται τα κράτη-μέλη που έχουν ε, πληγεί περισσότερο. Τώρα αντιμετωπίζουμε μια στιγμή ιστορική, τη μεγαλύτερη μετά από τον τελευταίο μεγάλο πόλεμο και πρέπει αμέσω να βρούμε τα κατάλληλα μέτρα. Το πρόγραμμα που ξεκάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να είναι φιλόδοξο. Δεν αρκεί να βρούμε μερικά χρήματα από την αγορά και κάποιου πολλαπλασιαστέ, με λίγο marketing, αλλά θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ανακτηθεί, για να ξαναστήσουμε στα πόδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για του πολίτε, του καταναλωτέ, τι οικογένειε και για την εμπιστοσύνη των επιχειρηματών και των εταιριών. Θα πρέπει να σώσουμε την απασχόληση στην Ευρώπη. Θα πρέπει και γι' αυτό το σκοπό να βρει ένα άλλο ρόλο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εδώ δεν ζούμε σε κανονικού καιρού. Η νομισματική πολιτική θα πρέπει να αλλάξει και μάλιστα όσο το δυνατόν περισσότερο. Θα πρέπει οι Ευρωπαίοι πολίτε να μην αγωνίζονται θα πρέπει τώρα τα Ευρωπαϊκά Συμβου... το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να δείξει αλληλεγγύη με του πλέον αδύναμου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μαρκέ. κυρία Βερκούνεν. Κυρία Βερκούνεν. Η κυρία Ρέγνερ. Ευχαριστώ. Τα θεμέλια τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι άνθρωποι και την βοήθεια μα τη χρειάζονται τώρα, όχι όποτε να είναι. Πρέπει να βρούμε μια απάντηση σε αυτή την κρίση. Θα πρέπει να έχουμε περισσότερο θάρρο, περισσότερη ελεγγύη και πολύ περισσότερη Ευρώπη. Πρέπει να φανούμε τολμηροί και να δούμε πώ θα βρούμε τους πόρους για αυτήν την οικονομική ανάκαμψη. Όχι όμως ε, από αυτούς που πλήρωσαν μέχρι τώρα φόρους, αλλά από αυτούς που απέφευγαν, όπως τους πολυεθνικούς ομίλους και τις επιχειρήσεις. Θα πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε τα κάτι μέλη που πηλήξαν ε, δρυμύτατα από την κρίση αυτή και ακόμη και τα κορονομόλογα θα πρέπει να τα σκεφτούμε. Θα πρέπει επίση να φανούμε αλληλέγγυοι με τι γυναίκε. Διότι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αντιμετωπιστεί η γυναική ανεργία που έχει αυξηθεί δραματικά. Θα πρέπει να βρούμε δραστικά μέτρα τα οποία φέρουν απτά αποτελέσματα, ορατά αποτελέσματα για όσου έχουν υποφέρει περισσότερο. Για όσου βρίσκονται στα σπίτια του και δεν πληρώνονται. Αυτέ οι γυναίκε που πρέπει να κάνουν μαθήματα στα παιδιά του και μπορεί και να χρειαστεί να τα φροντίσουμε χωρί να τα ειδικά κανεί. Ή αυτέ που απασχολούνται στα σούπερ μάρκετ. Όλοι ε, χρειάζεται ε, να υποστηριχθούν. Ένα ταμείο για τι γυναίκε που να δώσουν τι κατάλληλε απαντήσει. Ευχαριστούμε, συνάδελφε Ρέγνερ. Και τώρα για ένα λεπτό ο συνάδελφο Τέρα. Um, Η πρόεδρος Φοντερ Λάιον μας εξήγησε ο σκοπός είναι πως θα έχουμε μια δυνατή και ενωμένη Ευρώπη. Όμως, τι λένε οι φήμες. Ότι το πρόγραμμα αυτό ήδη έχει υποστεί περικοπές, ε, ήδη το πρόγραμμα αυτό δεν καλύπτει το πι δέλτα πι. Όμως έχουμε και την ε, στρατιωτική κινητικότητα πρόκειται για τη συνεργασία ΝΑΤΟ με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πρέπει αυτή η συνεργασία να υπονομευτεί. Έχουμε και το Green Deal, πάρα πολύ σημαντικό, αλλά και ακριβό πρόγραμμα. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί το ότι το ΠΔΠ θα προβλέπει αρκετούς πόρους, ούτω ώστε να μπορούμε να βοηθήσουμε τη γεωργία, τις επιχειρήσεις να πετύχουν τους στόχους. Αν δεν κάνουμε αυτό που πρέπει, τότε και εμείς είμαστε συνένοχοι στην οικονομική κατάρρευση με περισσότερο στρίμωγμα που θα τους προκαλέσουμε, γιατί οι γεωργοί είναι αυτοί που φέρουν περισσότερο. Ευχαριστούμε συνάδελφε Τέρας. Ευχαριστώ πρόεδρε που μου δώσατε το λόγο. Υπάρχουν κάποιοι στην Ευρώπη που κάθε μέρα ευχαριστούν που υπάρχει η ενιαία αγορά. Είναι αυτοί που δουλεύουν διασυνοριακά. Ε, για αυτούς ε, είναι το πιο σπουδαίο στις δύσκολες αυτές τις εποχές η ενιαία αγορά. Όταν λέμε για να, κάμψει, τι εννοούμε. Νομίζω ότι σημαίνει ότι θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κάποια πλήρως λειτουργούσα ενιαία αγορά, να Βία ε, οι Ανθρωπή ελεύθερα στη Σιλεσία. Το έχω δει αυτό. Πάρα πολύ όμω εκεί έχασαν τη δουλειά του. Γιατί τα κράτη-μέλη ε, φέρθηκαν εγωιστικά. Άρα θα πρέπει να το διαχειριστούμε το θέμα και αυτό το σχέδιο ανάκαμψη να ρυθμίσει το ζήτημα των δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και επομένω θα πρέπει να είναι πιο ολοκληρωμένη η εμβάθυνση. Ήρθε η ώρα ή τώρα ή ποτέ. η τωρα η ποτε Ευρώπη δεν θα πρέπει να έχει σύνορα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε συνάδελφε Κόχουτ και τώρα Κάζα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Τα μέσα ενημέρωση έχουν πληγεί πάρα πολύ από την πανδημία. Συνεχίζουν και διακινδυνεύουν τη ζωή του δημοσιογράφοι. Και όπως που γνωρίζουμε ε, έχει συρρυκνωθεί και η διαφήμιση και ε, οι συναδελφοί ε, επιμένουμε θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην εγκαταλείψει και αυτούς τους οργανωμένους θα πρέπει να τους δοθεί η βοήθεια που χρειάζονται. Βέβαια μερικοί προτείνουν να υπάρξει ένα μόνιμο ταμείο για τους δημοσιογράφους. Τα μέσα ενημέρωση είναι πολύ σημαντικά για τη δημοκρατία κανένα κράτος μέλος δεν θα πρέπει να έχει ε, κατάρρευση σε αυτόν τον ε, κλάδο. Η πανδημία έθιξε πάρα πολύ τα μέσα ενημέρωσης, άρα έθιξε και τη δημοκρατία σε πολλές χώρες. Εγώ θα συνεχίσω να πασχίζω με τους συναδέλφους ούτως ώστε να υπάρξει τελικά μια τέτοια ενίσχυση στο συντομότερο δυνατόν και έτσι θα ενισχυθεί η δημοκρατία μας. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε κύριε Κάζα. Για ένα λεπτό η συνάδελφος Γιόντσεβα. Ευχαριστούμε. Η ζωή και η υγεία δεν τιμή. Θα πρέπει να κάνουμε όλε τι απαραίτητε δαπάνε για την οικονομία και την υγεία. Όμω οι ευαλωτότεροι δεν μπορούν να ανακάμψουν τόσο γρήγορα όπω οι ισχυρότεροι. Η πανδημία φαίνεται να ε, προκαλεί διαφορετικέ επιπτώσει στα διάφορα κάτι μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να κάνω τι εξή ερωτήσει. Το πρόγραμμα ανάκαμψη δεν θα πρέπει να συμφωνηθεί μεταξύ κυβερνήσεων και κλεισμένων των θυρών. Θα πρέπει να επιτρέψει να υπάρξει δημοκρατικό έλεγχο και παρακολούθηση από το Ευρωκοινοβούλιο. Δεύτερον, είναι σημαντικό οι πόροι, τα κονδύλια να φτάσουν σε αυτού που τα χρειάζονται και όχι στου ολιγάρχε ή του λίγου. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθήσει ε, πραγματικά πώ χρησιμοποιούν αυτά τα κονδύλια τα κράτη-μέλη. Και η τελευταία, ε, παρατηρήση μου έχει να κάνει με, το, ε, με τις πραγματικές ροές. Εδώ πραγματικά καλό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κοιτάξει, να ε, επιτρέψει την ελεύθερη έκφραση και τα, να στηρίξει τα ανεξάρτητα μέσα μαζική ενημέρωση. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε την ε, κυρία Βάη. Τώρα για ένα λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλοί χάνουν ε, τη θέση απασχόλησή του στην παρούσα φάση. Χρειάζεται λοιπόν ένδειξη αλληλεγγύης. Χρειάζεται να βοηθήσουμε τους άλλους, αλλά δεν μπορούμε να προκαλέσουμε εξάρτηση. Θα πρέπει να φροντίσουμε επίσης να μπορέσουν όλοι να οργανωθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε ατομικό επίπεδο, προσωπικό επίπεδο, αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Άρα, να μην κοιτάμε τι προθέσει. Ε, είναι καλέ οι προθέσει, αναδιαφεσβήτητα, αλλά στι Βρυξέλλε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση δίζονται εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, χωρίς όρους. Αυτό δεν είναι καλό για τα άτομα αυτά. Και αυτό θα πρέπει να διτερηθεί ως αρχή, παρά την ε, κρίση του κορονοϊού. Είμαστε ενωσία δημοκρατίας, καινοτομίας. Θα πρέπει να σεβαστούμε την επικυριαρχία των κρατών μελών. Επίσης θα πρέπει να φροντίσουμε για τις ε, διασυνοριακές προκλήσεις και θέλουμε και δυτικό ανταγωνισμό και γι' αυτό λοιπόν θα υπερψηφίσω το ψήφισμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνάδελφε Βάης για ένα λεπτό η κυρία Σίλβα Περίρα. Ο κύριος Σίλβα Περίρα. Μικρό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το πρόγραμμα ανάκαμψη για την οικονομία που θα παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση να περάσει δύο σοβαρέ δοκιμασίε. Πρώτα απ' όλα, το, τη δοκιμασία τη αξιοπιστία και μετά τη δοκιμασία τη αλληλεγγύη. Για την αξιοπιστία. Δεν μπορεί να εδράζεται μόνο σε οικονομολογικέ ψευδεστήσει το πρόγραμμα αυτό. Πρέπει να έχει τα απαραίτητα μέσα για να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση ανευπροηγουμένου. Επίσης, η δοκιμασία του τεστ τη αλληλεγγύη Θα πρέπει να κινητοποιήσουμε τις απαραίτητες απενδύσει για να υπάρξει ανάκαμψη, χωρίς όμως να πιέσουμε τα κράτη-μέλη να περάσουν σε, ένα νέο, σε μια νέα κρίση των κρατικών χρεών. Αυτό θα πρέπει να το καλύπτει ο Ευρωπαϊκός Προπολογισμός με την προστασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να ε, υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες επιδοτήσεων στα κρατη χωρίς να παίρνουν τη μορφή δανείων. Να είναι ένα πρόγραμμα αξιόπιστο και αλληλέγγυο. Αυτό χρειάζεται τώρα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ζητάει περισσότερα από όσα απαιτούνται και χρειάζονται. Δεν ζητάει περισσότερα, αλλά δεν ζητάει και λιγότερα. Ευχαριστούμε συνάδελφε Σίλβα Περέιρα και για ένα λεπτό ο κύριος Μακάλιστερ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, θα ήθελα να κάνω μία επιπρόσθετη παρατήρηση μετά από την συζήτηση αυτή που άκουσα επί σχεδόν δύο ώρες. Με μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η πανδημία δεν γνωρίζει σύνορα. Ούτε θα έπρεπε να γνωρίζει σύνορα και η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωση Γι' αυτό πρόεδροι των Επιτροπών στο κοινοβούλιο αυτό προέβησαν σε μια κοινή δήλωση και ζήτησαν ε, ενισχυμένη συνεργασία με τους ε, γείτονε και τους εταίρους σε ό,τι αφορά τα θέματα καταπήγουσας ανάγκης, σε ό,τι αφορά και τις μοναδικές ε, επιδράσεις. Τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε δει τεράστιες προσπάθειες καλής θέλησης και συνεργασίας, αλλά βλέπουμε και απομονωτισμό μεγάλη, μεγάλο ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών σε ό,τι αφορά τον ε, ιατρικό εξοπλισμό και παραπληροφόρηση και κυβερνοεπιθέσεις. Αυτό καταδεικνύει ότι η πανδημία αυτή έχει παγκόσμια σημασία. Είναι παγκόσμια πρόκληση. Το το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο θα αποτελεί το βασικό εργαλείο αντιμετώπιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την υποστήριξη των εταίρων μα και στην άμεση γειτονία μα. Αυτά θα πρέπει να καλυφθούν στο μελλοντικό πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε Μακάλιστερ. Και τέλος να ακούσουμε το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Ξεκινάει ο Επιτροπός Εύκοβιτς καταρχάς. <clears throat> Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές. Και καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συζήτηση αυτή, γιατί ακούσαμε πολύ υπομονή, πολύ φιλοδοξία στα σχολεία σας. Και νομίζω ότι σε όλες τις παρεμβάσεις υπάρχει μια σαφής έκκληση προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να βγει από την κρίση αυτή πιο δυνατή, πιο σύγχρονη, πιο βιώσιμη και πιο αντακτική. Και νομίζω ότι αυτό είπαν οι επικεφαλής, η κυρία Γκαρσία Περές, ο κύριος Τσόλος και ο κύριος Λάμπερτς. Αυτό ζήτησαν. Δεν μπορώ να σας πω πόσο ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, εκτιμούμε τη συνεργασία με το Κοινοβούλιο, ιδιαίτερα στις τελευταίες εβδομάδες, όπου εξετάσουμε το πώς μπορούμε να δώσουμε στους πολίτες μας αυτά που χρειάζονταν. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στη διάσωση όσο πιο πολύ ζωών γινόταν στην αρχή και στη συνέχεια να διατηρήσουμε τις θέσεις απασχόλησης. Τώρα λοιπόν συζητάμε το πώς θα ξαναξεκινήσουμε την ευρωπαϊκή οικονομία, πώς θα ανακάμψουμε από τη δραματική αυτή κρίση. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γι' αυτό. Γιατί με την συνεργασία αυτή καταφέραμε να πετύχουμε τις τελευταίες εβδομάδες πάνω από 200 μέτρα κάποιες πολύ σημαντικές νομοθετικές προτάσεις τις οποίες εκκρίνετε εσείς και οι οποίες πραγματικά βοήθησαν συγκεκριμένα τον κόσμο επιτόπου για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης ανευπροηγουμένου. Πιστεύω ότι είναι χάρη στις προσπάθειες αυτές, στις ηρωικές προσπάθειες των εργαζομένων στον τομέα της υγείας, χάρη στην πειθαρχία των πολιτών, βλέπουμε η τρομερή αυτή η αριθμή των θυμάτων από τον κορονοϊό να μειώνονται. Όλοι όμως γνωρίζουμε ότι ήταν πολύ δύσκολη αυτή η περίοδος. Η μεγαλύτερη δοκιμασία όμως είναι ακόμα μπροστά μας το πώς θα καταφέρουμε να ανακάμψουμε από την κρίση αυτή, πώς θα μπορέσουμε να ξαναξεκινήσουμε την οικονομία μας, να επανέλθουμε σε μια φυσιολογική κατάσταση και όπως είπε ο κύριος Βέμπερ, ίσως αυτό θα είναι η στιγμή του Σούμαν για την δική μας γενιά. Γι' αυτό λοιπόν εκτιμώ σε αυτή τη συζήτηση. Γιατί όπως είπε ο κύριος Σίλβα Περέιρα, θα πρέπει να επιτύξουμε τέτοιο επίπεδο φιλοδοξία, τόλμης, για να αποδείξουμε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και την ευρωπαϊκή αξιοπιστία. Πώς θέλουμε να το πετύχουμε λοιπόν αυτό. Επιτρέψτε μου να κοιτάξουμε κάποια από τα βασικά στοιχεία των προτάσεων επί των οποίων εργαζόμαστε στην παρούσια φάση. Θέλουμε να βασιστούμε στην αντιδρασή μας σε έναν δυναμικό προπολογισμό για το μέλλον, ένα πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο με ένα ισχυρό εργαλείο ανάκαμψη, το οποίο θα δώσει μεγάλη οικονομική ενίσχυση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό πραγματικά αποτελεί μια φιλοδοξία άνευ Άρα διαφωνώ με τον κύριο Φερχόφστατ ότι τα πράγματα είναι όπως είναι πάντα. Προσωπικά παρακολούθησα τις διαπραγματεύσεις στον τελευταία δημοσιονομικό πλαίσιο και ποτέ δεν έχω δει τέτοιο επίπεδο τόλμης και φιλοδοξίας. Και πιστεύουμε ότι με τη δική σας υποστήριξη θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην πρόκληση αυτή, την οποία έχουμε όλοι μπροστά μας. Να σας διαβεβαιώσω ότι θέλουμε να πετύχουμε πολιτικές οι οποίες έχουν δοκιμαστεί. Θέλουμε δηλαδή να ενισχύσουμε το Ταμείο Συνοχής, να επικεντρωθούμε σε αυτούς που επλήχθησαν πιο σοβαρά κατά την κρίση. Θέλουμε να βελτιώσουμε την ε, εργασία της InvestEU του ορίζοντα που είναι πολύ σημαντικός για την υποστήριξη των επιστημόνων μας. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ επίσης τη σημαντική κοινωνική πτυχή της δουλειάς μας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα της φτώχειας. Το θέμα του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης θα πρέπει να λειτουργεί σωστά. Να μην ξεχάσουμε επίσης τις γυναίκες, τους γονείς και όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ισότητα μεταξύ των φύλων. Όλα αυτά τα θέματα θα είναι σημαντικά για την ανάκαμψή μας. Επιπλέον, έχουμε νέα εργαλεία φερεγγιότητας για να αποτρέψουμε τις χρεοκοπίες οι οποίες ενδεχομένως να προκληθούν από την κρίση και για να αναπτύξουμε νέα προγράμματα υγείας για να προετοιμαστούμε καλύτερα για το μέλλον. Και πάλι λοιπόν τονίζω ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου business as usual. Δεν είναι καθόλου ο συνήθως. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη αντίδραση σε μια κρίση. Επίσης, να απαντήσω σε αυτά που είπε ο κύριος Λάμπερτς, ε, Ερτου και Eichhout για την ε, οικονομική αυτή ισχύ που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε για να δώσουμε όθηση στην οικονομία μας. Θέλουμε να την καταστήσουμε πιο πράσινη, πιο βιώσιμη την οικονομία μας και νομίζω ότι αυτή η κρίση μας δίδαξε ότι θα πρέπει να είμαστε πιο ανθεκτικοί. Τι τα θέμα λοιπόν στρατηγικής αυτονομίας, τεχνολογίας, τεχνολογική επικυριαρχία. Σε αυτού τους τομείς θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε πιο έντονα από ό,τι στο παρελθόν. Προ όλου του συναδέλφου που ανέφεραν τη σημασία των ίδιων πόρων, να πω το εξή. Να σα διαβεβαιώσω ότι εργαζόμαστε και έχουμε ανοιχτέ όλες τις λύσεις ενώπιον μα τι ακούσαμε τι πιο πολλέ στη συζήτηση αυτή. Θα παρουσιάσουμε τι προτάσει μα, τι προτάσει εκείνε που πιστεύουμε ότι ενδεχομένω να γίνουν αποδεκτέ από όλου και να υποστηριχθούν, να τις υποστηρίξετε. Είναι σαφέ ότι αν θέλουμε να ανταποκριθούμε στην πρόκληση αυτή, Χρειάζεται την ε, σαφή υποστήριξή σας. Χρειάζεται εποπτεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν μου επιτρέπετε πριν κλείσω, κυρία Πρόεδρε, δύο παρατηρήσεις για θέματα τα οποία δεν ε, έχουν να κάνουν με το βασικό ζήτημα, αλλά παρόλα αυτά θέλω να τα αναφέρω. Τα θέματα του κυρίου ε, Όλιβιε και ο Μαρτζέ σε ό,τι αφορά το, την πρόσφατη απόφαση του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου. Παρά το γεγονός ότι μελετάμε σε βάθος την ε, απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η πρόεδρος μίλησε ξεκάθαρα, νομίζω. Είπε με σαφήνεια ότι σε ό,τι αφορά την, ε, τον πρωτεύοντα ρόλο του Ευρωπαϊκού Δικαίου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι αρχές αυτές τις οποίες είμαστε ευτεθειμένοι να προασπιστούμε και με την διαδικασία επί παραβάση ενδεχομένως και προς την κυρία Γιούντσεβα να πω το εξή. Να σας διαβεβαιώσω ότι εργαζόμαστε για μια έκθεση για το κράτος δικαίου. Θα μελετήσουμε ενδελεχώς όλα τα περιστατικά και το πώς οι κυβερνήσεις ε, άσκησαν αυτές τις ιδιαίτερες εξουσίες που είχαν στην κρίση για να μπορέσουμε να επανέλθουμε το συντομότερο δυνατόν στο κανονικό δημοκρατικό σύστημα. Όλα αυτά λοιπόν θα τα λάβετε το αργότερο στο Σεπτέμβριο στα γραφεία σας. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι κύριε Πρόεδρε για τη συζήτηση αυτή, για τις ιδέες, την ενθάρρυνση που ένιωσα κατά τη διάρκεια της συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ Επίτροπε Σεύκοβιτς. Και τώρα η κυρία Μπρινιάτς από το Συμβούλιο. members. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριε και κύριοι, χαίρομαι πολύ που μπορώ να σας μιλήσω και πάλι αυτοπροσώπως. Σας ευχαριστώ για αυτή την πολύ χρήσιμη συζήτηση και θα μεταφέρω τις απόψεις σας στους συναδέλφους μου και του συναδέλφου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τους συνεργάτες μας. Είναι άνευ οι συνθήκες που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Όμως, γι' αυτό απαιτείται να δουλέψουμε σκληρότερα προς όφελος των πολιτών και των οικονομιών μας. Όπως σας είπε και ο πρόεδρος Μισελ, ο κοινό μας στόχος είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο να δημιουργήσουμε μια μακροπρόθεση πρόθεσμη απόκριση για τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19. Εδώ απαιτείται να υπάρξει ευρωπαϊκή στήριξη με τη βοήθειά σας, ε, πράγμα που φάνηκε ότι υπάρχει σκοπός να γίνει και τις προηγούμενες εβδομάδες. Ο πρόεδρος της Επιτροπ... Η πρόεδρος της Επιτροπής σας έδωσε τις αδρές γραμμές ενός ανανεωμένου πολιτής δημοσιονομικού πλαισίου και τις δημοσιονομικές μας προοπτικές. Μόλις δούμε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα τοποθετηθούμε. Προς στιγμή δεν γίνεται να σχολιάσουμε την ουσία. Ε, οι προτάσει θα πρέπει να αναλυθούν ε, στο απαραίτητο επίπεδο με προσοχή από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όπως απαιτείται για να δημορφώσουμε τη θέση μας επί του κειμένου το ερχόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο θα μπορεί να είναι ένα νέο λήθο για την ανάκαμψη στην ευρωπαϊκή οικονομία. Θα πρέπει να νοικοδομηθεί και να ξαναδημιουργηθεί η νέα αγορά για να λειτουργήσει σωστά και, μετά την περίοδο, και στην περίοδο μετά το COVID. Θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι υπάρχουν μαζικέ δημόσιε επενδύσει. Ιδίω στα πρώτα χρόνια των νέων δημοσιονομικών ε, προοπτικών η ε, ευρωπαϊκή οικονομία μετά την κρίση θα πρέπει να είναι ανθεκτική και περισσότερο αυτάρκη, ώστε η ανάκαμψη να είναι γρήγορη και αποτελεσματική. Θα πρέπει να υπάρχει συνοχή και σύγκληση καθώ και αλληλεγγύη. Αυτά θα είναι τα πρώτα στοιχεία. Θα πρέπει να υπάρχει διαρκή σταθερή συνεργασία μεταξύ των θεσμικών μα οργάνων και αυτό θα είναι ένα απόσπαστο στοιχείο όλη αυτή τη διαδικασία. Η Προεδρία δεσμεύεται να διατηρήσει τι καλέ σχέσει συνεργασία που έχουμε ήδη δημιουργήσει προκειμένου να αποκριθούμε στην όλη κρίση και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να αφουγκραστούμε τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Έχω σημειώσει λοιπόν την ε, σημασία της έκθεσης νομοθετικής, την έκθεση πρωτοβουλία νομοθετικής υφής που ετοιμάζεται καθώς και το ψήφισμα. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πώς τοποθετείται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο προσκήνιο αυτής της κρίσης. Θα πρέπει να υπάρχει καλή θεσμική συνεργασία. Αυτό θα είναι ουσιώδους σημασία για όλη την τομεακή μας δουλειά. Θα πρέπει να εργαστούμε από για να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει έγκαιρη έγκριση των τομεακών προγραμμάτων και θα ανυπομονούμε να συνεργαστούμε περαιτέρω και μαζί σα από αυτόν. Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, πραγματικά ανυπομονώ για την συνέχεια τη συνεργασία μεταξύ των δύο θεσμικών μα οργάνων για να δημιουργήσουμε ένα φιλόδοξο πεδίο επί του οποίου θα δραστεί το μελλοντικό πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και από όπου θα μπορέσουμε από κοινού να αντιμετωπίσουμε τι μελλοντικέ προκλήσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Υπουργού Μπινιάκη. Εδώ κλείνουμε την σύνοδο και η ψηφοφορία για το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο παραμένει ανοιχτή και την πέμπτη και την... θα λάβει την πέμπτη και την Παρασκευή. Διακόπτεται η σύνοδος. Il Presidente. Allora, questi li devono... Λοιπόν, επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. κύριος Κρίστιαν Βαζίλ Τέρες εγκατέλειψε την ομάδα S&D και πήγε στην ομάδα ECR από τις 13 Μαΐου 2020 αποτελέσματα του πρώτου γύρου ψηφοφοριών Ίντα εγκρίνεται Γιούρι εγκρίνεται. Τραν εγκρίνεται. Τραν εγκρίνεται. Τραν εγκρίνεται. Ευρωπαϊκή Ένωση Μαυροβούνιο εγκρίνεται. Σερβία εγκρίνεται. Ευρωπαϊκή Ένωση Ινδία εγκρίνεται. Ευρωπαϊκή Ένωση Ουκρανία εγκρίνεται. Ευρωπαϊκή Ένωση Λευκορωσία εγκρίνεται. Εγκρίνεται. Σύμβαση ΙΚΑΤ εγκρίνεται. Μαυριτανία εγκρίνεται. Πι δελτα Π. εγκρίνεται. Καμποτάζ Γερμανία Ελβετία εγκρίνεται. Καμποτάζ Ιταλία Ελβετία εγκρίνεται. ανταλλαγή δεδομένων με Ηνωμένο Βασίλειο απορρίπτεται. Αντιρρήσεις για τη σόγια τροπολογία ένα μέρος πρώτο εγκρίνεται, μέρος δεύτερο εγκρίνεται. Απόφαση για την απαλλαγή FCH εγκρίνεται, Clean Sky εγκρίνεται, BBI εγκρίνεται, ΕΙΟΠΑ εγκρίνεται. Η CSL e εγκρίνεται. Η μη 2 εγκρίνεται. Shift to rail εγκρίνεται. ΕΑ e εγκρίνεται, ERA εγκρίνεται, EMSA εγκρίνεται, GSA εγκρίνεται, EMC DDA εγκρίνεται, ΕΑΖΑ e εγκρίνεται. ΕΑΖΟ εγκρίνεται. Κοινοβούλιο εγκρίνεται. Δικαστήριο εγκρίνεται. Συνήγορος πολίτη εγκρίνεται. Η DPS εγκρίνεται. Η ECA εγκρίνεται. ΣΕΔΕΤΕ εγκρίνεται. Συμβούλιο εγκρίνεται. Ενίζα εγκρίνεται. Σεντεφόπ εγκρίνεται. Η FCA εγκρίνεται. Η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης εγκρίνεται. Σέζαρ εγκρίνεται. Η ETF εγκρίνεται. Η Eurojust εγκρίνεται. Η ITER εγκρίνεται. Μπέρεκ εγκρίνεται. Eurofound εγκρίνεται. Acer εγκρίνεται. Η Γιουλίζα εγκρίνεται. Η IT εγκρίνεται. Η SA e εγκρίνεται. Η EDFs εγκρίνεται. Η IGE εγκρίνεται. ΕΣΜΑ εγκρίνεται. Τραπεζική αρχή εγκρίνεται. Αστυνομική Ακαδημία εγκρίνεται. Όσα εγκρίνεται. Η CHA εγκρίνεται. Η CDC εγκρίνεται. ΕΦΣΑ εγκρίνεται. Κομισιόν εγκρίνεται. FRA εγκρίνεται. COR εγκρίνεται. Frontex εγκρίνεται. Europol εγκρίνεται. ΕΜΕ εγκρίνεται και SC εγκρίνεται. Αυτές είναι οι ψηφοφορίες του απογεύματος. Περνάμε τώρα στο δεύτερο γύρο ψηφοφοριών. περνάμε στο πρώτο μπλοκ τροπολογιών για τα ψηφίσματα απαλλαγή και στην τελική ψηφοφορία για τις ε, αντιρρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 112 για την τροποποιημένη σόγια. Οι ψηφοφορίες θα γίνουν με τον ίδιο τρόπο που έγιναν και στον πρώτο γύρο από τις 8 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 9 και 4. Ψηφοφορία ανοίξει σε λίγο. Θα έχετε χρόνο για να ψηφίσετε. Τα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου θα ανακοινωθούν αύριο με την έναρξη της συνεδρίασης και ώρα 9. Οπότε, Τώρα διακόπτεται η συνεδρίαση η οποία θα επαναληφθεί αύριο 5η 14 του μηνός ώρα 9 η πρωινή. Ζητήσα τον λόγο. Όχι. σε διάταξη θα δημοσιευτεί στην σελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αγαπητοί συνάδελφοι, διακόπτεται η συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία. Καλή ψηφοφορία και τα λέμε αύριο.